Good afternoon, colleagues. Um, we can begin this afternoon's agenda. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, συνάδελφοι, με το σημείο 25, που είναι η καταπολέμηση της ε, διαφθοράς και συνέχεια στο ψήφισμα της Ειδικής Επιτροπής ΚΡΙΜ. Η Λόρα Φεράρα είναι η συγγήτρια στην τελευταία θητεία. Δημιουργήθηκε μια ιδιαίτερη ειδική επιτροπή με σκοπό την έρευνα της ε, διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος και των ε, τόσο. Προέκυψε λοιπόν ε, το σχετικό ψήφισμα του 2013 και τώρα λοιπόν θα κοιτάξουμε κατά πόσο έχουν εφαρμοστεί οι συστάσεις ε, και σκοπός είναι να βελτιωθούν τα ένομα μέσα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Φεράρα για να μας ε, παρουσιάσει το εγγραφό της. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα μάλλον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και οδησιογητές για αυτές τις υποδείξεις όσα μου είπαν ε, τις προηγούμενες μας συναντήσεις ε, στη συνάντηση με τους και οδησιογητές ακριβώς. Έχουμε ένα working document ε, σήμερα, αυτό θα εξετάσουμε και σαν στόχο το έγγραφο αυτό έχει θέση να παρουσιάσει ποιες είναι οι προσπάθειες, οι στόχοι ακριβώς ε, που έχουμε θέσει και η αφετηρία ήταν ε, η έκθεση του 2011 για το οργανωμένο έγκλημα και για το ψήφισμα του 2013 που εγκρίθηκε από την Ειδική Επιτροπή ε, περί εγκλήματος βέβαια δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες και το ίδιο χρονικό διάστημα με την ειδική αυτή επιτροπή για το έγκλημα και χρειάστηκε να περιορίσουμε κάπως εργασίες μας χρονικά πάνω σε ορισμένους ειδικούς στόχους που θα πρέπει να επιδιώκουμε και για να αποφύγουμε τα φτάσουμε και με μια έκθεση ε, πλατιά μεν αλλά που θα είχε πάρα πολλά θέματα και θα χανόμαστε ανάμεσα. Να δούμε λοιπόν τι συμμεριζόμαστε μαζί σας για αυτή την ενδιάμεση έκθεση τους στόχους και προς ποια κατεύθυνση θα μπορούσαν να πάνε αυτές οι εργασίες και να ακούσω περαιτέρω σχόλια και υποδείξεις από σας. Αφετηρία λοιπόν, το πρώτο πρόβλημα για να δούμε ποιες είναι οι διάφορες ενέργειες που θα πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της διαφθοράς και του εγκλήματος, θα πρέπει να δούμε το πρόβλημα ακριβώ λόγω της έλλειψης συνείδησης του περίπλοκου του προβλήματος αυτού και η μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς αποτελεί ένα πρόβλημα και ρυθμιστικό βέβαια, αλλά ταυτόχρονα ένα πρόβλημα πολιτιστικό. Ένα πρόβλημα το πώς αντιλαμβανόμαστε όλοι οι πολίτες το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει κοινή συνειδητοποίηση για το πόσο περίπλοκο είναι αυτό και το τι επικίνδυνο είναι λόγω της των εκφοβιστικών ενεργειών ε, στον τομέα. Άρα λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει συνειδητοποίηση κατάλληλη, αντίληψη κατάλληλη για το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το φαινόμενο το εκφοβιστικό από τις εγκληματικές οργανώσεις. Αυτές έχουν εξελιχθεί, έχουν αναπτυχθεί και έχουν αλλάξει και την εσωτερική τους οργάνωση ώστε να μοιάζει σχεδόν με μια πολυεθνική επιχείρηση και για να συγκεντρώσουν οι προσπάθειές τους εκεί που θα κερδίσουν περισσότερο ανάλογα με τα κενά, τα νομοθετικά, τα ρυθμιστικά ανάμεσα στα κράτη-μέλη, τις διαφορές και τις διάφορες προτεραιότητες που έχει το κάθε κράτος μέλος για να μπορέσει να ενεργήσει καλύτερα, να δραστηριοποιείται εκεί και να κατευθύνει τις ενεργειές του. Αυτό το δίκτυο. Ε, βέβαια θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει ένα κοινό, μια κοινή βάση νομοθετική λόγω της ειδική αυτής, ε, του ειδικού χαρακτήρα των εγκληματικών οργανώσεων ε, και γι' αυτό ακριβώς ενισχύθηκαν οι δυνατότητές τους ε, γιατί μπήκαν ακόμα και σε υγιείς οικονομίες κρατών μελών. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι από παρόμοια εγκλήματα το προϊόν μπαίνει ξανά ξεπλένεται στην ίδια την οικονομία του κράτους γιατί κυρίως οι μαφιόζικες αυτές οργανώσεις ε, έχουν ε, μια συνεργασία και σε εθνικό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο. Ξέρουμε από τις ενέργειές τους ε, από αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις ότι απλώνονται λοιπόν και σε ευρωπαϊκό γενικότερο επίπεδο και όχι μόνο εθνικό. Και γι' αυτό ακριβώς θα δούμε και αυτόν τον μηχανισμό και τη σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά φαινόμενα αντί να τα πάρουμε ξεχωριστά. Να δούμε, στο έγγραφο αυτοεργασία, αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια κοινή ανάλυση αυτών των δύο πτυχών για να δούμε πώς αλληλοσυμπληρώνονται αμοιβαία και τη σχέση ανάμεσα αυτά τα δύο η διαφθορά πολλές φορές είναι ένα πρώτο μέσο που χρησιμοποιείται από το οργανωμένο έγκλημα για να μπει μέσα να διεισδύσει στην πολιτική, στο κοινωνικό σύστημα, στην οικονομία ενός κράτους μέλος και να επηρεάσει τις διάφορες αποφάσεις και που, πάνε, που πάει το δημόσιο χρήμα, που πάνε οι επενδύσεις και να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και τους κανόνες της αγοράς και δεν υπάρχει πάνω σε αυτό το θέμα μια αποτελεσματική νομοθετική βάση. Και γι' αυτό ακριβώς οι διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε, να καταστήλουμε το φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε τη μάχη μας πάνω σε δύο, ε, μπροστά σε δύο μέτωπα. Και στην ε, καταπολέμηση αλλά και στην πρόληψη. Χρειάζονται και τα δύο. Χρειάζεται προληπτικά να προλάβουμε με ένα έλεγχο σταθερό και με παρεμβάσεις από τη στιγμή που υπάρχει συστηματική διαφθορά και μια περισσότερη διαφάνεια ε, στο τι κάνει το δημόσιο και να μπορέσει κανείς να αντιληφθεί τι σημαίνει ακριβώς νομιμότητα σε ένα κράτος και να υπάρξει μια κατάλληλη σχέση ε, ανάμεσα στον κανόνα και στην εξαίρεση και όχι όπως έχει τώρα αυτή η σχέση γιατί η διαφθορά θεωρείται πια κάτι το κανονικό και σχεδόν είναι νόμιμο δεν εκπλήσει πια κανένα παρόμοιο φαινόμενο διαφθοράς του οργανωμένου εγκλήματος σε ευρωπαϊκή κλίμακα ενώ αντίθετα θα έπρεπε να ντραπούμε πραγματικά για αυτές τις ενέργειες του οργανωμένου εγκλήματος που διαβρούν την οικονομία αλλά και τα θεμελίδη δικαιώματα των ε, Ευρωπαίων πολιτών για ένα υγιή κανόνα ανάμεσα στον κανόνα ακριβώς ε, και στην εξαίρεση τι σημαίνει αυτή η παρέκκληση με το οργανωμένο έγκλημα τη διαφθορά και στο έγγραφο εργασίας εξετάσαμε αυτά τα γενικότερα στοιχεία και τώρα προχωράμε σε ειδικούς τομείς παρέμβασης. Πώς τους επιλέξαμε ανάλογα με τις προτεραιότητες αυτής της ε, στιγμής της ιστορικής μπορούμε να πούμε χρονικής με τρεις τομείς παρέμβασης το οργανωμένο εγκλημά που έχει σχέση με, τις, ε, με τους πρόσφυγες, με το περιβάλλον και το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά που έχει να κάνει με την ε, διάθεση των χρημάτων που κερδίζουν. Το πρώτο θέμα θα δούμε για το εμπόριο ε, ακριβώς ε, ατόμων, ανθρώπων ε, και τι, πώς επεμβαίνουν στα κέντρα υποδοχής όσων ζητούν ε, άσυλο, για την ε, πώληση οργάνων, για τη σκλαβιά μπορούμε να πούμε και είναι ένας πολύπλατης τομέας σίγουρα και ακριβώς εκεί που έχει διεισδύσει το οργανωμένο έγκλημα και η διαφθορά ε, τα βλέπουμε καθαρά τι εύρος έχουν αυτές οι ενέργειες και έχουν δημιουργήσει πραγματικά ένα κύκλο εργασιών σαν κανονική επιχείρηση. Δεύτερο τώρα με το περιβάλλον ε, προσέχουμε ιδιαίτερα το θέμα της οικολογικής μαφίας όπως την αποκαλούμε για το περιβάλλον που πλήττουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών περισσότερο από την οικονομία είναι το δικαίωμα στην υγεία, στη ζωή την ίδια και γνωρίζουμε τη διείσδυση του οργανωμένου εγκλήματος στην όλη διαχείριση ας πούμε των αποβλήτων ε, και τοξικών αποβλήτων. Και γι' αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την καταστολή και την πρόληψη αυτών των εγκλημάτων που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, γιατί τα σημερινά μέτρα είναι και ανεπαρκή. Ταυτόχρονα όμως επηρεάζουν και τα οικονομικά των πολιτών. Έχουμε αυτό τον ε, άρρωστο μηχανισμό πραγματικά με αυτές τις παραβιάσεις ε, και εδώ ε, η προστασία του πολίτη είναι μια διαδικασία προσφυγή επί παραλήψη ε, απέναντι σε ένα κράτος μέλος που δεν σέβεται το περιβάλλον. Αλλά αυτή η προσφυγή για αυτή την παράβαση δεν είναι ότι αποκαθίσταται η νομιμότητα. Απλά και μόνο ένα πρόστιμο που θα πρέπει να πληρώσει το κράτος, η χώρα, επειδή δεν εφάρμοσε όπως έπρεπε την κοινοτική νομοθεσία. Και γι' αυτό ακριβώς είναι διπλή ζημιά για τον πολίτη και για τα θεμελιώδη δικαιώματά του αλλά και οικονομική ζημιά. Τρίτος τομέας παρέμβασης ε, που πάει το δημόσιο χρήμα με τις ε, αναθέσεις και τους διαγωνισμούς κλπ. Εκεί πολλές φορές ε, πληρώνουν, λαδώνουν τους δημόσιους λειτουργούς. Εδώ λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε και το ότι ασκούν έτσι ένα έλεγχο και εκφοβίζουν τον κόσμο για να μπορέσουν να κάνουν τις δουλειές τους. Εδώ λοιπόν πολλά πράγματα που είπαμε δεν έχουν, γίνει, δεν έχουν εισακουστεί μέχρι τώρα. Χρειάζεται μια ρύθμιση με ανιχνευσιμότητα το πού πάνε αυτά τα χρήματα, πού πάνε οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις καταλήγοντας για τις συστάσεις τις οποίες θα μπορούσαμε να απευθύνουμε με την έκθεσή μας αυτή νομίζω ότι σίγουρα θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε την προστασία των whistleblowers και των ε, συνεργατών και της δικαιοσύνης στο σύνολό της ε, και σύστημα προστασίας, ε, όλα αυτά τα πράγματα που έχουν βέβαια διαφορετικά το ένα από το άλλο. Να έχει ελάχιστες, ελάχιστα στάνταρτ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως και ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό προστασίας και ακόμα πώς θα χρησιμοποιηθούν κοινωνικά τα όσα έχουν κατασχεθεί γιατί αυτά, η χρηματική ανάθεση, η εισφορά κλπ. έχει μεγάλη σημασία για μια σωστή χρησιμοποίηση για κοινωνικούς σκοπούς των όσων έχουμε κατασχέσει από το οργανωμένο έγκλημα με μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτοκών, ανάμεσα στα κράτη-μέλη, με ένα κατάλληλο δίκτυο, με εθνικούς οργανισμούς για τη διάθεση αυτών των κατασχεθέτων ποσών ή υλικών και ακόμη ε, να, μπορέσουν, ε, να μπορέσουμε να έχουμε μια οικονομία κλίμακος με κατάλληλο προϊόντα που θα προκύψουν από αυτά τα κατασκευαστικά ποσά υλικά. Και εδώ αυτό όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη βάση πάνω στη οποία θα ακουμπήσουμε για την ε, τελική έκθεση. Από δική σας πλευράς τώρα, ολοκληρώντας, περιμένω υποδείξεις, σχόλια κλπ, ώστε να μπορέσω να εμπλουτίσω το όλο περιεχόμενο της έκθεσής μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Λόρα. Είναι εδώ ορισμένοι σκιώδεις. Θα τους δώσουμε το λόγο. Νάταλη Γκρισμπέρκ, σκιώδης από Άλντε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τη Λόρα Φεράρα για την παρουσίαση που μας έκανε. Ως ασκιώδης για την ομάδα Άλντε θα ήθελα να κάνω ορισμένες επισημάνσεις. Αρχικά είναι ιδιαίτερα σκόπιμο και επίκαιρο αυτό το έγγραφο που μας έδωσε ε, η Λάουρα. Το λάβαμε στη γαλλική μετάφραση μόλις χθες, αλλά ήδη είχα παρακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία η οποία συμπεριέλαβε σε μεγάλο βαθμό και τους επιμέρους ασκηώδης και αποτελεί μια καλή αφετηρία ε, για τη συνέχεια. Τώρα, επί του τύπου, σκοπός ε, ο σκοπός της έκθεσης είναι πολύ σημαντικός και ευχαριστώ τη Λάουρα που έδειξε αυτή την βούληση αλλά και κατέβαλε και την ε, προσπάθεια να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας, να επικεντρωθούμε λοιπόν σε κύρια σημεία, σε βασικές προτεραιότητες για αυτό που είχε θετηθεί το 2013 της Επιτροπής ε, ΚΡΙΜ ε, μετά την υπόθεση για Κολίνο. Και τότε είχε γίνει μια πολύ καλή ε, έκθεση. Ιδιαίτερα εμπιστευτομένη. Και από τότε μπορούμε να διαρωτηθούμε κατά πόσο ε, έχει δοθεί συνέχεια σε αυτή την πολύ ουσιαστική προσπάθεια, γιατί τα περισσότερα στοιχεία έμειναν χωρίς συνέχεια. Πρέπει λοιπόν να ιεραρχήσουμε ορισμένους τομείς ως προτεραιότητες για να είμαστε σίγουροι ότι θα καταφέρουμε να διασφαλίσουμε και θα αναγκάσουμε και τα κράτη-μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Είμαι υπέρ της στρατηγικής της Λάουρα, δηλαδή να επικεντρωθούμε σε λίγα και καλά στοιχεία, να μην φτιάξουμε αυτό το χριστουγεννιάτικο δέντρο, όπως λένε, το οποίο είναι με μένα ευχάριστο, αλλά στην πράξη δεν αποφέρει καρπούς. Εν συντομία θα ήθελα να ευχαριστήσω και τη Λάουρα επειδή έδωσε έμφαση στην αναγκαιότητα ευθυγράμμισης των επιμέρους εθνικών νομοθεσιών, ακόμα και αν αυτό είναι μεγάλη προσπάθεια και είναι και μακρύς ο δρόμος, όπως το ξέρουμε όλοι. Σε ό,τι φορά και την ε, μεταφορά των νομοθετικών έργων στην εθνική νομοθεσία, πολλές φορές υπάρχουν ε, ε, δυσκολίες και καθυστερήσεις. Χαιρετίζω και την έμφαση που δόθηκε και στην ομάδα μου γενικά αυτό μας ικανοποιεί, στους τρεις ε, συγκεκριμένους τομείς παρέμβασης που βλέπουμε στο έγγραφο, για σύνδεση μεταξύ εγκληματικότητας και μετανάστευσης, εγκληματικότητας και περιβάλλοντος και η σύνδεση που πρέπει να γίνει μεταξύ διαφθοράς και χρήσης αξιοποίησης δημοσίων ε, πόρων. Ήδη σε αυτό το έγγραφο εργασίας ε, υπήρξε αναφορά στην ε, προστασία που πρέπει να δώσουμε στους whistleblowers, σε όσους δηλαδή επισημαίνουν τα κακό κείμενα. Υπάρχει και αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ε, μετα... συνομπροστασία μέσα στο έγγραφο και αυτό είναι μια νέα ιδέα. Θα ήθελα να προσθέσω μόνο, βεβαίως αυτό θα το εξετάσουμε και στη συνέχεια κατά την εκπόνηση της έκθεσης. Θα ήταν σημαντικό λοιπόν να επικεντρωθούμε στην ε, φορολογία, στο ζήτημα των ε, φορολογικών παραδείσων και στην ε, φοροδιαφυγή. Βεβαίω και η Λάουρα θα μπορούσε όλα αυτά να τα συμπεριλάβει στην έκθεσή της. Γιατί το οργανωμένο έγκλημα, όπως λέμε πάντα, δεν έχει σύνορα. Γι' αυτό και η ανταπόκρισή μας θα πρέπει και αυτή να μην έχει σύνορα. Πρέπει λοιπόν να δοθεί ευρωπαϊκή απάντηση για να διαμορφώσουμε και να ενδυναμώσουμε τα ευρωπαϊκά μέσα, είτε αυτά είναι διασυνοριακά, όπου αυτό είναι απαραίτητο. Θεωρώ ότι είναι. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς ε, τα στοιχεία, αλλά είναι τόσο αστρονομικά που θα τα αναφέρω έτσι κι για να έχετε μια ιδέα της τάξης μεγέθους. 110 δις ευρώ κέρδη έχουν οι εγκληματικές οργανώσεις στην Ευρώπη. Διαβάζουμε. Πρέπει λοιπόν η απάντηση να είναι κοινή και ευρωπαϊκή. Και κλείνοντας, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, παρότι είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε και να ελοποιήσουμε αυτή την ιδέα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Εδώ και 30 χρόνια το συζητούμε και δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Γιατί υπάρχουν ορισμένες αντιστάσεις από κάποια κρατημέλη και βεβαίως ε, έχουμε αυτή την ατέρμονη συζήτηση για την εισαγγελία αλλά και σήμερα το πρωί για την τρομοκρατία όπου δεν προοδεύουμε αρκετά και συμπεραίνουμε ότι εάν δεν προχωρήσουμε αρκετά ακόμα και οι πιο φιλοευρωπαϊστές μεταξύ μας θα γυρίσουν οριστικά την πλάτη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Οι σκιώδεις λοιπόν τώρα και άλλοι συναδελφοί έχουν ζητήσει το λόγο. Η κυρία Γιώτοβα πρώτη. Θα ήθελα να συγχαρώ την Λάουρα για την καλή δουλειά που έκανε και για το έγγραφο εργασία που μας παρουσίασε. Είναι αναλυτικότατο πριν από κάποιες ημέρες έγινε μια κοινή συζήτηση των σκιωδών με την εισηγήτρια και αποφασίσαμε καταρχάς να υπάρξει μια εισαγωγή με τις προτεραιότητες και στις συστάσεις ότι θα θέλαμε να αναφέρουμε τα όσα προτείνουμε. Και χαίρομαι λοιπόν που έγινε αυτό γιατί συμμετείχα και στην Επιτροπή ΚΡΙΜ και κάναμε πολλά στην ε, έκθεση Ακούλενο. Και πραγματικά εύχομαι αυτή η κοινή έκθεση να έχει πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Όχι επειδή η αρχική έκθεση ήταν κακής ποιότητας, ήταν πολύ αναλυτική, αλλά δυστυχώς τα αποτελέσματα που έχει πετύχει μέχρι σήμερα είναι πολύ μέτρια. Η έκθεση λοιπόν αυτή, η οποία έχει να κάνει με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος περιλαμβάνει 120 συγκεκριμένες συστάσεις. Λίγες εκ των οποίων έχουν εφαρμοστεί ως τώρα. Ελπίζω λοιπόν η έκθεση αυτή να μπει στο επίκεντρο της προσοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν θα λαμβάνουν νομοθετικές πρωτοβουλίες και θα καταθέτουν προτάσεις. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν η έκθεση που προετοιμάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαφθορά στα κράτη-μέλη να ξεπεράσει την ε, έκθεση διαπίστωσης απλών γεγονότων και να εστιαστεί στα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει και αυτή η επικέντρωση στην έκθεση. Ελπίσεις να πω ότι πιστεύω ότι στην έκθεση αυτή μπορούμε να προσθέσουμε πολλά συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την εναρμόνιση, τη σύγκρουση συμφερόντων, τον παρανόμος ε, αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, βλέπετε. Και να μπορέσουμε να λιάνουμε αυτές τις διαφορές. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να περιλαμβάνουμε στο κείμενο το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία. Έχει μπλοκάρει στο Συμβούλιο αυτό το θέμα και φαίνεται ότι έχει καταλήξει σε αδιέξοδο επί του παρόντος τουλάχιστον. Πιστεύουμε λοιπόν ότι Όλοι έχουν τα συγκεκριμένα. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αναλάβει τα συγκεκριμένα του καθήκοντα γιατί πραγματικά έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι το θέμα των φορολογικών παραδείσων. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια ειδική επιτροπή και μια έκθεση της ειδική επιτροπής αυτής έχει διεγκρίθει. Ενδεχομένω λοιπόν να υπάρξει και μια δεύτερη επιτροπή τέτοιου είδους. Το θέμα όμως αυτό είναι σημαντικό και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παραλυφθεί από την έκθεση αυτή. Τέλος, ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχουμε ξεχάσει φαίνεται επί του παρόντος είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Ανθρωπιστική Βοήθεια σε τρίτες χώρες και οι πρακτικές διαφθοράς στις χώρες αυτές. Ε. Όλο και πιο πολλά στοιχεία λοιπόν λαμβάνουμε για το θέμα αυτό. Και εντωμεταξύ θα συνεχίσουμε το έργο μας για την έκθεση αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και ελπίζω και πιστεύω ότι χάρη στις κοινέ μας προσπάθειες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει τις προσπάθειές μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Φερ για όλα αυτά που μας είπε και ε, με τα στοιχεία των σκιωδών εισηγητών. Θα έπρεπε ίσως να αναφερθεί περισσότερο πώς εμείς χάσαμε τη μάχη κατά της διαφθοράς στην Ευρώπη και να χρησιμοποιήσουμε και μερικά παραδείγματα για να δείξουμε ότι από τις πολυεθνικές η διαφθορά άλλαξε την όλη φύση του εγκλήματος γιατί είναι μύθος ότι, ότι ε, πολεμήσαμε και κερδίσαμε δεν ξέρω, ξέρετε την υπόθεση Siemens ε, με πολλές περιπτώσεις διαφθοράς τις οποίες κατηγορήθηκε, πιάστηκε με αυτό φόρο και έχουμε και ένα συναγερμό κινέζικο τι μας λένε οι Siemens ε, ε, σε διάμεσους Κινέζους ε, πουλούσε αλλά πολύ κάτω τη συνήθους τιμής. Καταλαβαίνετε ότι όλες αυτές οι συναλλαγές ξεφεύγουν από την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη γιατί τίποτα δεν γίνεται εδώ κοντά. Είναι καθαρά τα βιβλία τους πρέπει να δείξουμε περισσότερο αυτή την ε, μάχη που δίνουμε που δυστυχώς όμως με ε, μηδαμινά αποτελέσματα και το ρόλο επίσης που παίζουν οι πολυεθνικές εταιρείες θα μπορούσε να προσθέσει κανείς ε, ότι ακριβώς δεν μπορούμε να πετύχουμε και την ειρήνη όπως είδαμε στο Αφγανιστάν λόγω της διαφθοράς ε, γιατί πήγε αλλού στο Ντουμπάι ένα μεγάλο μέρο ανθρωπιστικής βοήθειας είναι η μαύρη τρύπα που απορροφάει τα πάντα και, και δεν ανταποκρίνεται στο αίτημα στο διεθνές περί συνεργασίας για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε αυτά τα χαμένα χρήματα και θα πρέπει να μην πιστεύουμε πια ότι τα κείμενα τα νομοθετικά θα αλλάξουν τον κόσμο. Έχουμε πολλές ε, εκθέσεις, πολλές συμβάσεις. Είναι σημαντικές βέβαια αυτές, αλλά ακόμα και του ΟΗΕ για τη διαφθορά. Αυτά όλα δεν παρεμπόδισαν τις πολυεθνικές εταιρείε να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες μας ε, στην εφαρμογή. Χρειάζονται μέσα όμως. Εκεί δυστυχώς Ιταλία διαθέτει κατά της κοινωνικής μαφίας μια επιτροπή. Εδώ και 50 χρόνια την έχουν, ε, αλλά δεν έχει καταφέρει τίποτα, τίποτα να αλλάξει πάνω σε θέματα μαφίας στην Ιταλία. Στη ώρα θα ήθελα να προτείνω να συμπεριλάβει και ένα πίνακα με τα κράτη-μέλη τα πόσα χρήματα δαπανούν στη δικαιοσύνη σχέση με το ΑΕΠ τους βέβαια και να δείξουμε ότι απλά και μόνο λόγια μεγάλα ακούγονται και όχι χρήματα τα οποία αφιερώνουμε εκεί για αυτή τη μάχη. Όπως έγινε μια λάθος ερμηνεία από την σκιώδη συγκήτρια προηγουμένως σε αυτό που έγραψε η Φερέρα για τις πρόσφυγες δεν λέει ότι ε, φταίει οι πρόσφυγες για τη διαφθορά αλλά λέει ότι οι πρόσφυγες ακριβώς είναι θύματα της μαφίας που διαχειρίζεται τα κέντρα υποδοχής έτσι αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε στο τι τίτλο βάζουμε γιατί ο κόσμος ίσως δεν καταλαβαίνει από τον τίτλο τι λέμε και παρακάτω κάτι επίσης που είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε για αυτό το συναγερμό, ποτέ σημαίνει και την προστασία. Το Συμβούλιο καθαρά είπε, όπως και η Επιτροπή επίσης, ότι δεν επιθυμούν ελάχιστους κανόνες ε, προστασίας, πρέπει όμως να το υπενθυμίσουμε, να το υπενθυμίσουμε γιατί η διαφθορά δεν μπορούμε χωρίς ε, παρόμοια μέσα να την καταπολεμηθεί. Αυτό η συγγήτρια το τόνισε σωστά και επίσης ένα πρόβλημα που δεν το είδα αλλού. Όταν ακριβώς ε, προβαίνει σε κατάσχεση ε, από εγκληματικέ οργανώσεις ε, ας πούμε κόπεδα, σπίτια κλπ. κίνητα αλλά κανείς δεν τα αγοράζει μετά γιατί φοβούνται εφόσον ξέρουν ότι ανήκει στη μαφία καταλαβαίνετε αυτό τα αγοράζει τι κίνδυνο διατρέχει μετά και επίσης κάτι άλλο. Όταν ακριβώς ε, παγώνουμε λογαριασμούς και λοιπά αυτό το να διατηρηθεί ε, κοστίζει πολλά το να κατασχέσει κανείς ε, να το παγώσει μάλλον να το κρατήσει έτσι και ένα αεροπλάνο που μετέφερε ναρκωτικά κοστίζει χρήματα είτε ένα πλοίο κοστίζει χρήματα η συντηρησή του θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε τα πράγματα με κατάλληλα κείμενα και ρυθμίσεις πώς θα μπορούσαν αυτά τα αγαθά να πολλούνται. Γιατί στην Ιταλία, στην Γαλλία κλπ. ξέρουμε ότι η διαδικασία πολλές φορές διαρκεί 10 ολόκληρα χρόνια και το να κρατάει κανείς τα υποστεγά του για 10 χρόνια αεροπλάνο ε, είναι κάπως ανώφελο. Γι' αυτό λοιπόν να υπάρξει αυτή η δυνατότητα και για επιστροφή χρημάτων επίσης ε, αν ε, βέβαια τελικά δεν καταδικαστεί ο κατηγορούμενος. Αλλά καλό επίσης είναι ότι τονίζει την ε, τις εγκληματικές ενέργειες που κοστίζονται με το περιβάλλον. Και αυτό το παράδοξο ότι για τα απόβλητα με καταδικάζονται κράτη και ότι τελικά οι πολίτες στην Νάπολη της Ιταλίας πληρούν δύο φορές πιο ακριβά τα απόβλητά τους και εκεί η μαφία είναι ανακατεμένη. Αλλά τι κάνει, είναι δια μετακομιστής ε, δηλαδή ας πούμε τα απόβλητα από φαρμακευτικές ε, εταιρείες και εργοστάσια. Και άρα λοιπόν ε, δεν είναι μόνο τις μαφίες ευθύνη, είναι και των όσων παράγουν αυτά τα απόβλητα εδώ πέρα στην, στις φαρμακοβιομηχανίες η επιπτώση στην υγιεινή. Καταλαβαίνετε όποιο ζει εκεί κοντά σε αυτά τα βουνά αποβλήτων ασφαλώς η θνησιμότητα θα είναι πιο συχνή, συχνότερη και σε χαμηλότερη ηλικία ακριβώ από ότι ε, αλλού. Αυτό. Θα ήθελα να συγχαρώ στην εισηγήτρια, να συγχαρώ την εισηγήτρια την εργασία της και εύχομαι να αποτελεί κάτι το κενό τόπο από τη στιγμή που θα θίγει την ευθύνη των ότι δεν υπάρχει διάθεση και μέσα οικονομικά για την καταπολέμηση αυτών από πλευρά κρατών. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ζολή ήταν σκιώδη ε, από πλευράς Πρασίνων και η κυρία Γιώτοβα από πλευράς Σοσιαλδημοκρατών. Κύριο Μέλο, επόμενο ομιλητή σκιώδη από πλευράς ΕΛΚ. Συνάδελφοι, προτιμώ, μάλλον προσπαθώ να μείνουμε στο χρονοδιάγραμμα σήμερα το απόγευμα σε σχέση, αντίθεση με αυτά που συνέβησαν το πρωί. Αν μπορείτε λοιπόν ε, να τηρείτε το όριο των τριών λεπτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσθέσω να είμαι σύντομο. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση. Γιατί η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι προτεραιότητα σε όλο τον κόσμο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Βεβαίω ε, η διαφορά δεν αφορά όλα τα κρατημέλη με τον ίδιο τρόπο. Αυτό το είπε η κυρία Φεράρα. Τώρα, υπάρχουν ε, σημεία κοινά, αλλά και ιδιαιτερότητες. Σε μια έκθεση δεν γίνεται μόνο να φέρουμε την Ιταλική πραγματικότητα, ούτε να αξιοποιήσουμε ως πολιτικό εργαλείο αυτή την έκθεση ε, αναφερόμενη στις ιδιαιτερότητες ε, της Ιταλίας και μόνο. Πρέπει να φέρουμε την έκθεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να μιλήσουμε για τα προβλήματα που ε, απαντούν σε άλλες χώρες της Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την πολιτική λιτότητα, για παράδειγμα, είναι ένα σημαντικό θέμα. Πράγματι, είναι κοινό παρονομαστή η καταπολέμηση τη διαφθορά. Όμως, εάν προσπαθήσουμε να πολιτικοποιήσουμε την ε, πάλι κατά της διαφθοράς, τότε κάποιοι από εμά ε, δεν θα αξιοποιήσουμε αυτό το μέσο. Ξέρετε ότι είμαι Πορτογάλος, ε, στη χώρα μου υπήρχε πρόγραμμα λιτότητας το 2011 και μετά. Η Τρόικα έφυγε από την Πορτογαλία τον Μάιο του 2014 και όλοι συμφωνούμε σε ό,τι αφορά τη σοβαρότητα της διαφθοράς σε όλες τις χώρες. Όμως, εάν για παράδειγμα θέλουμε να μιλήσουμε για πολιτικές λιτότητας όταν εξετάζουμε τη, τα θέματα διαφθοράς, τότε ξεφεύγουμε από το θέμα. Και γι' αυτό ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να δίνουμε πολιτικό περιεχόμενο και μόνο σε μία έκθεση, γιατί ο κίνδυνος είναι ε, να απομακρυνθούμε από το θέμα της έκθεσης. Εάν τώρα για κάποιες πολιτικές ομάδες αυτή η πολιτική λιτότητα ε, ήταν κάτι αναπόφευκτο που αποτέλεσε απόρρια της κατάστασης στις εμπλεκόμενες χώρες που δεν μπορούσαν να λάβουν άλλη χρηματοδότηση για παράδειγμα, τότε για άλλους ε, η λιτότητα μπορεί να ήταν η ενσάρκωση του κακού και να αποτελεί πρόσχημα για οτιδήποτε. Έχουμε λοιπόν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να πολιτικοποιούνται και υπάρχουν και άλλα στοιχεία νομικού χαρακτήρα που υπάρχουν σε ορισμένες χώρες και όχι σε άλλες. Η πραγματικότητα όμως ξέρουμε ποια είναι. Αλλά αυτό που αναφέρετε αφορά μία χώρα. Είναι υπερβολικό να προσπαθήσετε αυτό να το γενικεύσετε για όλες τις χώρες. Μετά βεβαίω υπάρχουν και ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά και μας ενδιαφέρουν όλους. Όμως είναι δύσκολο να εξετάσουμε αυτή την προβληματική δεδομένων ε, των ειδικών συμφερόντων των πολιτικών ομάδων. Κάποια στοιχεία μπορεί να είναι πολύ σημαντικά για να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Όμως ε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει και σύγκρουση συμφερόντων. Για παράδειγμα, στα κρατικά μυστικά. Υπάρχουν λοιπόν και αντιεπιχειρήματα ως προς όλα αυτά. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάζουμε και να τα αντιπαραβάλλουμε στο ζήτημα της ε, προστασίας. Ε, πρόσωπος των Πρασίνων μίλησε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι μια πρόοδος. Η συζήτηση που γίνεται, όντως, αλλά η συνθήκη της Λισαβόνας έθιξε για πρώτη φορά αυτό το ζήτημα. Για παράδειγμα, είπαμε ότι ανάλογα με την ε, μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο των Κρατών Μελών θα προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε το επίπεδο αποδοτικότητας των ποινικών ερευνών και αυτό θα διευκολύνει τη μεγαλύτερη συνεργασία των δικαστικών αρχών. Κάποιος δικαστής που ασκεί δίωξη βάσει μιας υποψίας ε, μπορεί να ζητήσει από τον εισαγγελέα άλλης χώρας ε, να συλλέξει τα στοιχεία, τα αποδεκτικά στοιχεία που τον βοηθήσουν ε, κατά την διαδικασία. Υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία αυτό το κείμενο. Κύριε Πρόεδρε, βλέπω ότι θέλετε να με διακόψετε, αλλά μιλώ πολύ λιγότερο από τους υπόλοιπους. Θα μείνω εδώ. Ο Πρόεδρος. Ναι, όλοι μιλούν πάνω από πέντε λεπτά όμως ε, και αυτό θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Εγώ απλώ σας παρακάλεσα να μιλήσετε τρία λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, το λέω επειδή δεν είχατε χρησιμοποιήσει το σφυράκι σας. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν ήθελα να μακρηγορήσουμε, γι' αυτό το είπα το σφυράκι, όταν το σηκώνω ψηλά θέλω απλώ να είμαι ευγενικό. Αν δεν το βλέπετε όμως και αυτό θα αρχίσω να το χτυπάω. Και όλοι το γνωρίζουν αυτό. Επόμενος ε, σκιώδης που ακολουθεί αυστηρούς κανόνες ε, πειθαρχίας, ο κύριος Δεγιόγκ Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και λεκονικός. Το πρώτο σχολείο μου Ήμουν μέλο ε, τη Επιτροπή ΚΡΙΜ τότε και προσπαθήσαμε να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο του χριστουγεννιάτικου δέντρου. Καταλήξαμε βεβαίως σε αυτό το αποτέλεσμα ακριβώ με πολλές πολύτιμες συστάσεις. Αλλά επειδή ήταν ε, τεράστιο ο κατάλογο, είναι εύκολο και για τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα να διαλέξουν αυτό που του αρέσει μόνο για να εφαρμόσουν. Ε, εν είδη γενικού κανόνα λοιπόν, ελπίζω αυτή η έκθεση να επιβεβαιώσει το κείμενο που έχουμε ήδη υιοθετήσει και ε, να, να περιοριστεί μόνο σε νέες ιδέες. Τρία στοιχεία θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτον, διεθνή συνεργασία. Σίγουρα υπάρχει έλλειμμα από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά το ΟΓΡΕΚΟ, το Συμβούλιο τη Ευρώπη ε, και τη διαφθορά. Υπάρχουν ακόμα και εντάσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΟΗΕ. Ο ΙΕ ζητά να υποβάλει εκθέσεις και δεν ακούω ε, τίποτα και για τον ε, ΟΣΑ που επίσης έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Μην μένουμε δηλαδή μόνο στα μέτρα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να προτείνουμε και στη συνεργασία της Ένωσης με, άλλα, με άλλους οργανισμούς. Επί της ουσίας τώρα άλλο στοιχείο για ε, τους δημόσιους πόρους. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό. Ιδίω ό,τι αφορά τις δημόσιες προμήθειες. Βλέπετε ότι το ελεκτικό συνέδριο ε, επισημαίνει σημαντικό ρυθμό σοβαρών σφαλμάτων. Κατά τη γνώμη μου, διερωτώ με μάλλον, είναι μόνο σφάλματα ή κάτι παραπάνω. Θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες από αυτού. Και τέλος, Κάτι το οποίο είναι σημαντικό είναι η πρόληψη. Για παράδειγμα, δημοσιογραφία. Δεν είναι μόνο έλλειψη πόρων για την ερευνητική δημοσιογραφία. Υπάρχει και αυξανόμενος εκφοβισμός των δημοσιογράφων. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και θα πρέπει να αναφέρει την προστασία των δημοσιογράφων εδώ. Αναφέραμε τους whistleblowers προηγουμένως. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ κάποιες ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε αυτό τον τομέα, αλλά και για τα κράτη-μέλη. Και νομίζω ότι είναι εφικτό να βρούμε, να καταλήξουμε σε μια διατύπωση που να αντικατοπτρίζει αυτή την ιδέα. Και άλλε διατάξει που είναι σημαντικέ. Είχαμε έκθεση στην Αργεντίνη για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Ε, ιδίως για μέτρα διαφάνεια ό,τι αφορά την ε, ιδιοκτησία. Και κάτι τελευταίο. Σύνδεση των δύο τομέων πρόληψης οργανωμένου εγκλήματος και διαφθοράς αφενός και άλλων μέσων που εγκρίνουμε. Για παράδειγμα, η οδηγία περί εμπορικών μυστικών μπορεί να υπονομεύσει ενδεχομένω τα δικαιώματα των whistleblowers. Αναφέρονται και συγκεκριμένε πρακτικέ εντό επιχειρήσεων και μετά αναφέρουμε τι μονοπρόσωπε ε, εταιρείε αυτό μπορεί να ανοίξει το δρόμο για ε, κάποιες επιχειρήσεις ταχυδρομικής στηρίδας ε, και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει συνοχή στην, στην ε, Εθνική Νομοθεσία και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Η κυρία Κάουφμαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω, αν συντομία, Καταρχάς για να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που επικεντρώθηκε σε κάποια σημεία κλειδί και πιστεύω ότι είναι πολύ καλό αυτό ε, ως βάση για τη μελλοντική μας εργασία. Το μοναδικό σημείο που ήθελα να αναφέρω στην παρούσα φάση είναι στο τέλος το θέμα της, ε, και των ε, αγαθών κοινωνική χρήση. Εδώ λοιπόν η εισηγήτρια προτείνει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο, ένα δίκτυο εθνικών ε, υπηρεσιών για την ε, διαχείριση και την αποθήκευση δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων. Δεν είμαι βέβαιη κατά πόσον σε όλα τα κράτη-μέλη υπάρχουν ε, τέτοιες υπηρεσίες αρμόδιες. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, καλώς. Ιδάλλως θα έπρεπε να απευθύνουμε έκκληση στα κράτη-μέλη να δημιουργηθούν τέτοιες υπηρεσίες. Και κατά δεύτερον, ήθελα να πω ότι δεν ε, μπορώ να καταλάβω πώς ακριβώς θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι ο τομέας αυτός, τον οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή την χρήση των πόρων για κοινωνικούς στόχους και σκοπούς, εδώ να βρεθεί λοιπόν ένας μηχανισμός ο οποίος ε, θα είναι και πρακτικός. Αυτό απευθύνω ως έκκληση στην εισηγήτρια, να κοιτάξει δηλαδή πιο πολύ τον κλάδο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Η κυρία Λόριστον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω ιδιαίτερα αυτά που είπε ο κύριος Ντογιόγκ για την ε, σημασία της ελευθερίας του τύπου και της ε, δημοσιογραφίας της διερευνητικής. Γιατί όταν κάναμε τις σχετικές αναλύσεις, κοιτάξαμε ε, αναχώρα τον δίκτυ ελευθερίας και βλέπουμε λοιπόν πόσο μεγάλη σύνδεση υπάρχει μεταξύ της ελευθερίας του τύπου και της ελευθερίας από τη διαφθορά. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε πόρους για την ελευθερία και την, ε, τα ποιοτικά μέσα ενημέρωσης. Ύστερα, να κοιτάξουμε την ψηφιοποίηση, γιατί η ψηφιακή ένωση, οι ψηφιακές υπηρεσίες δίνουν μεγαλύτερε ευκαιρίε διαφάνεια. Και θα έπρεπε να πω από την δική μου, από την δική μου εμπειρία από μια χώρα όπω η Εσθονία. 90% της φορολογίας γίνεται διαδικτυακά. Όλες οι συναλλαγές πάνω από 1.000 ευρώ πρέπει να αναφέρονται στις φορολογικές υπηρεσίες από πλευράς των επιχειρήσεων και αυτό βοηθά πολύ στο να υπάρχει έλεγχος και σωστές πληροφορίες και διαφάνεια φυσικά. Ύστερα, αυτή η νοοτροπία, η κουλτούρα της εμπιστοσύνης. Κοιτώντας και πάλι τι σχέση υπάρχει μεταξύ της ε, έλλειψης διαφθοράς και άλλων στοιχείων ε, εξαρτάται από το επίπεδο το, της ποιότητας της τη της εμπιστοσύνης στους Αυτό τι σημαίνει ότι η διαφάνεια η δημοσίευση των δεδομένων, η δημοσίευση των ε, δημόσιων διαγωνισμών, ε, των δημόσιων στρατηγικών, ψηφιακή λοιπόν ε, αγορά και διαφάνεια και έλλειψη διαφθοράς. Βασικά συστήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Χουάν Φερνάντο. Να μην χάσω την ευκαιρία να είμαι και εγώ επικοδομητικός για το θέμα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά και από την έκθεση της Επιτροπής Κρίμη για το οργανωμένο έγκλημα και τη διαφθορά στην Ευρώπη. Και κάτι που θα ήθελα να προσθέσω, γιατί δεν θα ήθελα να ξεχαστεί, είναι το εξή. Να μην υποτιμάμε τη σημασία της διασυνοριακής πανευρωπαϊκής α, παιδείας κατά της διαφθοράς. Εγώ ως ε, κάποιο που έχει εργαστεί στον τομέα του ποινικού δικαίου, πρέπει να σας πω ότι η εμπειρία μου είναι η εξή. Να μην ε, υπερβάλλουμε σε ό,τι αφορά τη σημασία του τύπου, γιατί ο τύπος σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι εξίσου διεφθαρμένος όπως και τα πολιτικά καθεστώτα. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να τονίσουμε την διάσταση της εκπαίδευσης, της παιδείας κατά της διαφθοράς από τις χαμηλότερες ε, τάξεις. Μια πηγή ελπίδας για την ανατροφή των παιδιών και των νέων με μια νέα ανατροπή, με μια νέα αντίληψη κατά τη διαφθοράς και αποτελούν και τον καλύτερο τρόπο για την καταπολέμηση της διαφθοράς ε, από την κοινωνία των πολιτών προς ε, τα θεσμικά όργανα και από τα θεσμικά όργανα προς την υπόλοιπη κοινωνία, από πάνω προς τα κάτω δηλαδή. Top down. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε σε ό,τι αφορά το τελικό σχέδιο της έκθεσης την, το οποίο συζητάμε εδώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και ε, έχουμε λίγο ξεπεράσει τα χρονικά μας όρια. Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σχολιάσει εν συντομία αν γίνεται. Ναι, καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Λάρα Φεράρα για την πολύ καλή αυτή βάση και για τη δική μας δουλειά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με μεγάλη προσοχή λοιπόν ακούσαμε τα διάφορα σημεία τα οποία ανέφερε. Θα ήθελα να κάνω κάποια λίγα σχόλια γιατί αν αρχίσω να σχολιάζω όλες τις παρατηρήσεις θα μακρηγορήσω. Θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζω τη σύνδεση αυτή που γίνεται μεταξύ διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος. Και εμείς σε μία υπηρεσία τα δουλεύουμε αυτά στην Επιτροπή. Επίσης εκτιμώ ιδιαίτερα την σχέση και τη σύνδεση ε, των δύο αυτών θεμάτων σε ό,τι αφορά και θέματα ε, του πόσο μπαίνουν στην κοινωνία. Δεν υπάρχει επίσης ένα, κανένα θέμα που να μπορεί να επιληθεί μόνο με την νομοθεσία, ακόμα και αν εφαρμοστεί στο επακρόν η νομοθεσία. Χρειάζονται και άλλα μέτρα. Ένα λοιπόν θέμα είναι, σε σχέση με την νομοθεσία, ότι θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο τομέας αυτός μέχρι πρόσφατα και ακόμα ε, αποτελεί θέμα τρίτου πυλώνα. Άρα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο και σχεδόν ανέφικτο, μη ρεαλιστικό να πιστέψουμε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν ε, πανευρωπαϊκοί κανόνες για κάποια θέματα. Συνεχίζονται μένει οι εργασίες για την αξιολόγηση της νομοθεσίας και την εκτίμηση του κατά πόσον μπορεί να εφαρμοστεί σε κάποιους κλάδους, προωθούμε και άλλα θέματα. Να θέσω δύο. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά και τις συστάσεις σας σε ό,τι αφορά την κοινωνική χρήση των ε, δημευθέντων και κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων και χρησιμοποιούμε λοιπόν μια πλατφόρμα η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή εδώ και κάποια χρόνια. Είναι πλέον λειτουργική και υπάρχει σχετική συνάντηση κάθε μήνα με τα τρία αρμόδια γραφεία και υπάρχουν ήδη και κατάλογοι με τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά πιο σημαντικό είναι ότι τώρα έχουμε αρχίσει και αναπτύσσουμε τους υπεύθυνου διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Πιστεύουμε ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο αρμόδιο για να μοιράζονται και τις ε, σχετικές εμπειρίες και προκειμένου να υπάρχουν ευρωπαϊκά δίκτυα για την κοινωνική κνέου χρήση τέτοιων κατασκευθέντων περιουσιακών στοιχείων. Ε, και, θέμα, και στο θέμα των δημοσίων συμβάσεων φυσικά υπάρχει και σχετική οδηγία. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι μία από τις βασικές διατάξεις είναι να εφαρμοστεί η ηλεκτρονική αυτή ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέχρι το 2010. Κοιτάμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη στο θέμα των δημοσίων συμβάσεων και σε τι αφορά τα ευρωπαϊκά, τους ευρωπαϊκούς ε, πόρους στο ευρωπαϊκό εξάμεινο οικονομικής διακυβέρνησης που είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί φτάνει μέχρι τους αρχηγούς κυβερνήσεων και κρατών και εδώ λοιπόν κοιτάμε τα θέματα δημοσίων συμβάσεων και τέλος με ένα πιο ρεαλιστικό τρόπο ένα κοινό project ε, των ιδιωτικών εταιριών το οποίο υποστηρίζεται και από την ε, Transparency International και άλλους τέτοιους θέματοφύλακες της διαφάνειας σε διάφορες περιοχές των κρατών μελών. Για παράδειγμα, στην έκθεση κατά της διαφθοράς, ασφαλώς εξετάζουμε όλα τα θέματα αυτά και ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή τι θα γίνει με την έκθεση μέχρι του χρόνου. Θα σταματήσω εδώ, ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, αυτό είναι το σχέδιο εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει τα συμπεράσματα εκτενών συζητήσεων. Δεν θέλω να στερήσω το χρόνο και από τα άλλα θέματα τη ημερήσια διάταξη, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Συγχωρήστε μα, λοιπόν, θα πρέπει να ολοκληρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα εν συντομία να δώσω το λόγο στην ε, εισηγήτρια, αλλά καταλαβαίνει ότι δεν έχουμε χρόνο. Σας παρακαλούμε εν συντομία. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα και από του Κιώδης. Ίσως θα μπορούσε να κάνεις κάποια καταλεκτικά σχόλια. Και φυσικά προσβλέπω και στο τελικό κείμενο της έκθεσης. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδες συγγητές και τους υπόλοιπους συναδέλφους που πήραν το λόγο για αυτά τα πολύτιμα στοιχεία που μου πρόσφεραν. Ε, βέβαια, είδα τις διάφορες απόψεις για αυτό το έγγραφο εργασίας και την τοποθέτηση γενική και έτσι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην οριστική κατάληξη, την οριστική σύνταξη. Πάντως αποτελεί άριστη αφετηρία το σημείο αυτό για να εργαστούμε από κοινού και να πετύχουμε ένα έγγραφο εργασία που να συμμεριζόμαστε όσο γίνεται περισσότερο όλοι μας. Και εκτίμησα τις διάφορες υποδείξεις για τους ε, φορολογικούς παράδεισους ε, σίγουρα θα πρέπει να εμπνευστούμε από την έκθεση που μόλις η Ειδική Επιτροπή ε, ψήφισε και μετά με τη γνωμοδότηση επίσης από πλευράς της Αρμόδιας Επιτροπής. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε όπως τα είπε και η συνάλφος Γιώτοβα της ε, σύγκρουση συμφερόντων μπορούμε να πούμε και ότι πώς διεισδύει το οργανωμένο έγκλημα ε, στους διάφορους οργανισμούς, στις τρίτες χώρες ε, για την ανθρωπιστική βοήθεια που προσφέρουμε και εκεί σίγουρα σημαντικά χρήσιμα στοιχεία με τη γνωμοδότηση ακριβώς της αρμόδιας επιτροπής. Ε, για τον πίνακα που είπε και η συνάδελφα Ζουλή, για να δείξουμε καλύτερα τη σχέση ανάμεσα στο πόσα προσφέρουν για τη δικαιοσύνη τα διάφορα τη σχέση, με τα κράτη-μέλη σε σχέση με το έπτος, χρειάζεται να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Να πω ότι αναθέσαμε στο IPRS σε αυτό το Ινστιτούτο μια μελέτη για το κόστος. Τι σημαίνει αυτό οικονομικά, επειδή ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν διαθέτουν ε, κοινή ρυθμίσεις νομοθετικές για τη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος και έτσι με την έκθεση, με τη μελέτη αυτή ίσως ληφθούν πιο συγκεκριμένα μέτρα για να φτάσουμε και σε αυτό που υπόθηκε από πλευρά συναδέλφου μέλο. Ο στόχος δεν είναι μόνο να έχουμε μια τοποθέτηση ιταλική, τη θέση την ιταλική. Έτσι πρέπει να το αποφύγουμε και χαίρομαι που όλοι οι σκιοδησιητές ανήκουν σε διαφορετικά κράτη-μέλη, Άρα λοιπόν ο καθένας θα μπορούσε να προσφέρει ένα στοιχείο ε, και σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του και τις γνώσεις του αλλά σύμφωνα και με το από ποια χώρα προέρχεται. Και τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης ε, τα οποία θα είναι σε ευρωπαϊκή κλίμακα θα αποτελέσουν βάση, περαιτέρω βάση για να μπορέσουμε να κάνουμε και συστάσεις που να συμπεριλάβουμε στην έκθεση όπως και ο Σνάφος Ντεγιόγκ για τη διεθνή συνεργασία και όσα οι περισσότεροι μίλησαν για την προστασία του δημοσιογραφικής έρευνας. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο. Ευχαριστώ και την Επιτροπή για τη στήριξή της εργασία αυτή και για τη διάφορα στοιχεία που προτείνονται για τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία και όλα αυτά θα χρησιμεύσουν στην τελική σύνταξη της εργασίας. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και τους κοιόδης και τα μέλη που συμμετείχαν ενεργά σε αυτή τη συζήτηση. Είναι πολύ καλά τα σημάδια και ελπιδοφόρα και για την ίδια την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ας προχωρήσουμε τώρα στο σημείο 26. Ε, παρουσίαση της μελέτης ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έγκριση μεταξύ συστημάτων και νομοθεσίας προστασίας δεδομένων ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ενωμένων Πολιτειών. Φρανσίσκο Μπόνι θα κάνει την παρουσίαση, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και συνεργάτη Πανεπιστημίων του στη Γερμανία και μετά θα έχουμε έναν γύρο ερωταπαντήσεων. Βεβαίω αυτό είναι κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα και με τις ε, υφιστάμενε προκλήσεις. Γιατί αυτό συνδέεται και με την γενικότερη ομπρέλα προστασία δεδομένων. Κυρία Βόενγκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου δίνετε να ε, παρουσιάσω αυτή την μελέτη. Μου ζήτησαν να κάνω μια συγκριτική μελέτη μεταξύ νομοθεσίας ε, Ευρωπαϊκή Ένωσης είπα στο ό,τι αφορά δεδομένων ε, για σκοπούς επιβολής του νόμου, αλλά και για σκοπούς ασφαλείας, γιατί αυτά συνδέονται. Αυτή η μελέτη εκπονήθηκε εν ώψη και τη μελλοντική ε, Συμφωνία Ομπρέλα και ενδεχομένω και ενό νέου ασφαλούς λιμένα. Η μελέτη αναφέρεται στην ε, εκδοχή του Σεπτεμβρίου Είχα κάνει μια πρώτη εκδοχή του κειμένου στην αρχή, πριν το Σεπτέμβρη και μετά την επικαιροποίησα. Το πρώτο βήμα της μελέτης αφορά το ενωσιακό δίκαιο και τα μέσα του Συμβουλίου της Ευρώπης και το δεύτερο αφορά συγκεκριμένες πτυχές ε, του αμερικανικού δικαίου. τα ειχέγγυα προστασία δεδομένων στο Αμερικανικό δίκαιο είναι αρκετά περίπλοκο και είναι πολύ δύσκολο να τα συγκεντρώσει κανεί όλα αυτά τα στοιχεία. Υπήρξε μελέτη του καθηγητή Μπινιάνη, Πανεπιστήμιο ε, της Ουάσιγκτον, που ανέλυε ορισμένε από αυτέ τι ε, πτυχέ. Βασίστηκα λοιπόν σε αυτή τη μελέτη και προσέθεσα ορισμένες νέες εξελίξεις όπως είναι η δικαστική προσφυγή και ε, το Freedom Act. Στο ενωσιακό δίκαιο τώρα, τα ευρήματά μας. Είναι σαφές λοιπόν ότι από το 2009 και μετά κατά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Σαββόνας έχουν ενισχυθεί ε, οι νομικές πράξεις που συνδέονται με την προστασία δεδομένων, θεωρούνται πρωταγενές δίκαιο μέχρι το 2009 δεν ήταν ε, πρωτογενής, τομέας, πρωτογενής πηγή δικαίου ή προστασία και δεν συνδεόταν με τον ε, τρίτο ή πρώην τρίτο πυλώνα. Η νομολογία ήταν περιορισμένη και γι' αυτό παραπέμπω ε, και στην ομολογία του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Αυτό θα αλλάξει τώρα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει δύο πολύ σημαντικές υποθέσεις, υπόθεση Σρέμς και συγκράτησης διατήρηση δεδομένων. Θα αναφερθώ εν συντομία σε αυτές τις δύο υποθέσεις. Βασίζονται στις πρωτογενείς πηγές δικαίου, πηγές πρωτογενείς δικαιωμάτων, άρθρο 16, άρθρο 7 του Χάρτη των Δικαιωμάτων και το άρθρο 8 του Χάρτη. Θα αναφερθώ στην πρώτη υπόθεση, διατήρηση δεδομένων γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική για την επεξεργασία των ε, δεδομένων των ε, κρατουμένων και στον τομέα επιβολής του νόμου. Το δικαστήριο λοιπόν αναφέρει γενικές αρχές που θα πρέπει να γίνονται σεβαστές σε αυτό το τομέα. Για παράδειγμα, αφορά την ε, συλλογή, διατήρηση και πρόσβαση συγκεκριμένα δεδομένα που αποτελούν ξεχωριστές παραβάσεις και έτσι απαιτείται και ξεχωριστή αιτιολόγηση. Αυτό είναι σημαντικό στη φορά την ε, διαβίβαση δεδομένων μεταξύ ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ. Αναφέρει το δικαστήριο δεν ε, έχει σημασία κατά πόσο μπορούν οι κρατούμενοι να αποδείξουν ότι υπήρξε κάποια παράβαση. Μπορούν όπως και να έχει να πάνε στο να προσφύγουν στο δικαστήριο. Απαιτείται σύνδεση με την με την απειλή στη δημοσιοσφάλεια και τα δεδομένα που έχουν διατηρηθεί. Υπάρχουν και άλλες αρχές όπως είναι περιορισμένες περίοδοι διατήρησης, διευρυμένη εποπτεία και κανόνες ασφάλειας δεδομένων που θα πρέπει να ισχύουν σε αυτό το ε, τομέα. Η υπόθεση ΣΡΕΜΣ τώρα αφορά δύο ζητήματα. Οι ε, δυνατότητες που έχουν οι αρχές επιβολής του νόμου, δεν θέλω να επιστρέψω λεπτομέρειες, όμως ε, οι αρχές προστασίας δεδομένων ε, καλούνται να ερευνήσουν αξιώσεις και αιτήματα πολιτών ακόμα και αν ισχύει η απόφαση της Επιτροπής. Άλλες πτυχές της Υπόθεση ΣΡΕΜ συνδέονται με την ακύρωση της απόφασης Safe Harbor. Το ξέρετε όλοι φαντάζομαι. Ήταν ε, πολύ σημαντική αυτή η δικαστική απόφαση. Η βασική, μαζική πρόσβαση ε, αποτελεί παραβίαση της ουσίας αυτών των δικαιωμάτων. Δεν υπήρχε ε, δικαστική αναθεώρηση, ή έλεγχος δεν υπήρχε ανεξάρτητη επιβολή. Υπήρχε και μια διάταξη που απέτρεπε την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου γιατί υπήρχε, ήταν κυρίαρχο το Αμερικανικό δίκαιο. Όλα αυτά οδήγησαν στην κατάργηση της απόφασης. Όχι μόνο στο πρωτογενές δίκαιο βρίσκουμε τέτοια πρότυπα για την επιβολή του νόμου, αλλά και στο δευτερογενές δίκαιο. Στην οδηγία 9546 πιο συγκεκριμένα, του 2002, 58, κανονισμό 45-2001 και απόφαση πλαίσια 2008-977 για την προστασία δεδομένων στον τομέα της επιβολής του νόμου. Προσπάθησα να αναλύσω όλο αυτό το πλέγμα, γιατί ε, υπάρχουν πολλά διαφορετικά στοιχεία και να εντοπίσω ορισμένες κοινέ ε, αρχές ε, σε ό,τι φορά την προστασία, την πρόταση για την προστασία δεδομένων στον τομέα επιβολής του νόμου. Κατάληξα στι αξίε βασικέ αρχέ. Βεβαίω έχουμε και την επιβολή του νόμου, πρότυπα ποιότητα που θα πρέπει να τηρούνται, ανεξάρτητη εποπτεία και αναθεώρηση, πολύ σημαντικό. καθώς και η διαβίβαση σε τρίτες χώρες. Κάποια στοιχεία θα πρέπει να ρυθμίζονται και αυτό προκύπτει και από την υπόθεση SREMS. Ε, υπάρχουν χρονικά περιθώρια για την διατήρηση δεδομένων, δικαιώματα και ένδικα μέσα των ε, προσώπων, ε, οι αυτοματοποιημένες αποφάσεις ε, και το profiling, η διαμόρφωση προφίλ, δεν πρέπει να βασίζονται σε συγκεκριμένο αλγόριθμο. Τώρα για την ομολογία του Δικαστήριου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το άρθρο 8 είναι βασική διάταξη, το γνωρίζετε. επόμενη διαφάνεια. Η νομολογία βάσει το άρθρο 8 για τα μέτρα που συνδέονται με την επιβολή του νόμου είναι ιδιαίτερα κληρωμένο γιατί το δικαστήριο ήταν αρμόδιο ε, για, αυτά τα μέτρα από το 1970 και μετά. Έχουμε λοιπόν ε, ευρύτατη ε, νομολογία από το δικαστήριο θα να δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Και πολλές φορές παραπέμπει σε αυτές τις αρχές και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σαφής προσδιορισμός των περιστάσεων και των περιορισμών της αποθήκευσης, διαφορετική μεταχείριση των δεδομένων ανάλογα με το αν πρόκειται για ύποπτα πρόσωπα ή όχι, ε, όχι στην μαζική αποθήκευση, συγκεκριμένα χρονικά όρια, όλα αυτά τα δικαιώματα που βλέπετε, μεταξύ άλλων και κοινοποίηση μετά την παρακολούθηση. Συνοψίζοντα λοιπόν ε, στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο βλέπουμε ότι και στο πρωτογενέ και στο δεύτερογενέ δίκαιο ε, παρέχεται προστασία των ε, δεδομένων και το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακολουθούν αυτή την αρχή. Τώρα περνούμε στο Αμερικανικό Δίκαιο. Έχω μοιράσει την ανάλυση σε δύο τμήματα, εχέγγυα και περιορισμοί των ε, εχεγγύων. Βλέπετε ότι είναι λίγες οι αμερικανικές εγγυήσεις. Έχουμε την τέταρτη ε, τροπολογία, ε, το Privacy Act και το Readers Act. Με τη νέα αυτή νομοθετική πράξη του 2015 για τη δικαστική προσφυγή, ε, υποτίθεται ότι υπάρχει επανόρθωση των αδυναμιών του Αμερικανικού Δικαίου, αλλά αυτό δεν ισχύει. Ουσιαστικά έχουμε τέσσερα ένδικα μέσα για τους Αμερικανούς πολίτες που θα πρέπει ε, να εφαρμόζονται και για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά αυτό δεν ισχύει σε ό,τι φορά την, ε, τον νόμο περί δικαστικής προσφυγής. Το τρίτο και τέταρτο ένδικο μέσο λοιπόν για το Privacy Act ε, είτε δεν ισχύουν είτε ισχύουν σε περιορισμένες περιπτώσεις. Το τρίτο δεν ισχύει για κανέναν. Το τέταρτο ε, ισχύει αλλά για λίγες περιπτώσεις, με πολύ περιοριστικό τρόπο. Η νομική πράξη λοιπόν περί δικαστικής προσφυγής δεν καλύπτει όλες ε, τις ελλείψεις που υπήρχαν ε, στο αμερικανικό σύστημα. Η νομική πράξη δικαστικής προσφυγής περιορίζει τις δυνατότητες προσφυγής μόνο σε λίγες περιπτώσεις αφορά μόνο τις ε, χώρες που καλύπτονται, δηλαδή έχουν υπογράψει τη συμφωνία και συμπεριλαμβάνονται στην πράξη και για τα μητρώα που καλύπτονται, δηλαδή όλα τα δεδομένα που έχουν διαβαστεί. Όχι τα δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση, για παράδειγμα, οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής. Και αυτό αφορά και τους, ε, τα πρόσωπα που καλύπτονται, δηλαδή Ευρωπαίοι πολίτες και όχι αλλοδαποί. Δύο φορές μιλούμε, γίνεται αναφορά στις, στους περιορισμούς ε, των υπολείπων ε, νομικών πράξεων και έτσι υπάρχει εξαίρεση από την υποχρέωση εφαρμογής. Και δεν είναι πολύ σαφή τα πράγματα, πώς συνδέονται δηλαδή τα δύο μεταξύ τους. άλλοι περιορισμοί ε, σε ό,τι αφορά την ε, συλλογή δεδομένων. ECPA, FISA, Patriot Act. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί ε, μπορείτε να τα βρείτε και στη μελέτη της άλλης καθηγήτριας που προανέφερα. Στο Freedom Act μόνο επιφέρει σημαντική βελτίωση ιδίω για τους Αμερικανούς υπηκόους. Για παράδειγμα έχουμε συγκεκριμένους όρους επιλογής, χρονικά περιθώρια, και ένα είδος εποπτική αρχής, αλλά μόνο για τους Αμερικανούς υπηκόους. Ε, τα υπόλοιπα που δεν έχουν τροποποιηθεί, η εκτελεστική διαταγή 1233 και κλασικές διαταγές ΦΑΙΖΑ Ακόμα και αν λήξουν όμως αυτές οι ρήτρες, υπάρχουν ακόμα νομικές διατάξεις για τη μαζική παρακολούθηση. Δεν αλλάζει αυτό με το Freedom Act. Βλέπετε ότι υπάρχουν ε, πολλά στοιχεία που μπορούμε να αναφέρουμε, πολύ περιορισμένο πλαίσιο σε φορά την ειδική σφαίρα ζωής και με τη νέα νομική πράξη για τη δικαστική προσφυγή δεν επαναρθώνεται κατάσταση όπως είπαμε, αφορά κυρίως τους Αμερικανούς υπηκόους και υπάρχουν πολύ σημαντικέ διαφορέ και είναι απαραίτητο οι ευρωπαϊκέ προποθέσει να συμπεριληφθούν σε μελλοντικέ συμφωνίε. Γιατί υπάρχουν τέτοιε προποθέσει. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Είμαι στη διάθεσή σα για τυχόν ερωτήσει. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συνάδελφοι, ε, συγγνώμη, αλλά έχουμε καθυστέρηση γιατί ξεκινήσαμε και καθυστερημένα και ζητώ συγγνώμη για το θέμα αυτό λοιπόν να περάσουμε πάρα αυτά στους κοιόδης. Να περάσουμε λοιπόν στους κοιόδης. Όποιος δεν θέλει να πάρει το λόγο, ε, δεν χρειάζεται να τον πάρει. Ο κύριος Φως. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ νομίζω καταρχάς ότι ο εισηγητής ε, θα έπαιρνε πρώτος το λόγο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν ε, κυρία καθηγήτρια για την παρουσίαση αυτή και βλέπουμε λοιπόν πόσο περίπλοκο είναι αυτό το θέμα. Αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η εκτίμησή σας. Πόσο συγκρίσιμα είναι τα συστήματα προστασίας δεδομένων ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού. Και θα μπορούσαμε να πούμε στη ΣΥΠΑ ότι υπάρχει μια κάποια προστασία ότι υπάρχει αντίστοιχο επίπεδο προστασίας. Ξέρω ότι είναι δύσκολη η σύγκριση αυτή, αλλά θα ήθελα να ακούσω τη δική σας εκτίμηση. Γιατί εγώ δύσκολα μπορώ να το εκτιμήσω. Και έχουμε ασχοληθεί με το θέμα αυτό τόσο πολύ. Ίσως εσείς όμως που έχετε παραπάνω εμπειρία θα μπορούσατε να κρίνετε με καλύτερο τρόπο και νομίζω ότι εδώ έχουμε κάνει πολλά τον τελευταίο καιρό. Έχουν βελτιωθεί κάπως τα πράγματα και γι' αυτό ενδεχομένως ε, να μπορούμε με πιο ήσυχη τη συνείδησή μας να ξεκινήσουμε και τις δημερίες διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Ο Γιωχάνες ε, δεν είναι σκιώδης γιατί είναι ασφαλώς ο εισηγητής. Αν θέλεις να θέσεις ε, ένα ερώτημα και μετά θα ακούσουμε τον Μάριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κανένα πρόβλημα για το ποιος θα πάρει πρώτο στο λόγο. Θα ήθελα να μου πείτε στην μελέτη Ένα θέμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας. Ποια είναι τα δικαιώματα τα οποία με τις ε, συλλογικές αγωγές και το ε, Umbrella Agreement καλύπτονται. Καλύπτονται δηλαδή από αυτές τις σύμφωνίες ε, τις συλλογικές. Τι επιπλέον δικαιώματα δίνονται. Μας ενδιαφέρει. Ποια είναι λοιπόν η προστιθέμενη αξία, η ενδεχόμενη προστιθέμενη αξία μιας τέτοιας συμφωνίας. Και όλα όσα κατοχυρώνονται συνάδουν ε, με τα κεκτημένα μας. Όλα όσα εντάσσονται δηλαδή στον, ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ανταποκρίνονται στο επίπεδο των όσων έχει ζητήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, που ήσασταν και σύντομοι. Μάριν Λόρσεν, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμη αυτή η έκθεση, αυτή η παρουσίαση. Γιατί είναι πάρα πολύ ωφέλιμη αυτή η πρακτική σύγκριση για μας. Ρωτώ λοιπόν, Ποια είναι η διαφορά στη γενική προσέγγιση, δεν την αναφέρατε. Οι Αμερικανοί βασίζονται πιο πολύ σε μια προσέγγιση βάση κινδύνου, εμείς όχι. Πώς μπορούμε να συγκρίνουμε λοιπόν αυτές τις δύο προσεγγίσεις, αυτά τα δύο συστήματα, έχουν υπέρ και κατά φαντάζομαι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την εφαρμογή του δικαίου, τι βλέπουμε τώρα, ότι υπάρχουν πρακτικές εφαρμογής νόμου που προέρχονται ως νοοτροπία πιο πολύ από τις είπα. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε λοιπόν αυτή τη σύγκριση της διαφορετικής φιλοσοφίας για την προστασία των δεδομένων. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Άλλος ένας ε, σκιώτης, ο Τίμωτη, δεν θέλει το λόγο. Πολύ ωραία. Ο Φερνάντο, μία τελευταία ερώτηση παρακαλώ να κάνει. Θα είμαι σύντομος. Δεν υπάρχει δικαστική αγωγή στη ΣΥΠΑ για μας, τους Ευρωπαίους πολίτες. Είναι εκπληκτικό. Υπάρχει κάποια εμπειρική αναφορά Ευρωπαίων πολιτών που έχουν ζητήσει προστασία στη ΣΥΠΑ και δεν την έχουν λάβει. Και αυτό το, αυτός ο αρνητικός αντίκτυπος για το αίτημα προστασίας δικαιωμάτων στο δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ. Ποιος είναι? Ευχαριστώ και τώρα να δώσουμε λόγο, το λόγο στην καθηγήτρια για να απαντήσει τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομη. Καταρχάς προς τον κύριο Φως ε, να απαντήσω για τη συγκρισιμότητα των νομικών συστημάτων και των δικαιωμάτων. Είναι δύσκολο να απαντήσουμε γιατί συγκρίνουμε, ξέρετε, δύο διαφορετικά πράγματα. Μίλαμε αχλάδια. Γιατί στις ΗΠΑ είναι αντίστροφα τα πράγματα από ό,τι στην Ευρώπη. Αυτό που προστατεύεται έχει να κάνει μόνο με τους ε, Αμερικανούς πολίτες. Γι' αυτό και είναι τόσο δύσκολο να υπάρξουν συγκρίσεις και επίσης είναι διαφορετικές οι νομικές παραδόσεις. Αυτό που κάνουν οι Αμερικανοί είναι να περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής των νόμων, ενώ εμείς κυρίως προσπαθούμε να τα λάβουμε υπόψη και να εφαρμόσουμε την αναλογικότητα. Και τα Freedom Act και τα Judicial Reform Act, όλα αυτά είναι πολύ περιορισμένα εξ αρχής. Έχουν να κάνουν με ένα συγκεκριμένο τομέα εφαρμογής για τους Αμερικανούς ε, πολίτες. Αυτό έχει να κάνει με τις δικαστικές σας θέλετε και προφανώς ε, σημαίνει μια τεράστια διαφορά. Άρα δεν ε, υπάρχει κάποιο περιεκτικό privacy framework στην Αμερική. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ανάλογα δικαιώματα σε καμία περίπτωση. Για τον κύριο Αλμπρέχτ κατά πόσον ε, η συμφωνία ομπρέλα αυτή, η συμφωνία πλαίσιο αυτή έχει επιπρόσθετη ευρωπαϊκή αξία, κατά πόσον μπορεί να ενταχθεί στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, είναι τμήμα του Privacy Act ε, των δικαιωμάτων που ε, αφορούν τον πολίτη, αλλά ένα πολύ μικρό τμήμα. Η μία δυνατότητα προάσπιση δικαιωμάτων είναι ανύπαρκτη, κάποιες άλλες είναι πολύ πολύ περιορισμένες. Και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι περιορισμένες. Γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι ό,τι ισχύει για τους Αμερικανούς στο Privacy Act θα μπορούσε να ισχύει και για τους Ευρωπαίους. Και πάλι δεν θα υπήρχε συγκρισιμότητα γιατί και πάλι οι νόμοι θα ήταν σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από ό,τι αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, στο θέμα της διαφορετικής προσέγγισης. Ναι, όπως είπατε. Όπως είπα, λοιπόν, στα αγγλικά συνεχίζει η ομιλήτρια. Το πεδίο εφαρμογή της νομοθεσίας είναι πολύ περιορισμένο στις ΗΠΑ. Μεγάλη διαφορά. Εμείς ως Ευρωπαίοι προσπαθούμε να τα ζυγίσουμε τα πράγματα κατά περίπτωση, να τα δούμε ποια είναι η αναλογικότητα. Δεν υπάρχει αυτό στην Αμερική. Περιορίζεται το πεδίο εφαρμογή και μόνο σε αυτό το περιορισμένο πεδίο εφαρμογή ισχύουν οι νόμοι και αυτό αποτελεί μια βασική διαφορά. Πέρα από τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων το θέμα της ιδιωτικής σφαίρας του privacy δεν είναι θέμα θεμελιδός ε, δικαιώματος των Ευρωπαίων πολιτών, μόνο για Αμερικανούς. Αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά. Τα εμπειρικά αρχεία για τους Ευρωπαίους πολίτες που ζητούν ένδικα μέσα στις ΗΠΑ. Εγώ αναμίχθηκα λίγο στην ε, υπόθεση ΣΡΕΜΣ και προσπαθήσαμε και στο παρελθόν να ζητήσουμε τη χρήση ενδικών μέσων στη ΣΥΠΑ. Δεν υπήρξε απάντηση, δεν υπήρξε καμία επιτυχία. Κάθε φορά λαμβάναμε μία επιστολή που μας έλεγε ουσιαστικά ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς, πάτε πουθενά άλλο. Να απευθυνθείτε. Θα σε ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος για την έκθεση και για την παρουσίαση της έκθεσης σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι που ήσασταν και τόσο σύντομοι για το θέμα αυτό. Μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτά που προβλέψαμε μέσω email. Το επόμενο θέμα του Τίμωθη Κέρκοπ που δεν μπόρεσε να μας ενημερώσει χθε για την εξέλιξη των τριμερών διαλόγων για το PNR, ε, επειδή είχε πρόβλημα να καταφτάσει εδώ στη συνεδρίαση. Να δώσουμε το λόγο στον Τίμο πρώτα για το θέμα του PNR. Άρα, συνάδελφοι, θα μας παρουσιάσετε η Θή τι γίνεται με τους τριμερείς διαλόγους για το θέμα του PNR. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, να δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Κυρκόβο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ χθε. Υπήρχαν διάφορες δυσκολίες στο σύστημα μεταφορών ανά την Ευρώπη. Φαντάζομαι τα ακούσατε. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση για το PNR. Έχουν γίνει τέσσερις τριμερείς διάλογοι και η πέμπτη προβλέπεται για αύριο συνάντηση έχει σημειωθεί σημαντική προόδο για πολλά κύρια ζητήματα και είμαι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξει συμφωνία μέχρι τα τέλη της χρονιάς. Βεβαίω, βασίζομαι και στη στήριξη των συναδέλφων μου εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στο Συμβούλιο προκειμένου να επιτευχθεί αυτό ο σκοπό. Και ελπίζω η αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων να συνεχιστεί όπω έχει γίνει μέχρι τώρα. Ας σας ε, περιγράψω την κατάσταση για τα κύρια ζητήματα. Πρώτον, για τις πτήσει εντός τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Συμβούλιο ξεκάθαρα ανέφερε ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να συμπεριληφθούν ε, στο πεδίο εφαρμογή τη ε, οδηγία. Τα κράτη-μέλη θεωρούν ότι οι πτήσει εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμπεριληφθούν, ούτω ώστε να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία και η διακίνηση ε, ανθρώπων, ναρκωτικών ουσιών και άλλων κατηγοριών εγκληματικών δραστηριοτήτων να είναι πιο σημαντική η, αυτή η καταπολέμηση. Εάν δεν υιοθετηθεί το μέσο ε, σύντομα, τα κράτη-μέλη ε, δεν θα ε, οδηγηθούν σε κανένα εναρμονισμένο σύστημα PNR και θα διαμορφώσουν εθνικά συστήματα PNR με αποκλίνοντες κανόνες, ιδίως ό,τι αφορά τις δικλείδες ασφαλίσεις και την προστασία δεδομένων. Σε ορισμένα κράτη-μέλη, Πρόεδρε, 80% των δεδομένων πτήσεων είναι, αφορά πτήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο βεβαίω διατηρεί επιφυλάξει ό,τι αφορά τη συμπεριλήψη των ε, ε, δεδομένων πτήσεων εντό Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει. Για την περίοδο κράτηση και διατήρηση των δεδομένων. Είναι κάτι το οποίο εξετάσαμε εντελεχώ. Το ζήτημα αυτό βεβαίω είναι ιδιαίτερα λεπτό και υπάρχει σημαντική απόκληση στη θέση των τριών θεσμικών οργάνων καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Μετά από μακροσκελείς συζητήσει, πιστεύω ότι κινούμαστε προς ε, μια συμβαστική λύση στην οποία να μπορούμε να αποτεχθούμε όλοι. Το Συμβούλιο αρχικά ζήτησε πέντε έτη, ενώ το Κοινοβούλιο 30 ημέρες. Επομένω, είναι σαφές ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν κάπως πίσω. Όμως, ε, ό,τι και αν ε, αποφασίσουμε τελικά, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να είναι αναλογικό. Οτιδήποτε είναι πάνω από 12 μήνες, κατά τη γνώμη μου δεν είναι αναλογική λύση. Και σε αυτό θα ήθελα να επιμείνω, Πρόεδρε. Πεδίο εφαρμογή οδηγία. Εξετάσαμε και αυτό το θέμα. Το Κοινοβούλιο ήθελε έναν κλειστό και συντομότερο κατάλογο και αυτό αποτελεί προτεραιότητα και για το Κοινοβούλιο και για μένα προσωπικά ως εισηγητή. Η συζήτηση για τον κατάλογο των αδικημάτων και κατά πόσο θα πρέπει να συμπεριληφθούν και τα για το διεθνέ έγκλημα, τα διεθνή αδικήματα θα πρέπει να συνεχιστεί. Η πρόταση του Κοινοβουλίου για την συμπερίληψη PNR ε, για τους non-carrier οικονομικούς φορείς. Ε, το Συμβούλιο αναφέρει ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην ε, συμβαστική πρόταση του Συμβουλίου της Προεδρίας, γιατί αυτό θα δημιουργήσει τεχνικές ε, δυσκολίες για τα κρατημέλη. Δεν θέλει το Συμβούλιο να επιφορτήσει τα κρατημέλη με αυτό το άχθος ε, συλλογή δεδομένων που κανονικά δεν θα συνέλεγαν. Επίσης υπάρχει προβληματισμός ότι τα δεδομένα αυτά δεν θα είναι αρκετά ποιοτικά. Ταυτόχρονα τα κράτη-μέλη θέλουν να αποφύγουν ε, κενά στην ασφάλεια. Γι' αυτό το λόγο το Συμβούλιο πρότεινε μία βαθμιδών προσέγγιση οι εθνικές αρχές ε, μπορούν να τα ελέγξουν αυτούς τους μηχανισμούς υπό το εθνικό τους πλαίσιο και ε, στο μέλλον θα μπορούσαμε να εξετάσουμε βάση στοιχείων αν είναι, πρέπει να γίνει υποχρεωτικό ή όχι. Μπορούν και είναι διατεθειμένοι η Επιτροπή μάλλον να εξετάσει αυτή την επιλογή, αλλά θα χρειαστεί χρόνο για να το δει. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών προτείνει το Κοινοβούλιο άρθρο 7. Συζητήσαμε και το άρθρο 7 με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που προτείνει το Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο δεν δέχεται τα δεδομένα να ανταλλάσσονται αυτομάτως. Συμβούλιο και Επιτροπή θεωρούν ότι η αυτόματη ανταλλαγή όλων των στοιχείων δεν θα πληρεί τις προϋποθέσεις που μας απασχολούν ιδιαίτερως, αναγκαιότητα και αναλογικότητα. Όμως, Πρόεδρε, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γίνεται η ανταλλαγή ε, σχετικών συναφών και χρήσιμων πληροφοριών. Αυτό είναι κύριο ζήτημα αν θέλουμε να ε, θεσμοθετήσουμε ένα μέσο που κατά τη γνώμη μου είναι και αποτελεσματικό και πολύτιμο. Ανταλλαγή δεδομένων PNR με την Europol. Βεβαίως και θα ήθελα η Europol να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οδηγία. Η Επιτροπή επισημαίνει την ότι η ανταλλαγή αυτή με την Europol θα πρέπει να συνάδει και με την νομική της βάση υπό τον νέο κανονισμό 2. Η σύνδεση μεταξύ PNR και του νέου πακέτου προστασίας δεδομένων. Οι διαπραγματεύσεις για τη ε, διασύνδεση αυτή συνεχίζονται. Το Συμβούλιο προτείνει να γίνει μια δυναμική παραπομπή στην νομοθεσία προστασίας δεδομένων σε αυτή την οδηγία PNR. Πρόεδρε, κάτι στο οποίο είμαι αδιάλακτος είναι μια πλήρης, ένας πλήρης και εύρωστος μηχανισμός αναθεώρησης. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι η νομοθεσία που θα υιοθετήσουμε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα λειτουργεί, θα είναι αποδοτική και θα λειτουργεί σωστά μετά από ένα ε, εύλογο χρονικό διάστημα. Και πάνω απ' όλα, Πρόεδρε, θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε οι προϋποθέσεις που έχουν θεσμοθετηθεί από την δικαστική απόφαση του δικαστηρίου για την διατήρηση δεδομένων θα αντικατοπτρίζονται και σε αυτή τη διαδικασία αναθεώρησης. Αυτό είμαι ε, πολύ συγκεκριμένος, το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Αυτά εν συντομία, Πρόεδρε. Ο επόμενος τριμερής διάλογος θα διεξαχθεί αύριο και ελπίζω και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία την οποία θα μπορέσει να στηρίξει η πλειοψηφία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συνάδελφοι, συνήθως ε, δεν υπάρχουν ερωτήσεις σε ό,τι φορά την ενημέρωση για τους τριμερείς διαλόγους. Έχουμε σκιώδεις και δύο συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Δεν έχουμε χρόνο. Έχουμε και άλλα σημαντικά θέματα στην διάταξη. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω τώρα, εάν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο για να κλείσουμε τον κατάλογο μελητών. Παρακαλώ πείτε μας τώρα, αν θέλετε να πάρετε το λόγο. Σηκώστε το χέρι σας παρακαλώ για να σας σημειώσουμε. Not if you're an assistant, obviously. Um, I'm just doing this because... Το κάνω αυτό για να έχουμε χρόνο και για τα άλλα σημεία της ημερής διάταξης. Okay, you may now... Can they put their hands yes. down now? Yes. Okay, you can put your hands Κατεβάστε τα χέρια. Να ακούσουμε λοιπόν όλα τα μέλη της Επιτροπής. Ε, προφανώς δεν θα πρέπει να ξαναξεκινήσουμε όλη την συζήτηση. Σας παρακαλώ λοιπόν να είμαστε συνοπτικοί, γιατί δεν μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε όλη τη συζήτηση για το PNR. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Φως. Σας παρακαλώ να είστε πολύ σύντομοι. Ναι, κοιτάξτε, θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω για την καλή εργασία. Ο εισηγητή παρουσίασε πάρα πολύ καλά πόσο διαφοροποιημένε και αποκλίνουσε είναι οι απόψει, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά και μεταξύ των δεσμικών οργάνων. Και νομίζω ότι απέδειξε πόσο απομονετικό είναι. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια μα υπέβαλε πολύ καλέ προτάσει. Και νομίζω δεδομένου και του πόσο επίγοντο είναι το θέμα αυτό, πόσο επίγοντο είναι το θέμα αυτό, ε, καλό θα κάναμε να ολοκληρώναμε λοιπόν το θέμα αυτό και γι' αυτό λοιπόν δεν θα μακρηγορήσω και να ευχαριστήσω πολύ τον ε, συνάδελφο. Η κυρία Σίπελ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πάντα καταλάβαινα ότι ρόλος του εισηγητή ήταν ο εξή. Εφόσον υπάρχει εντολή διαπραγμάτευσης, φυσικά ο εισηγητή θα πρέπει να ακολουθήσει την εντολή αυτή και θεωρώ ότι ο Τιμωθή λοιπόν θα συνεχίσει να το πράττει αυτό. Παρ' όλα αυτά, πώς να το πω, φιλικά και ευγενικά. Είμαι κάπως ε, συγχυσμένη για κάποιες από τις προτάσεις του Συμβουλίου. Είναι πάρα πολύ κατεπήγον να ψηφίσουμε το συντομότερο δυνατόν, όχι μόνο τον Γενάρη, πολύ πιο νωρί. Γιατί, αναρωτιέμαι, ο εισηγητής αρχικά είχε προβλέψει περίοδο μεταβατική τριών ετών. Δύο έτη τώρα πλέον. Άρα τι διαφορά έχει αν αποφασίσουμε τώρα σε δύο ή τέσσερις εβδομάδες. Έχει ακόμα χρόνο μπροστά μέχρι να εφαρμοστεί. Είμαι επίση αισιόδοξη για το γεγονό ότι στο πακέτο για την προστασία των δεδομένων σημειώνεται πρόοδο. Καλό αυτό. Αυτό θα έχει επιπτώσει και για του επιβάτε, αλλά τώρα απειλούμαστε ότι αν δεν συμφωνήσουμε γρήγορα γρήγορα, βιαστικά βιαστικά, θα προχωρήσουν μόνο του τα κράτη-μέλη και τότε θα είναι πολύ κακά τα πρότυπα προστασία των δεδομένων. Πραγματικά ενοχλούμε, ενοχλούμε. Γιατί αν ε, δηλαδή ακολουθήσουν μόνο τους την οδό αυτή τα κράτη-μέλη θα είναι κακό το πακέτο. Τι, τι, τι, σχέδια είναι αυτά και ελπίζω, εν περιπτώσει, ο εισηγητής να συνεχίσει να προσπίζει τα όσα συμφωνήθηκαν στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας υπενθυμίσω ότι και στα τρία κείμενα διαπραγμάτευσης οι ενδοευρωπαϊκές πτήσεις δεν συμπεριλαμβανόντουσαν. Γιατί να συμπεριληφθούν τώρα λοιπόν σε αυτό το τελικό αποτέλεσμα και κατά δεύτερον, ακούσαμε μία παρουσίαση στην αίθουσα που αφορούσε και τις ε, δικαστικές υποθέσεις και μας υπενθύμησε ότι το δικαστήριο πρόσφατα αποφάνθηκε ότι η μη διακριτική διαχείριση των δεδομένων δεν συνάδει με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε κατά κάποιο τρόπο να μπει και αυτό στην οδηγία. Ευχαριστώ. Στία, Δίας Δεμέρα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω λοιπόν μία δήλωση. Μία δήλωση για τον κύριο Κίρκοφ και την εργασία του ο οποίος προσέφερε ιδιαίτερες υπηρεσίες. Ξέρετε τι είναι να αντιπαρτεθεί κανείς στο οργανωμένο έγκλημα, στην τρομοκρατία, αλλά εδώ ορίστηκε ακριβώς για το PNR το ευρωπαϊκό ορίστηκε σαν εισηγητής είναι, πρόκειται για ένα εργαλείο ιδιαίτερα χρήσιμο, απαραίτητο, ώστε οι δημοκρατικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσουν να εγγυηθούν καλύτερα την ασφάλεια των Ευρωπαίων και να πολεμήσουν το έγκλημα σε κάθε εκδήλωσή του. Κατά την άποψή μου κύριε Πρόεδρε το Κοινοβούλιο θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και των υποχρεώσεών του. Ακριβώς όπως το κάναμε πολλές φορές. Είμαστε υπεύθυνοι, το δείξαμε πολλές φορές και νομοθέτες και πολίτες μας κοιτάζουν με μεγάλη προσοχή. Υποστηρίζω την εργασία του κύριου Κύρκοφ. Είναι η πρέπουσα, η αρμόζουσα προσοχή και να μπορέσουμε να ψηφίσουμε θετικά το ευρωπαϊκό ΠΕΝΑΡ και αυτό πριν να τελειώσει ο χρόνος. Γιατί τρέχει το έγκλημα πολύ πιο γρήγορα από την νομοθεσία. Γι' αυτό ακριβώς λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μειονέκτημα και θα πρέπει να το καταλάβουμε και για τους άλλους, για μένα, για την ομάδα μου. Αυτό το πράγμα αποτελεί μια ύψιστη προτεραιότητα. Τίποτα άλλο κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Άννα Ευχαριστώ κύριε Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία σε ό,τι αφορά αυτήν την αντίσταση που αναφέρατε για, τους, ε, για συγκεκριμένη κατηγορία εμπορευομένων. Μιλάτε για τις πτήσεις τσάρτερ που θα συμπεριλαμβάνονται ή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και θα, τους, και θα καλούνται να δώσουν στοιχεία ή θα εξαιρούνται. Και ποια θα είναι, τι αξία θα έχει το PNR αν υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κύρκο και όπως είπε και ο συνάδελφος πριν από λίγο έχει τη χάνει της υποστήριξής μου άλλωστε όπως από την αρχή για αυτό το δύσκολο έργο Παρακαλώ μήπως θα μπορώ να πω κάτι σχετικά με την εφαρμογή επειδή είναι κατεπήγον το θέμα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν να, έχω τη δυνατότητα, να έχουμε τη δυνατότητα να επιταχύνουμε όπως ακριβώς και άλλες φορές και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Τιμωθή μίλησες για 12 μήνες τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό που προτείνεις για 12 μήνες ή μήπως κάτι λιγότερο και κάτι ακόμα υποστηρίζω και, τα ενδο, και τις ενδοκινοτικές πτήσεις. Συμφωνώ ότι ε, αν δεν το κάνουμε θα συνεχίσουμε με το PNR το δικό τους και θα έχουμε την ίδια κατάσταση όπως ίσχυε μέχρι τώρα και δεν θα έχουμε πετύχει τίποτα. Ευχαριστώ. Ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κέρκοβ για την αισιόδοξη έκθεσή του και ιδίω για τις ε, διασφαλίσεις που μας δίνει ότι όλες οι πολιτικές ομάδες μπορούν ε, να εργαστούν από κοινού. Παρόλε τι διαφωνίες μας νομίζω ότι όλοι μπορούμε να... Ε, ότι έχουμε ένα κοινό στόχο και ότι όλοι θέλουμε αυτό το πακέτο και πραγματικά νομίζω μπορούμε να πετύχουμε αυτό τον ε, σκοπό ε, και το PNR και το πακέτο ψήσεων να κατευθύνονται προς ε, τον ίδιο σκοπό, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων κτλ. Με εξέπληξε αυτό που είπατε για τη δυναμική παραπομπή το πακέτο προστασία δομένων. Δεν κατανοώ τι ακριβώς εννοείται με τον όρο δυναμική παραπομπή. Ξέρουμε πολύ καλά τι, συνέβη όταν, τι συμβαίνει όταν έχουμε οδηγία ή κανονισμό. Είναι σημαντικό να υπάρχει συνοχή μεταξύ των δύο και, να, και των δύο να έχουμε ένα συγκεκριμένο σαφές πλαίσιο. Κύριε Κάκοβ, θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ. Να απαντήσω σε ορισμένες από τις παρατηρήσεις, ίσως όχι σε όλες. Όπως ξέρετε, είναι μια διαδικασία που διαρκεί εδώ και πολύ καιρό τώρα και είχαμε κάποια σύνθετα ζητήματα τα οποία ακόμα τα εξετάζουμε. Δεν θέλω λοιπόν να προδικάσω το τελικό αποτέλεσμα. Απλώς επεσήμανα του τομείς στους οποίους θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης ή ευελιξίας και του τομείς όπου δεν υπάρχει τέτοιο. Ιδίω το θέμα των περιόδων διατήρησης. Ήθελα να το επισημάνω. Είπα στις παρατηρήσεις μου ότι η παρούσα πρόταση για την διατήρηση δεδομένων για μια περίοδο που οι προτάσεις Άλλη πρόταση έκανε λόγο για 5 έτη, για άλλη για 30 ημέρες. Υπάρχει λοιπόν ε, μεγάλη συζήτηση. Προσωπική γνώμη τώρα. Και νομίζω ότι και άλλοι συναδελφοί συμφωνούν μαζί μου ότι οι πρόταση, προτάσεις άνω των 12 μηνών δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. Για πολλούς λόγους. Βεβαίως και ασκώ μεγάλες πιέσεις. Είναι δύσκολη κατάσταση γιατί και το Συμβούλιο είναι ιδιαίτερα αποφασισμένο και κάνει σκληρή διαπραγμάτευση. Θέλουν πραγματικά να διατηρήσουν τις προτάσεις άνω των 12 μηνών. Εγώ λοιπόν επιμένω από πλευρά μου. Το άλλο ζήτημα τώρα. Για τους οικονομικούς φορείς που δεν είναι μεταφορείς, non-carrier economic operators. Και εδώ υπάρχει μια διάσταση απόψεων και στο Κοινοβούλιο και εκτό σε ό,τι αφορά τι υποχρεώσεις για συγκεκριμένε κατηγορίες όπως είναι οι τσάρτερ εταιρείε και άλλες. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όπου από ό,τι φαίνεται κάθε χώρα έχει διαφορετική άποψη. Θα ήθελα εδώ να δω κατά πόσο θα μπορούσαμε ε, να ακολουθήσουμε μια σταδιακή ε, προσέγγιση, step by step, ούτως ώστε οι εθνικές αρχές να εξετάζουν κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα ε, είναι απαραίτητο να υπάρχει υποχρετική κάλυψή τους. Θα ήθελα όμως τώρα από την Προεδρία να λάβω κάποια επιβεβαίωση ως προς την καλύτερη θέση που μπορούν να προσφέρουν προς το Κοινοβούλιο. Παρεμπιπτόντως, ε, το χρονικό πλαίσιο. Κανείς δεν μπορεί νομίζω να με κατηγορήσει ότι προσπαθώ ε, να περάσω έτσι να το οτιδήποτε από το Κοινοβούλιο. Παρόλα τα φρικτά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο αυτή τη στιγμή, που τείνουν να οθούν τους πολιτικούς να δρουν ε, γρήγορα και βεβαιασμένα. Εγώ είμαι πολιτικός και όπως είπατε και εσείς ε, πολύ ευγενικά και στο παρελθόν έχω έρθει αντιμέτωπος με τέτοια φαινόμενα τρομοκρατίας όπως έχουμε λοιπόν άμεση εμπειρία. Όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν είναι σωστό να αντιδρούμε γρήγορα και βεβαιασμένα όσο επίγουσες και αν είναι, σε, και οι καταστάσεις. Όμως αυτό το μέτρο έχει δει πολλές δημοκρατικές επιθέσεις να συμβαίνουν ενώ εμεί συζητούμε αυτά τα μέτρα. Τώρα λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο που πιστεύω ότι μπορούμε να κλείσουμε μια συμφωνία και με τα άλλα θεσμικά όργανα και θα αντανακλά με πολύ καλό τρόπο και τους προβληματισμούς του Κοινοβουλίου. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να επιτύχω, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Αν δεν ξέρετε, η τελευταία τρίγμερη διάλογο είναι αύριο και θα ακούσουμε ένα ευθετό χρόνο ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή. Ευχαριστούμε και του ε, συναδέλφου που ήταν τόσο συνοπτικοί. Και πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο και πάλι αφορά τον κύριο Κέρκοπ πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την παρουσίαση της ε, ερώτησης για τα hotspots και τις κρατικές αυτές δράσεις. Να ρωτήσω τον εισηγητή κατά πόσον θέλει να κάνει κάποια εισαγωγικά σχόλια. Έχετε το λόγο. Όντως, πρόεδρε, δεν θα μακρηγορήσω. Νομίζω ότι ήδη έχω απασχολήσει πολύ την Επιτροπή και καλό είναι να μην εξαντλήσω την υπομονή σας και την καλή σας θέληση, αλλά είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η έκθεση για την επανεκατάσταση θα αποτελέσει εκ νέου ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας, γιατί η ασφάλεια και όχι τόσο η μετανάστευση έχει κυριαρχήσει στα, στις ειδήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Αλλά αυτό νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάσει τις αποφάσεις που θα πρέπει να λάβουμε για τη μετανάστευση και δεν έχουν ναι, καταστεί λιγότερο εύκολες αυτές οι αποφάσεις. Χρειάζεται λοιπόν πολιτική βούληση για να εξευρεθούν λύση, λύσεις. Και η επανεγκατάσταση προβάλλεται ως μία λύση τέτοια. Ως εισηγητής λοιπόν πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός ο οποίος δεν θα πολλώσει περαιτέρω, θα πρέπει να συνάδει επίσης με το νομικό μας πλαίσιο και τις ε, κανονισμούς του Δουβλίνου και τους ελέγχους εξωτερικών συνόρων και οποιοδήποτε μηχανισμός ε, τέτοιος θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα εύρυθμα λειτουργών σύστημα για την μετανάστευση. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτή την μεταεγκατάσταση, πρέπει να έχουμε στην υπόψη μας ότι για να λειτουργήσει ένα τέτοιο μόνιμο σύστημα μετεγκατάστασης θα πρέπει και το κεκτημένο να θεωρείται ότι λειτουργεί σωστά στο σύνολό του. Αυτή η μετεγκατάσταση θα λειτουργήσει μόνο εφόσον υπάρχει εμπιστοσύνη και στην παρούσα φάση πρέπει να ομολογήσω ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερε τέτοιε ενδείξει για εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα ελαττώματα των κατεπηγών των μηχανισμών ε, μετεγκατάστασης και να διδαχθούμε όταν θα κληθούμε να οικοδομήσουμε ένα πιο μόνιμο τέτοιο μηχανισμό. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτός ο μηχανισμός ε, κατεπήγουσης κατάσταση δεν λειτουργεί όπως θα έλειψε και το Κοινοβούλιο και κάποια κρατημέλη. Χρειάζεται ένα πολύ πιο στεναρό πλαίσιο από αυτά που παρουσιάζαμε ως τώρα. Χρειαζόμαστε το μηχανισμό αυτό προκειμένου να κοιτάξουμε και άλλα θέματα όπως ε, η κατανομή, οι αγωγές, οι επιστροφές, η χρηματοδότηση, η ένταξη, η συνοριακή έλεγχη, η εξέταση των ε, αιτήσεων. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε συνολικά και δεν θα πρέπει να τα πασαλείψουμε βιαστικά αυτά για να είναι τάχα αποτελεσματική η εφαρμογή. Γιατί τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ταιριάζουν όχι μόνο για αυτή την κρίση, αλλά και για κάθε μελλοντική κρίση η οποία ενδέχεται να ακολουθήσει σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα. Άκουσα ότι οι σοσιαλιστές δημοκράτες, το ΕΛΚ και άλλες ομάδες έχουν ζητήσει μία προσέγγιση πακέτου συνολική. Και ως εκ τούτου είμαι να συνεργαστώ στενά με την κυρία Γκριγιόμ τις επόμενες εβδομάδες για να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε από κοινού προς τα εμπρός. Ελπίζω να έχω έτοιμη την έκθεσή μου για να σας την παρουσιάσω και στην Επιτροπή στις αρχές του επόμενου έτους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα να ακούσουμε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι έχει να μας πει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πρότασή του για τον ε, έκτακτο μηχανισμό μετακατάστασης υιοθετήθηκε από την Επιτροπή στις 9 Σεπτεμβρίου με τη βάση του άρθρου 78 τροποποίηση του κανονισμού του Δοβλίνου. Για να σας δώσω ένα πλαίσιο, το ευρύτερο πλαίσιο. Και το Σεπτέμβριο είχαμε δύο έκτακτους ε, μηχανισμούς ε, μετακατάστασης που τέθησαν σε ισχύ από την Ιταλία και την ε, Ελλάδα. Συνολικά 160.000 ετούντες εμπλέκονταν. Τώρα γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει έναν μόνιμο μηχανισμό μετεγκατάστασης. Το άρθρο 78.3 που χρησιμοποιήθηκε για τις πρώτες ε, δύο περιπτώσεις που προανέφερα ισχύει μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ε, με έκτακτες δηλαδή ροές μεταναστών. Δεν αρκεί όμως αυτό το δυναμικό πλαίσιο για έναν μόνιμο μηχανισμό μετακατάστασης. Ισχύει μόνο δηλαδή για έκτακτες περιστάσεις. Και επίσης είχαμε την αίσθηση ότι αν βασιστούμε στο 78.3 παρεμβαίνουμε στις αποφάσεις του κανονισμού του Δοβλίνου για βάσει του οποίου τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για τις διαδικασίες ασύλου. Γι' αυτό πρέπει να γίνει πρόταση στο πλαίσιο του κανονισμού του, Δουβλίνου ε, και μια πρόταση που συνδέεται με το, 70, με το άρθρο 78. Γι' αυτό η Κομισιόν μετά τους δύο έκτακτους μηχανισμούς ε, πρότεινε να υποβάλει αυτή την πρόταση. Τώρα, τι συμπεριλαμβάνει η πρόταση συμπεριλαμβάνει εξουσιοδότηση προς ε, την ε, Επιτροπή να κινητοποιήσει τον μηχανισμό μετεγκατάστασης από τα κρατημέλη εάν ε, διαπιστώσει ότι το κράτος μέλος έχει αντιμέτωπο με μια σοβαρή και έκτακτη κατάσταση κρίσης. Εδώ έχουμε ένα πολύ πιο συγκεκριμένο και ασφαλώς προσδιορισμένο πλαίσιο από ό,τι αυτό που προκύπτει από το άρθρο 98.3. Η κατάσταση κρίση διαπιστώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν η κρίση δηλαδή είναι τέτοιου μεγέθου, ούτω ώστε να ασκεί τεράστια πίεση και είναι επιλεσματικό αυτό, ακόμα και για ένα καλά προετοιμασμένο σύστημα ασύλου, το οποίο λειτουργεί ε, βάσει όλων των ε, σχετικών πτυχών του ευρωπαϊκού κεκτημένου επί του ασύλου. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των ετούντων και των ε, γενικών αφήξεων τους προηγούμενους έξι μήνες. Η αύξηση των ε, αριθμών σε σχέση με την ίδια περίοδο την προηγούμενη χρονιά και τον αριθμό των ετήσεων κατά κεφαλήν ετήσεων... κατά τους προηγούμενους 18 μήνες. Για να προσδιορίσουμε τώρα τον αριθμό των προσφύγων, των ετούντων άσυλο που θα πρέπει να μετακατασταθούν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, και τον αριθμό των ετούντων κατά κεφαλήν στα κράτη-μέλη τους τελευταίους 18 μήνες, τη δυνατότητα των κρατών μελών, την ικανότητα δηλαδή ε, του συστήματος ασύλου και τη συμμετοχή των κρατών μελών σε προηγούμενες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης. Δηλαδή, εάν ένα κράτο μέλο συμμετείχε κατά το παρελθόν σε άλλα μέτρα αλληλεγγύη και αυτό θα λαμβάνεται υπόψη εδώ. Η πρόταση συμπεριλαμβάνει ε, μια κλίδα κατανομής που βασίζεται σε τέσσερα κριτήρια, 40% πληθυσμό, 40% ΑΕΠ και το υπόλοιπο 20% ε, διορθωτικά κριτήρια όπως είναι ο κατακεφαλήν αριθμός ε, τον άσυλο 10% και 10% συνδέεται με το ποσοστό ανεργίας αυτό το κράτος μέλος πεδίο εφαρμογή του μηχανισμού θα ισχύει μόνο για υπηκότητε που αναγνωρίζονται γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση άνω του 75% για να δίνουμε τη μέγιστη ε, διασφάλιση στο κράτος μέλος μετακατάστασης ότι τελικά δεν θα λάβει έναν ε, παράτυπο μετανάστη αλλά θα είναι πιο πιθανό να, δώσει, να υποδεχθεί κάποιον στο οποίο θα αποδοθεί το καθεστώ του πρόσφυγα. Τώρα έχουμε και συμπληρωματικά μέτρα, ένα οδικό χάρτη που θα δίνεται από το κράτο μέλο από το οποίο θα γίνεται μετακατάσταση και εφόσον ε, βρισκόμαστε στο πλαίσιο του Δουβλίνου, αυτό συνδέεται και με το άρθρο 33, Μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων. Οι διαδικασίες είναι οι ίδιοι με το άρθρο 783. Πολύ σημαντικό είναι, και εδώ παρπέμπω και στα σαγωγικά σχόλια του κ. Κέρκοβ, του εισηγητή, ο μηχανισμός προβλέπει πιο συγκεκριμένα κανόνα για να αποτρέπονται οι δευτερογενείς ε, κινήσεις, μετακινήσεις μάλλον. Τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να επιστρέφουν έναν ετούντα άσυλο που έχει κρυφά και παρανόμως ε, μετακινηθεί σε δεύτερο κράτος μέλος. Ο εισηγητής είπε για το δεύτερο ότι πρώτα πρέπει να αποκτήσουμε εμπειρία με τους έκτακτους μηχανισμούς. Κλείνοντας τις παρατηρήσεις μου, θα ήθελα μόνο να πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εν μέσω μια σοβαρής κρίσης που αποσταθεροποιεί ολόκληρο το σύστημα Σέγγεν και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι της γνώμης ότι Πρέπει να έχουμε αξιόπιστο και πολύ συγκεκριμένο και στεναρό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να είναι ο κανονισμός του Δουβλίνου, γι' αυτό και υποβάλλουμε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τώρα να δώσουμε το λόγο στην Προεδρία για να μας ενημερώσει. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο να σας πω ότι για την εργασία, για την πρόταση αυτής της Επιτροπής, για αυτό το μηχανισμό, ε, το Συμβούλιο εξακολουθεί τις εργασίες του, συνεχίζει τις εργασίες του σε τεχνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Και εγώ που έλεγα να σας ζητήσω να είστε σύντομος. Πολύ χαίρομαι που το έκανα. Μπορούν να βγάλουν τα συμπεράσματά τους ε, τα μέλη της Επιτροπής. Είναι μεγάλος ο κατάλογος. Και τώρα θα ήθελα να ακούσουμε τον ε, jean Σέμπρι Τι γίνεται για την, με την Ελλάδα και την Ιταλία. Πριν πάρει το λόγο, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να μας πούν τώρα κατά πόσον θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση αυτή. Αν θέλετε λοιπόν να σηκώσετε το χέρι σας τώρα, ξέρω ότι σας προβληματίζω λίγο, αλλά για να ξέρουμε πόση ώρα έχουμε, γιατί σε πολλές περιπτώσεις ε, μπαίνουν με τελευταία στιγμή κάποιοι και έχουμε προβλήματα. Άρα, συνάδελφοι, θα κλείσω τον κατάλογο, γιατί είναι και πάρα πολύ μακρύς. Σας παρακαλώ, λοιπόν, μην ζητήσει κανείς άλλους ε, το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτέ, σα ευχαριστώ που μα καλέσατε στη συζήτηση αυτή για να σα ενημερώσουμε για τη δουλειά μα, για την Ιταλία και για την Ελλάδα, για την μετεγκατάσταση, όπου συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με του ενδιαφερόμενου φορεί για να πετύχει το πρόγραμμα αυτό από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστηρίξη για το Άσυλο. Να δούμε λοιπόν ποιοι είναι επιλέξιμοι για επανεγκατάσταση στην παρούσα φάση, γιατί αυτό εξαρτάται και από τα κριτήρια του 75% για την διεθνή προστασία. Έχουμε Σύρους από την Ερυθρέα, άτομα από το Ιράκ, από την Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, άτομα λοιπόν τα οποία είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα αυτό και άτομα τα οποία είναι χωρίς κράτος, αλλά κατοικούν ή διατείνονται ότι κατοικούν σε μία από τις χώρες αυτές. Κάποια γεγονότα τώρα, κάποια στοιχεία. 34.953 άτομα θα επανακατασταθούν από την Ιταλία, 63.302 από την Ελλάδα, 54.000 έχουν τοποθετηθεί σε ομάδα για μετέπειτα μεταγκατάσταση και από ό,τι ξέρετε η Σουηδία ήδη έχει ζητήσει να συμμετάσχει στο έργο αυτό. Η εφαρμογή θα πάρει δύο χρόνια. Να σας διαβεβαιώσω ότι οι δικαιούχοι που μεταγκαταστώνται έχουν όλοι καταχωριστεί και τους έχουμε πάρει και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Τι κάνουμε τώρα λοιπόν, ποιος είναι ο ρόλος μας. Να σας δείξω κάποιες εικόνες. Καταρχάς, παρέχουμε πληροφορίες με το που κατεβαίνουν από τα καραβιά. Σε άτομα από τα οποία ενδεχομένως να είναι επιλέξιμα. Τους εξηγούμε τα έργα με μετεγκατάστασης, τους εξηγούμε και τις διαδικασίες παροχής ασύλου. Αυτό βλέπετε στην πρώτη ε, φωτογραφία, μια ομάδα στη Λέσβο, στην Ελλάδα. Τέτοιου είδους δουλειά. Ύστερα, η καταχώρηση. Και πάλι λοιπόν υποστηρίζουμε στη διαδικασία καταχώρησης τα κράτη-μέλη, τον ετούντον άσυλο. Ύστερα έχουμε την εργασία συντηριάσματος, αν θέλετε όπου τα άτομα τα οποία είναι επιλέξιμα τα ταιριάζουμε στα κράτη-μέλη, στα οποία θεωρούμε ότι μπορούν να εγκατασταθούν και μετά έχουμε τα θέματα αναχώρησης και άφηξης. Στην παρούσα φάση έχουμε άτομα τα οποία έχουν εγκατασταθεί σε μία σειρά περιοχών, στην Ιταλία, στα hot spots, ε, στη Λαμπεντούζα, που παρέχουμε πληροφορίες, Βίλα Σικάνια, όπου γίνεται κυρίως καταχώρηση, στο Μιλάνο, στη Ρώμη και στην Κατάνια. Θα σας εξηγήσω γιατί Μιλάνο και Ρώμη πιο μετά. Στην Ελλάδα. Έχουμε άτομα στη Λέσβο και συντόμως στην Αθήνα στο URTF. Βλέπετε λοιπόν στο χάρτη ότι τα hot spots που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι στη Λέσβο και τα υπόλοιπα που προγραμματίζονται Χίο, Σάμος, Λέρος και Κος δεν έχουν ακόμα ανοίξει. Στην Ιταλία, Λαμπεντούζα, την οποία και μόλις ανέφερα, και τα άλλα hot spots, Τράπανη, Πότσα, Λαγκούστα, Ταράντο, ακόμα είναι στη φάση προγραμματισμού και σχεδιασμού. «175 εμπειρογνώμονες». 174 ζητήσαμε μάλλον. Μέχρι τώρα μας έχουν δώσει 176. 30 άτομα έχουμε αναπτυγμένα στην παρούσα φάση και μιας και δεν έχουν ανοίξει ακόμα όλα τα hotspots, βλέπουμε ότι έχουμε αναπτύξει επαρκές ε, προσωπικό στην παρούσα φάση. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι πολύ διαφορετική πραγματικότητα στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό να υπάρχει ευελιξία στην προσέγγιση λοιπόν. Αυτά είναι αυτά που σας έλεγα και προηγουμένως. Οι εμπειρογνώμονες τους οποίους έχουμε λάβει. Προκλήσεις. Γιατί είμαστε τόσο αργοί. Γιατί είμαστε τόσο αργοί, γιατί πήρε τόσο καιρό αυτή η διαδικασία. Δεν έχουν ακόμα καταστεί λειτουργικά όλα τα hot spots, όπως σας είπα. Κάποια εξ αυτών δεν έχουν ακόμα ανοίξει. Και προφανώς έχουμε και θέματα επιμελητίας, βασικά πράγματα, όπως για παράδειγμα ε, μια γραμμή IT σε ένα νησί. Αυτά παίρνουν χρόνο. Ε, έλλειψη γραφείων επίσης. Επίσης υπάρχει και μία απροθυμία, πρέπει να το πούμε και αυτό, από τα άτομα τα οποία προορίζονται προς μετεγκατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική η διάσταση των πληροφοριών. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τους πληροφορήσουμε σωστά, να τους ενημερώσουμε σωστά και να, το, ξέρουν ότι αυτή η διαδικασία είναι σωστή και αυτή που πρέπει να ακολουθηθεί. Τι προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε για να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις. Καταρχάς επικεντρωνόμαστε στις ε, ροές που είναι και εκτός των hot spots και γι' αυτό έχουμε άτομα στο Μιλάνο. Προσπαθούμε να βρούμε άτομα λοιπόν τα οποία ενδεχομένως να έχουν μπει από το ποτσάλο που δεν αποτελεί hot spot στην παρούσα φάση και τώρα βρίσκονται στην Ιταλία και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις ομάδες αυτές και να τις ε, κάνουμε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Επίσης αναπτύσσουμε κινητά γραφεία σε όλα τα νησιά στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να εργαστούμε στις τοποθεσίες αυτές μέσα σε λίγες ημέρες. Έχουμε επίσης κινητές ομάδες όπως σας είπα, ποτέ δεν ξέρουμε πού θα καταφτάσει η βάρκα και αυτό πιστεύαμε ότι καλό ήταν να υπάρχουν κινητές ομάδες. Μια ομάδα στη Ρώμη, για παράδειγμα, η οποία μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα εφόσον χρειαστεί. Η ευελιξία πάντα αποτελεί το σημείο κλειδί σε οποιαδήποτε προσέγγιση. Βλέπετε λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία τώρα των ατόμων που έχουν μετεγκατασταθεί ως τώρα και βλέπετε, σας εξήγησα και στο παρελθόν, προηγουμένως ότι τα αριθμητικά στοιχεία δεν είναι τόσο υψηλά. Έχουμε όμως και κάποιες ιστορίες ε, επιτυχής. Μία οικογένεια, την οποία την παρακολουθήσαμε από την αρχή μέχρι το τέλος, καταχωρίστηκε στη Λέσβο, στην Ελλάδα, και η όλη διαδικασία από την καταχώρηση μέχρι το νέο του σπίτι στο Λουξεμβούργο και τα παιδιά τους να πηγαίνουν και σχολείο ήδη στο Λουξεμβούργο πήρε δύο εβδομάδες. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι το πρόγραμμα αυτό μπορεί να στεφτεί με επιτυχία αν συνεργαστούν ε, με λέγγυο τρόπο όλα τα μέρη ασφαλώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ας περάσουμε απευθείας ε, στα μέλη. Ξεκινούμε από τους κοιόδης. Τζρόμι Λέναρτς, από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Κέρκοφ για την εισαγωγή μα, που μας έδωσε αλλά και την ΕΑΖΟ και το Συμβούλιο ε, για τη συμβολή του. Ε, είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτή την πρόταση, αλλά ήδη έχουμε κάνει πολλά στο Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τις δύο αποφάσεις του Συμβουλίου για τις 40.000 και 120.000 πρόσφυγες που θα μετακατασταθούν από Ελλάδα και Ιταλία. Δεν ξεκινάμε λοιπόν από το μηδέν και ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι εμού περιλαμβανομένου, απογοητευτήκαμε από τι αποφάσει και το γεγονό ότι το Κοινοβούλιο δεν ενεπλάκει επισήμως με στη δικασία συναπόφασης και επιμείναμε πολύ στη γνωμοδότηση που δώσαμε ότι οποιοδήποτε μόνιμο ε, μηχανισμός θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και το Κοινοβούλιο ω ε, συνομοθέτη. Αυτό μας δίνει μεγάλες δυνατότητες να βοηθήσουμε, να σχεδιάσουμε αυτό το νέο μηχανισμό στην Ευρώπη, αλλά αυτό ενέχει και μεγάλες ευθύνες για μας. Ευθύνες να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόταση με γρήγορο, ενωμένο και αποδοτικό τρόπο. Προσβλέπω λοιπόν σε περισσότερες συνομιλίες με τους αδέλφους, Συμφωνώ με τον, με τον ότι μπορεί να λειτουργήσει αυτό το σύστημα μόνο αν οι υπόλοιπε πτυχέ τη ολιστική προσέγγιση στην ε, μετανάστευση αρχίζουν να υλοποιούνται. Και αυτό ισχύει και για την επιστροφή πολιτική, εξωτερική προστασία των συνόρων, μάλλον προστασία των εξωτερικών συνόρων, τα hot spots. Μετά την σημερινή παρουσίαση δεν είμαι πιο αισιόδοξο προ αυτά τα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά την και την πρόταση, Νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν έχουμε προσδιορίσει πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όρους ε, και σημεία αναφοράς. Αυτή τη στιγμή στην πρόταση τα benchmarks αυτά δεν υπάρχουν. Η πρόταση μας λέει τι θα υπολογίσουν, αλλά όχι τι ακριβώς είναι στα μία ροή, για παράδειγμα. Και πολύ φοβάμαι ότι αν συνεχίσουμε σε αυτή την οδό, θα έχουμε ένα αντίστοιχο ε, κείμενο με αυτό των προσωρινών μηχανισμών. Ναι, χαιρόμαστε που κάτι υιοθετείτε, αλλά τελικά τι θα, τι εφαρμοστεί. Και δύο σύντομα ερωτήματα μου επιτρέπετε προς την ε, Κομισιόν. Εξετάζουμε αυτή την ε, πρόταση νομοθεσίας, ενώ ταυτόχρονα η Κομισιόν έχει ανακοινώσει μία ενδελεχή αξιολόγηση του κανονισμού του Δουβλίνου που θα οδηγήσει σε αναθεώρηση. Επομένω, ε, πώς θα ε, επηρεάσει αυτή την ε, αναθεώρηση του συνόλου της νομοθεσίας αυτή η πρόταση. Δεύτερον, η υιοθέτηση των μόνιμων μηχανισμών κρίσης δεν αποτρέπει στο Συμβούλιο να υιοθετεί και έκτακτους μηχανισμούς αντιμετώπισης κρίσεων υπό το άρθρο 73, αν ακούσουμε καλά γιατί να αξιοποιήσει το Συμβούλιο τον μόνιμο μηχανισμό αντί των άλλων αποφάσεων κρίσης σε ό,τι αφορά τη μετακατάσταση. Μάριον Ντάλι, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ, θα μιλήσω στη μητρική μου. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κέρκοβ για τις παρατηρήσεις του. Βλέπουμε πώς μπορούμε να κινηθούμε από εδώ και πέρα. Ως ε, S&D θεωρούμε ότι αυτός ο μυθικός φάκελος είναι εξαιρετικά σημαντικός. στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μετανάστευσης και Ασύλου. Στη σημερινή παρουσίαση βλέπουμε ότι, και απο, απορρέει μάλλον αυτή την παρουσίαση, ότι χρειαζόμαστε πολύ συγκεκριμένε δράσεις και όλα αυτά τα σχέδια να γίνουν πραγματικότητα. Δεν έχει νόημα να έχουμε συμφωνία επί της μετακατάσταση αν όλα αυτά μείνουν ε, στα λόγια και δεν ε, αλλάξει κάτι στην πράξη. 150 άτομα έχουν μετακατασταθεί βλέπουμε, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πράγματι, έχουμε αυξημένη εισρωή ε, μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη και δεν έχει νόημα να κρύβουμε το πρόβλημα κατά το χαλί και να αφήνουμε ε, μόνες ε, τις χώρες που ε, πλήττονται περισσότερο από αυτό το φαινόμενο. Τα όσα είπε ο εκπρόσωπος του ΕΑΣΟ. Βλέπετε πόσο σημαντικός είναι και ο ρόλος του, των κρατομελών εδώ και πόσο σημαντική είναι η συμβολή τους. Τώρα, κάποια στοιχεία που για μένα είναι σημαντικά. Πρώτον, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν θα μειωθεί δραστικά ο αριθμό των ε, προσφύγων. Γι' αυτό πρέπει να δείξουμε έμπρακτη αλληλεγγύη. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό ο φάκελο για να εφαρμοστεί στην πράξη η αρχή τη αλληλεγγύη. Και θα πρέπει αυτό να συμπεριληφθεί και σε έναν, ε, μια νομοθετική διάταξη που θα μπορεί αυτομάτως να ενεργοποιείται. Βλέπουμε τη σημασία του κανονισμού του Δοβλίνου, αλλά και ότι κάποιες διατάξεις ε, ε, πλήττουν την νομοθεσία στην Ευρώπη, γιατί βλέπουμε στην ουσία ότι το Δουβλίνο δεν λειτουργεί καλά. Και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε μας δείχνουν ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να απομακρυνθούμε από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί είναι ιδιαίτερα ασαφής. Πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι για παράδειγμα, πώς ορίζεται η κρίση. Πολύ ασαφής ο ορισμός. Άλλα στοιχεία που θα πρέπει να εξετάσουμε. Ε, επιθυμώ την συνέχιση της συνεργασίας με τον εισηγητή και τους σκιώδεις στις επόμενες εβδομάδες και ελπίζω να καταλήξουμε σε, μία, σε ένα αποτέλεσμα που θα κάνει διαφορά. Ευχαριστώ. Από πλευρά Άλντε, η Σεσίλια Βίξτρομ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. εντυπωσιακά τα στοιχεία και οι εικόνες που μας παρουσιάσατε. Τα success story που αναφέρατε για την μετακατάσταση των 130 ατόμων από την Ελλάδα. Εγώ ήμουν στην Ελλάδα εκείνη τη στιγμή όταν έγινε η μετακατάσταση και ήταν πραγματικά μια επιτυχία. Όμως 131 άτομα δεν μας στάνει αυτό. Την επόμενη μέρα όμως από τους ίδιους μετα μετεγκατεστημένους ε, διαδόθηκε αυτή η είδηση προς άλλους ε, που έρχονται εκείνη τη στιγμή στην Ελλάδα ότι τι ωραία που είμαστε στο Λουξεμβούργο και όλοι ξαφνικά θέλουν να πάνε στο Λουξεμβούργο. Όμως πρέπει να δούμε τι σημαίνει για παράδειγμα με τον Υπουργό Εξωτερικών ε, της Εστονίας, ε, με τον οποίο συναντήθηκα ε, στις ΗΠΑ. Είπαν ότι προσπαθούσαν να βρουν άτομα που ήθελαν να μετεγκατασταθούν, όμως δυστυχώς η παραπληροφόρηση είχε δράσει πολύ νωρίτερα. Επομένως, αυτά τα πρόσωπα είναι ευάλωτα, προσπαθούν να ξεφύγουν από εμπόλεμες ζώνες, από διώξεις και φοβούνται τόσο πολύ να ξαναβρεθούν στην ίδια κατάσταση και έτσι διστάζουν ακόμα και να μπουν σε ένα αεροπλάνο και να μετακατασταθούν. Τι μπορεί να γίνει, θα ήθελα να μου πείτε, εάν υπάρχουν ομάδες ψυχολογικής υποστήριξης. Γιατί είναι σημαντικό να σπάσουμε αυτό τον κύκλο της παραπληροφόρησης που δέχονται αυτά τα άτομα και να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη, ιδίω ό,τι αφορά αυτά τα ευάλωτα άτομα. Γιατί γενικά θέλουμε να μετακαταστήσουμε 160.000 άτομα. Με αυτή την ταχύτητα θα μας πάρει περίπου 75 χρόνια από τώρα. Εκτός και αν γίνει κάτι, αν υπάρξει μια δραστική αλλαγή. Θα ήθελα να μου, να πείτε λοιπόν ποια μέτρα προβλέπονται για τη μετακατάσταση όχι μόνο ενός 15-30 ε, ατόμων, αλλά μια σωρία ατόμων. Δεύτερον, η Σουηδία πραγματικά έχει κατακλειστεί αυτή τη στιγμή από πρόσφυγες. Πριν από μερικές εβδομάδες δεν υπήρχαν άλλα στρώματα στη χώρα. Δεν μπορούσαμε καν να αγοράσουμε στρώματα. Έχουμε βάλει πρόσφυγες παντού, σχολεία, εργοστάσια, στο πάτωμα χωρίς καν ένα στρώμα. Ο κόσμος κοιμάται έξω, στο δρόμο και έχει έρθει ο χειμώνα. Με θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν πλέον στη Σουηδία. Κάνει κρύο λοιπόν, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, να τη χειριστούμε. Τι συμβαίνει λοιπόν αυτή τη στιγμή με την μετακατάσταση προσφύγων από τη Σουηδία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και προς συναδέλφους που δεν το γνωρίζουν, μιλούμε για δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες κάθε εβδομάδα. Τώρα έχουν λίγο πέσει ε, τα νούμερα μετά από τα δρακόντια μέτρα που ε, πήρε η κυβέρνηση, αλλά η κατάσταση είναι αφόρητη γενικά. Και είχαμε ζητήσει τη μετακατάσταση πριν από ένα μήνα. Τι έχει συμβεί από τότε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Από τους Πρασίνους, η Σκάκελερ έχει το λόγο. Σκιώδης. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω όσο είπαν οι συνάδελφοι ότι είναι καλό που υπάρχει η πρόταση αυτή όταν υπήρξε και ο κατεπήγον μηχανισμός ε, μέτρων. Είπαμε ότι θέλουμε ένα μόνιμο σύστημα ως συνομοθέτες για να υπάρχει και μια διάρκεια και συνέχεια. Αυτό φυσικά και σε σχέση με την μεταρρύθμιση του Δουβλίνου που ελπίζουμε ότι θα γίνει και υπάρχει και ένα θέμα του πώς θα τα συνδέσουμε αυτά. Άρα, θεωρώ ότι είναι καλό που υπάρχει αυτή η πρόταση για το μέσω αυτό το οποίο υποστηρίζουμε ως πράσινοι. Είναι καλό επίσης που θα ληφθεί η απόφαση από την Επιτροπή όταν υπάρχει κατεπήγον χαρακτήρας. Δεν λέω να μην υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές. Οδηγία προσωρινή προστασία από τα κρατημέλια αλλά υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπορεί να ανακηρύξει κατάσταση κατεπίγουσας ανάγκης. Και νομίζω ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε. Το όριο του 75% είναι αυθαίρετο, πιστεύω. 70% θα ήθελα. αν θεωρήσουμε ότι έχουμε αντλήσει και τα διδάγματα από το παρελθόν. Οι Αφγανοί, μια πολύ σημαντική ομάδα μεταναστών, είναι στο 74% εξαιρούνται και αυτό μας οδηγεί σε πάρα πολλούς ε, Αφγανούς στην Ελλάδα που δεν έχουν δυνατότητα μετεγκατάστασης. Να δούμε λοιπόν την πράξη, στην πράξη τι γίνεται να δούμε λοιπόν μεγάλες ομάδες προσφύγων που έχουν καθεστώς προσφύγων και θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τον καταπήγον μηχανισμό μετεγκατάστασης, θα πρέπει να μην ζητάμε στους ε, πρόσφυγες να ζητούν άσυλο στην πρώτη χώρα άφηξης, γιατί αυτό οδηγεί σε επιπλέον ε, γραφειοκρατικό άχθος για την Ιταλία, για την Ελλάδα, προτού γίνει η μετεγκατάσταση αυτή η διαδικασία χορήγηση ασύλου θα γίνει έτσι κι αλλιώ στη χώρα άφηξη μετά τη μεταγκατάσταση, αλλά νομίζω ότι έχει νόημα να μην χρειάζεται να κάνουν όλε τι διαδικασίε και τι διεκπαιρεώσει στην Ελλάδα και στην Ιταλία για να υπάρχουν λιγότερα γραφειοκρατικά βήματα. Και νομίζω ότι προκαλεί και μία δυσπιστία ότι μπορεί να μην θέλουν να ζητήσουν υλό τα άτομα αυτά γιατί ξέρουν πόσο υπερφορτωμένες είναι αυτές οι χώρες και ενδεχομένως λοιπόν να μην έχουν εμπιστοσύνη σε όλο το σύστημα και συμφωνώ ότι η ενημέρωση αποτελεί ένα βασικό ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να υπάρχουν από πλευρά τη υπηρεσία επαρκή άτομα επιτόπου και στα hot spots. Γιατί το θέμα είναι να υπάρξει επιτάχυνση της διαδικασίας μέσω των hot spots. Αλλά από την άλλη χρειάζεται και χρόνος να μιλήσει κανείς στους πρόσφυγες, να τους εξηγήσει τι ακριβώς είναι η μετακατάσταση, ποια είναι τα ωφέλη και για τις χώρες. Γιατί πού να ξέρει ίσως κάποιος ε, πώς είναι το Λουξεμβούργο. Όλα αυτά λοιπόν παίρνουν χρόνο. Συμφωνώ επίσης ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τις δευτερεύουσες μετακινήσεις. Αυτό είναι σημαντικό και το έχουμε πει και στον καταπήγον μηχανισμό, αλλά νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ακολουθεί τη σωστή προσέγγιση. Λέτε ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, οι κινήσεις του μεταναστών. αλλά αυτό δεν επηρεάζει απαραίτητα τις δευτερεύουσες ε, μετακινήσεις. Αν λάβουμε υπόψη τον κοινωνικό περίγυρο, τις οικογένειες των προσφύγων, τότε, τότε και μόνο μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα συνενέσουν για την ε, μετακαταστασή τους και αυτό νομίζω ότι αποτρέπει τις δευτερεύουσες μετακινήσεις και δημιουργεί και λιγότερες ε, λιγότερο δημοκρατικό ε, γραφειοκρατικό άκθος και έτσι λοιπόν αυτό ενδεχομένως ε, προκαλεί και προβλήματα σε ό,τι αφορά την οδηγία για τα δικαιώματα των ε, προσφύγων. Νομίζω λοιπόν ότι καλό είναι να υπάρχει πρόληψη της δευτερεύουσα ε, μετακίνηση. Επίσης, να δούμε και την ε, περίοδο αναμονής. Γιατί αν πούμε σε έναν μετανάστη που μόλις έχει φτάσει στη Λέσβο ότι κοιτάξτε, έχουμε αυτό το φανταστικό πρόγραμμα, αλλά θα μα πάρει δύο μήνες μέχρι να σου βρούμε που θα πας. Και δεν ξέρουμε αυτού τους δύο μήνες που θα πας και τι θα κάνεις και πώς θα ζήσεις με τι χρήματα θα ζήσεις. Ε, πολλοί κόσμος ενδεχομένω να αρνηθεί. Άρα θα πρέπει αυτή η περίοδος αναμονής να είναι πιο σύντομη, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να λάβει μια γρήγορη απάντηση. Και μια ερώτηση προς την Επιτροπή. Ναι, γιατί δεν είμαι ακόμα 100% βέβαιη. Τα κράτη-μέλη πληρώνουν κρίματα για να απαλλαχθούν από την υποχρέωση αυτή για ένα έτος. Έχετε καθόλου εμπειρία από αυτό το σύστημα. Δηλαδή, ποσοστό ΕΠ. Πιστεύετε πραγματικά ότι αυτό θα οθήσει τα κράτη-μέλη στο να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Κοιτάξτε, δεν θέλω να σας πιέζω, αλλά είναι μεγάλος ο κατάλογος των ομιλητών και έχουμε και άλλες δύο μεγάλες εκθέσεις. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό βέβαια. Αλλά σας παρακαλώ να έχετε υπόψη σας και το ρολόι. Η FDD Λόρα Φεράρα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα χαιρόμουν να ξεκινήσω από αυτό που άκουσα από πλευράς ε, δόκτωρα Σκέμπρη στο τέλος ε, ε, από τη στιγμή που θα υπάρχει αλληλεγγύη θα λειτουργήσουν τα πάντα. Αν θέλουμε να βασιστούμε στους αριθμούς, λείπει αυτό το πνεύμα σήμερα. Μόνο 14 κράτη-μέλη είπαν ότι δίνουν θέσεις ε, για την μετεγκατάσταση σε 160.000, δηλαδή είναι πολύ λίγα και 129 σε δυνατότητα 39.600 30 σε 66.000 τόσους. Όπως σας είπα, όπως είπε και ο Γιούνκερ με το 2100 ούτε τότε δεν θα έχουμε τελειώσει ακόμα αυτούς 160.000. Αυτό για τα κατεπήγοντα μέτρα. Μιλάμε για κατεπήγοντα έτσι. Καταλαβαίνετε τι θα συμβεί με τον όλο μηχανισμό τον υποχρεωτικό. Να πω κάτι σύντομα ότι συμμερίζομαι μαζί σας τη χθεσινή εμπειρία και ήταν ο δέκτωρ Κέμπρι Πάρν και στην ετήσια συνάντηση Κόζακ και με αρκετούς βουλευτές από διάφορα κράτη-μέλη συνομιλήσαμε για αυτή τη μεταναστευτική ροή. Και υπήρχε μια άρνηση, μια αναχέτηση, ένα εμπόδιο σαφές, συγκεκριμένο, σκληρό από διάφορα ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένας κατάλληλος μηχανισμός ε, για τις υποχρεωτικές ποσοστώσεις ας πούμε και κράδεντας ε, την αρχή της επικουρικότητας, ε, την κυριαρχία των μενομοκρατών μελών. Δεν μπορεί να επιβάλλει δηλαδή το η Ευρώπη σε ένα κράτος μέλος σε αυτή την μετεγκαταστήτη χώρα του Αυτό κατά της συνεργασίας και της αλληλεγγύης που εμφανίζεται στο άρθρο 80 και στην κοινή πολιτική για το άσυλο στο 78 άρθρο της συνθήκης. Θα ήθελα να βασιστώ Μάλλον, αν θέλουμε να βασιστούμε στα σημερινά στοιχεία και την αντιμετώπιση τη σημερινή, η μελλοντική προοπτική δεν είναι και τόσο ρόδινη. Αυτά λοιπόν. Σύμφωνα συμφωνώ με την κυρία Σκέλλερ, τη συνάδελφο, σχετικά με το ποσοστό του 75% καλύτερο θα ήταν να το μειώσουμε ακόμη περισσότερο, τουλάχιστον το 70%, ώστε να δίνουμε δυνατότητα και σε άλλους, άλλους πρόσφυγες από άλλες τρίτες χώρες να μπορούν και αυτοί να επανεγκατασταθούν όπως ε, αναφερθήκαμε σε Αφγανού πολύ σωστά. Και ακόμα ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη διαφόρων δυνατοτήτων ε, με δευτερεύουσες κινήσεις, περαιτέρω ροές ε, μεταναστευτικές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Λάουρα. Ευχαριστώ που ήσουν και σύντομη. Το εκτιμώ ιδιαίτερω. Ο κύριος Ντουπχέ, παρακαλώ. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Στα γρήγορα, πολύ γρήγορα, φεντεραλιστής Ευρωπαίος είμαι, γι' αυτό με την ελεγγύη απέναντι σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα αυτό είναι και επιλογή και υποχρέωση, αλλά αντιμετωπίζω ένα κάποιο πρόβλημα με το ολοχρόνο διάγραμμα σχετικά με τις προτάσεις αυτές. Ταιριάζει να ξεκινάμε πάνω σε ένα μηχανισμό μόνιμο από τη στιγμή που βλέπουμε απογοητευτικά αποτελέσματα ακριβώς για 160.000 την εγκατάστασή που είπαμε με τα μπουρλα κλπ. ότι ήταν μεγάλη απόδειξη αλληλεγγύης. Εδώ για ορισμένα κρατη κράτη-μέλη για την κοινή γνώμη υπάρχουν και πολιτικές θεωρήσεις που θα πρέπει να μπαίνουν στο παιχνίδι και ορισμένες στιγμές θα πάνε καλά τα πράγματα, άλλες στιγμές όχι. Θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, τι δυνατότητες υπάρχουν μέσω του χρονοδιαγράμματος που είναι πολύ σημαντικό και επίσης κάτι άλλο. Αυτό που το εξετάζουν έτσι η κοινή γνώμη στα διάφορα κράτη, θα έχουμε και περιφερειακές εκλογές. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε ακριβώς πριν να κεντρωθούμε σε ένα μηχανισμό και μόνο. Είχε δίκιο ε, ε, αυτό, ε, αυτό που ακούσαμε από πλευρά Ρακοφοπ. Εδώ δεν δέχονται οι πολίτες ένα μόνο στοιχείο της πολιτικής που θα εφαρμόσουμε, έτσι δύο πράγματα τα οποία και μου δημιουργούν εμπόδια με αυτό το μηχανισμό όπως προβλέπετε. Πρώτα απ' όλα μια εξαίρεση σχετικά με το Δοβλίνο. Εντάξει, υπέρ είμαι ιδιαίτερα, δεν γίνεται αλλιώ. Αλλά δύο ορ περιορισμοί υπάρχουν, το 40% και το 75%. Για ένα κράτο μέλο δεν θα μπορούμε να έχουμε παραπάνω από 40% που θα μπορούσαν έτσι να υποφεληθούν από αυτή την εγκατάσταση. Πού βασιστήκαμε για να το ρυθμίσουμε έτσι, ποιο κριτήριο, βάσει ποιου κριτηρίου. Και ακόμα, ξέρουμε πώς αντιμετωπίζουν παρόμοια κατάσταση που θα μπορούσαν να υποφεληθούν από αυτό το μηχανισμό μεταγκατάστασης σε σχέση τουλάχιστον με τους οικονομικούς μετανάστες που δεν μπορούν να υποφεληθούν. Θα γίνει μια εκτίμηση ακριβώς τι γίνεται, ποιο τι, πού κλπ. Σε ποιους θα αφορά. Κάτι όμως που με ενοχλεί περισσότερο είναι η δεύτερη εξαίρεση. Τα κράτη-μέλη που θα έλεγαν όχι, όχι δεν συμμετέχουν στο μηχανισμό μεταγκατάσταση Θα κάνουν. Θα πληρώσουν 0,02% σαν πρόστιμο. Κάθε κανονός το ξέρει ότι αν υπάρχει μια επιλογή ανάμεσα σε δύο πράγματα, ό,τι κοστίζει λιγότερο, αυτό θα επιλέξετε. Αν το κόστος 20.000 να δεχτείτε είναι υψηλότερο από ένα πρόστιμο, τότε θα διαλέξετε το πρόστιμο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες που δεν το θέλουν και ορισμένε χώρε τη κεντρική Ευρώπη. Ανάμεσα στο 0,002 σαν πρόστιμο πρέπει να πληρώσουμε και τα υπόλοιπα να πάρουμε 20-30 προσφύγες ε, γιατί ε, καθορίζονται τώρα τα κριτήρια. Θα κάνουν του υπολογισμού και θα πούνε «Α, το πρόστιμο». Και αν υπάρξουν πολλές κράτη που κάνουν παρόμοιε ε, ε, υπολογισμού, αυτού. τα κράτη που θα έπρεπε κανονικά να υποδεχτούν αυτού που θα έλεγαν όχι για τον κόσμο αυτό, τότε αυτός ο μηχανισμός ο απαλλακτικός της εξαίρεσης δεν είναι υγιής. Νομίζω ότι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει τρομερές διαφορές, σημαντικές διαφορές, μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολο ανάμεσα σε διάφορες ε, χώρες που θα δεχτούν να συμμετάσχουν σε αυτή την ελληνική και άλλες χώρες που δεν θα το δεχτούν. Βεβαίως πρέπει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα στην πράξη, γιατί μιλούμε για ανθρώπους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο μηχανισμός μεταγκατάστασης θα ισχύει μόνο για τις ε, υπηκότητες ε, που αναγνωρίζονται στο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, άνω των 90%. Όμως, οι επιμέρους υπηκότητες έχουν πολύ διαφορετικά ποσοστά αναγνώρισης από τα επιμέρου κρατη κράτη-μέλη. Επομένω, οι πιθανότητε ε, κάποιου να ε, λάβει το καθεστώς ή μάλλον ε, να τύχει διεθνού προστασίας εξαρτάται σε συγκεκριμένο βαθμό από την χώρα στην οποία θα τον στείλουμε. Θα ήθελα να μου πείτε με ποια βάση θα ληφθούν αυτές οι αποφάσεις και από ποιον. Από πλευρά σε τούτος άσυλο, κάποια κράτη-μέλη είναι πιο ελκυστικά από ό,τι άλλα για πολλούς λόγους. Από πλευρά και από σκοπιά κρατών μελών, ορισμένοι σε άσυλο είναι πιο αποδεκτοί ή επιθυμητοί από ό,τι άλλοι. Και αυτό είναι γεγονό. Αυτέ οι προτιμήσει πώ θα επηρεάσουν τη διαδικασία λήψη αποφάσεων και θα την επηρεάσουν και είναι ρεαλιστικό να θεωρεί κανείς ότι μπορούμε να αποτρέψουμε μια τέτοια ε, δευτερογενή μετακίνηση αυτών που έχουν μετακατασταθεί. Η κυρία Κέλλερ τώρα είπε ότι η προτίμηση των ετούντων άσφαλων θα πρέπει να λαμβάνεται ε, όσο γίνεται τώρα υπόψη, το οποίο από μόνο ότι είναι λογικό. Όμως, από την άλλη, Αυτές οι προσωπικές προτιμήσεις είναι αυτές που μας οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση, όπου μια χούφτα κρατών μελών ε, λαμβάνουν σχεδόν το σύνολο των αιτήσεων ασύλου, ενώ άλλες ε, χώρες δεν λαμβάνουν σχεδόν καμία. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιώταβα, παρακαλώ. Thank you, Ευχαριστώ, θα μιλήσω βουλγαρικά. Ευχαριστώ τα περισσότερα στοιχεία έχουν ήδη υποθεί. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημαντικά ζητήματα. Πριν το καλοκαίρι εγκρίναμε τον προσωρινό μηχανισμό μετεγκατάστασης. Ήταν πολύ δύσκολο να εγκριθεί από τα κρατημέλη, αλλά στην πράξη τι συμβαίνει δεν υλοποιείται. Αυτό βλέπουμε σήμερα. Δεν ε, είναι δυνατόν ε, να μα ικανοποιούν τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τη μετακατάσταση αυτή τη στιγμή. Το ερώτημά μου είναι από εδώ και πέρα πώ ε, θα κινηθούν τα πράγματα, πώς θα, ποια θα είναι η διασύνδεση μεταξύ των προσωρινών και μονίμων μηχανισμών. Γιατί πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει με αυτά τα 160.000 άτομα. Και νομίζω ότι έχει αλλάξει δραστικά η κατάσταση από το καλοκαίρι και μετά. Αναφερθήκαμε για τις μεγάλες εισρωές ε, στην Ελλάδα και στην Ιταλία, όμως αυτό συνεχίζεται και μάλιστα αυξάνεται. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το συσσωρευμένο ρυθμό ατόμων. Ε, το ίδιο ισχύει και για τα Δυτικά Βαλκάνια τι θα κάνουμε εκεί. Ε, έχει αρχίσει η ανέγερση φραχτών, το οποίο ε, διαμορφώνει και πολύ δύσκολη κατάσταση για την Ελλάδα. Και για, σε ό,τι αφορά τον ε, μόνιμο μηχανισμό, θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο δημιουργία hot spots στι χώρε προέλευση. Γιατί από ό,τι φαίνεται ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να τα χειριστεί αυτά τα ζητήματα μόνη τη. Θα ήθελα επίση να, μου πείτε ποιε αλλαγέ προβλέπονται στον κανονισμό του Δουβλίνου και πώς αυτές οι αλλαγές ε, θα ε, αλληλεπιδράσουν ε, με το μόνο μηχανισμό. Ευχαριστώ. Uh, thank you, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω καταρχάς ότι συμφωνώ με αυτά που είπε ο εισηγητής κ. Κέρκοπ. Πρέπει να διδαχτούμε και από τα πρετικά προγράμματα, ασφαλώς. Εκ παραλλήλου όμως, πρέπει να σας πω ότι έχω και κάποια ερωτηματικά. Που προκύπτουν από αυτά που μας είπε η ΑΣΟ Η απόφαση του 2015 2023 του Συμβουλίου αναφέρει ότι αν δεν υπάρξει καταχώρηση, ο τον άσυλος θα, άσυλο θα εξαιρεθεί από τη διαδικασία μετεγκατάστασης. Αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υποδεικνύουν κατά πόσον ένα ετών άσυλο έχει περάσει και έχει εισέλθει από hot spots. Αναφέρεται μόνο η ημερομηνία άφηξης και όχι ο τρόπος άφηξης. Η αντιπροσωπεία του ΕΝΒΑ λοιπόν είναι σαφής. Αν δεν υπάρχει καταχώρηση δεν υπάρχουν δικαιώματα γιατί δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει καλή θέληση από τους κρατικούς φορείς ε, σε αυτό το θέμα. Θα απαιτήσουμε λοιπόν ε, αυστηρά εχέγγυα για όσα, θα, όσα δικαιώματα προβλεφθούν στο νομοθέτημα. Για την έκθεση τώρα της ΕΑΖΟ. Πρέπει να σας πω ότι άκουσα με προσοχή και δύο θέματα με απασχολούν. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι απόλυτα λειτουργικά όλα αυτά hot spots ακόμα. Κατανοητό. Πρόκειται για μια τεράστια οργανωτική πρόκληση. Αλλά ακριβώς για αυτόν τον λόγο αναφέρεται ότι τα, οι ροές μεταγκατάστασης θα εστιαστούν στο εξωτερικό των hot spots. Και ω εκ τούτου δεν καταλαβαίνω ακριβώς. είμαι βέβαια τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Αν λέμε ότι οι ροέ μετεγκατάσταση ε, θα εστιαστούν εκτό των hot spots, υπονομεύουμε τον ίδιο το ρόλο και τη λειτουργία των hot spots. Άρα, να είμαι σαφή. Πραγματικά λέτε ότι ο κόσμος δεν θα πρέπει να περνάει από τα hot spots γιατί δεν μπορούμε να το οργανώσουμε αυτό ως εγχειρήμα. Θα πρέπει λοιπόν να το διευκρινίσουμε αυτό για να καταλάβουμε τι σημαίνει και το hotspots. Γιατί αν ο κόσμος μπορεί να παρακάμψει τα hotspots και να περάσει από άλλα κανάλια, θα χάσουμε οποιαδήποτε επισκόπηση και η διαδικασία μετακατάστασης θα είναι σχεδόν αδύνατο να εφαρμοστεί. Τέλος, να απαντήσω στη συνάδελφο Κέλλερ ότι συμφωνώ μαζί της. Αν ζούσαμε σε ένα τέλειο ιδανικό κόσμο, αλλά Δυστυχώς δεν ζούμε σε έναν ιδανικό κόσμο. Αν ακολουθούσαμε τη λογική σας, φυσικά θα θέλαμε να δώσουμε στον κόσμο το δικαίωμα της επιλογής. Αλλά αυτό θα σήμαινε ότι οι ίδιες οι χώρες που έχουν υπερβολικό φόρτο αυτή τη στιγμή, υπερβολική επιβάρυνση στην Βετική Ευρώπη, θα ήταν αυτές που εκ νέου θα επιβαρύνονται επιβαρύνονταν. Ίσως λοιπόν να χρειάζεται πιο πολύ ισορροπία, προκειμένου να υπάρχει κάποια αναλογία, προκειμένου βορρά, Νότος, Ανατολή και Δύση να μπορούν να επιμεριστούν τα φορτία αυτά κάπω πιο ισότιμα. Θα ήθελα να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστέ στην προσέγγιση μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σίπελ. Και πολύ ζητώ συγγνώμη από του συναδέλφου που ζητούν τώρα το λόγο. Το διευκρίνησα όμω εξ αρχή ότι είχα κλείσει τον κατάλογο των ομιλητών. Είμαστε πραγματικά σε απελπιστική κατάσταση σε ό,τι αφορά το χρόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γενικώ πώ υποστηρίζω την ιδέα να υπάρχει ένα μόνιμο μηχανισμό επανεγκατάσταση. Συμφωνώ επίση και με αυτά που είπε ο Τίμωθη Κύρκο, ότι φυσικά ένα μέτρο δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, δεν είναι πανάκια. Πρέπει να δούμε όλη την εικόνα, τη συνολική προσέγγιση, όπω διαμορφώνεται. Το πρόβλημα που έχω είναι ότι δεν βλέπω και ενδεχομένως η απάντηση του Συμβουλίου να αποτελεί μια υπόμνηση προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά δεν βλέπω τα κράτη-μέλη πραγματικά να δεσμεύονται σε αυτή την συνολική προσέγγιση. Άρα, 140 πρόσφυγες έχουμε εντάξει σε αυτό το πρόγραμμα μετακατάστασης και θυμάμαι ότι το Συμβούλιο ανακοίνωνε μετά το καλοκαίρι ότι μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου θα υπήρχε μετεγκατάσταση 40.000 προσφύγων. 140. Πολύ καλά. Αλλά πώς ελπίζουμε ότι με έναν άλλο μηχανισμό μετεγκατάστασης θα βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Άκουσα και κάπως μου ενόχλησε το γεγονός ότι ο Τίμωθη μιλάει για pull factors, για παράγοντες προσέλκυσης. Τι μιλάμε, τι λέμε, είναι πόλεμος έλξης, ο, ο πόλεμος της Συρία, ο πρόσφυγας από την Ερυθρέα έρχεται στη Γερμανία επειδή του δίνουν χρήματα. Εγώ θεωρώ ότι αυτοί οι παράγοντες έλξης είναι τα βασικά πρόβλημα της ε, προσφυγιάς. Δεν μας ενδιαφέρει όμως ο πόλεμος στη Συρία. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή μέχρι ότου άρχισαν να ξεχυλίζουν οι πρόσφυγες στα σύνορά μας για το Λίβανο και στην Ιορδανία. Δεν μας ένοιαζε που οι καταβλισμοί ήταν ε, υπερπλήρης μέχρι που άρχισαν να καταφθάνουν στην Ευρώπη. Δεν δίναμε καν χρήματα στην υπατή αρμοστία του, του ΟΗΕ για να έχουν τρόφιμα αυτοί οι άνθρωποι. Και τώρα μιλάμε για pull factors, για τέτοιους ε, παράγοντες έλξης. Τι να πω, γελίο και ευγενικά το λέω. Εγώ όταν πέφτω για ύπνο βλέπω εφιάλτες ότι θα συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη για τη μετεγκατάσταση την ημέρα που δεν θα έρχεται πλέον κανένας πρόσφυγας στην Ευρώπη γιατί κλείνουμε τα σύνορα, ορθώνουμε φράχτες, αναθέτουμε τέτοια καθήκοντα για τους πρόσφυγες στην Τουρκία και σε αφρικανικές χώρες και παρεπιπτόντως δεν δίνουμε και αρκετά χρήματα για να αντιμετωπιστούν οι αιτίε του προβλήματος της χώρας της Αφρικής. Όλα αυτά λοιπόν που κάνουμε εδώ είναι γελία. Και θέλω να αποσταλεί ένα σαφές μήνυμα από τα κρατημέλη ότι έχουν και κάτι άλλο να κάνουν προτίθεται να κάνουν και κάτι άλλο πέρα από το να ορθώνουν φράχτες και να δίνουν κονδύλια. Θέλω να αναλάβουν τις ευθύνε τους τα κράτη-μέλη, να πάρουν τους πρόσφυγες που τους αναλογούν, άτομα τα οποία τρέχουν και προσπαθούν να γλιτώσουν από την δίωξη και μετά να δούμε για νέα μέτρα. Ευχαριστώ. Τελικώς ε, μιλήσε και ο Κύρκος. Ευχαριστώ, μιλήσω ελληνικά. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Το ένα αναφέρεται στο 40% το οποίο είναι το maximum ε, σχετικά με τις δηλώσεις, με τις αιτήσει ασύλου των τελευταίων έξι μηνών. Επειδή η ροή των προσφύγων δεν είναι γραμμική, αλλά κάνει spikes, δηλαδή το χειμώνα είναι πάρα πολύ χαμηλά και ξαφνικά την άνοιξη πετάγεται ψηλά, αν δεν πάρουμε αυτό υπόψη θα έχουμε συγκέντρωση πάρα πολλών προσφύγων μέχρι να περάσουν οι μήνες και να έχουν και αυτοί δικαίωμα. Ένα δεύτερο, είναι η τρύπα που ανοίγει για να πληρώνουν τα κράτη αντί να δέχονται πρόσφυγες. Βεβαίως στην αιτιολογική έκθεση αναφέρει φυσικές καταστροφές και κάτι άλλο, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί μια πλημμύρα σε μια ε, περιοχή, σε μια επαρχία μπορεί να κάνει όλη τη χώρα να μην μπορεί να δεχτεί πρόσφυγες. Είναι μια τρύπα την οποία πρέπει να κλείσουμε. Και για την έκθεση της ΕΑΣΟ. Είπαμε για 150 οικογένειες. Τον Οκτώβριο μόνο μπήκανε 50.000 πρόσφυγες στη Μητυλίνη. Αυτή τη στιγμή όμως στη Μόρια, στο Καράτε Πέι, στην Αθήνα, δεν έχουμε 49.850 πρόσφυγες οι οποίοι περιμένουν με λαχτάρα να μετακινηθούν μέσω του μηχανισμού. Τους έχουμε στην ειδωμένη και προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτό που κάνετε με το να μην μπορείτε να οδηγήσετε, να μην μπορείτε να καλλιεργήσετε την εμπιστοσύνη των προσφύγων ώστε να μείνουν στους χώρους ώστε να μπορέσουν μετά να μετακινηθούν μέσα από το μηχανισμό, στην ουσία τορπιλίζει όλη την προσπάθεια αν έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι τα κράτη θα ανταποκριθούν τότε να πείτε ότι μόνο όσοι πρόσφυγες περάσουν και μείνουν στα hot spot μόνο αυτοί θα μπορέσουν να μετακινηθούν στις άλλες χώρες μόνο αυτοί θα γίνουν δεκτοί. αν όμως δεν το πιστεύετε αυτό τότε εσείς οι ίδιοι δίνετε στους πρόσφυγες αυτό που αυτή τη στιγμή κάνουν να μην έχουν καμία εμπιστοσύνη στην ελλάδα καμία εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή ένωση και να προσπαθούν με κάθε τρόπο εκτός μηχανισμού να μετακινηθούν προς όποια χώρα ελπίζουν είτε είναι το λουξεμβούργο σήμερα είτε η γερμανία χθε να φτάσουν. σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γερικό. Μια πρόταση. Ναι, κύριε Γκόμες. Κατανοώ ότι το ΕΑΖΟ δεν έχει τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, όμως δεδομένων των συνεπειών για χώρες όπως η δική μου, Πορτογαλία, που είπαν ότι είναι διατεθειμένες να υποδεχθούν πρόσφυγες και δεν έρχονται οι πρόσφυγες. Τι συμβαίνει. Uh, Ευχαριστώ, Άννα. Πριν δώσω το λόγο στους ε, ομιλητές. Ένα σύντομο σχόλιο, γιατί για τρίτη φορά σήμερα είχαμε πολύ υψηλό αριθμό ομιλητών. Ελέγχω τι συμβαίνει και στις άλλες επιτροπές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, γιατί έχουμε τα πιο σημαντικά ζητήματα που εξετάζουμε. Αν δείτε την μισή διάταξη σήμερα, τα πιο φλέγοντα συζητούμε σήμερα. Και αν δείτε και την ποιότητα των παρεμβάσεων, είναι εξαιρετικές. Ε, θίγονται όλα ε, τα εύλογα ρωτέ. Είναι τεράστια η κλίμακα και ο όγκος των ζητημάτων που εξετάζουμε, γι' αυτό και είναι δύσκολη η κατάστασή μα. Ε, ζητώ να ακολουθείτε του κανόνες πειθαρχία. Είναι τεράστιο ο κατάλογος ομιλητών. Ποτέ δεν έχω ξαναδεί τέτοια ένταση στι συζητήσει και στου διαλόγους. Κάποια στιγμή αρχίζουμε και διαγράφουμε σε μία της μέσης διάταξη γιατί ξεπερνούμε το χρονικό όριο. Αυτή τη στιγμή τα κρατάω τα ζητήματα, αλλά σίγουρα θα πρέπει να περιορίσω το χρόνο ομιλία στη συνέχεια. Θα τα συζητήσουμε με τη γραμματεία. Παράλληλα όμως υπάρχουν και πολλά νομοθετικά ζητήματα τα οποία δεν μπορούμε να ε, αναβάλουμε. Μια σύντομη προειδοποίηση. Γιατί είναι μεγάλο άγχος και για μένα, αν θέλετε, όταν προσπαθώ να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση σε τόσο σημαντικά ζητήματα. Σας ευχαριστώ όμως όλους. Ε, Στρέφουμε τώρα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπό τον χρονικό περιορισμό, μπορείτε να απαντήσετε σε αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα που σας ετέθησαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την, για την ε, πολύ ζωντανή συζήτηση. Αναφέρθηκαν πολλά στοιχεία. Πρώτον, ε, να συνοψίσω κάποια ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά την αργή έναρξη υλοποίηση ε, του μηχανισμού και, το, και την επιφυλακτικότητα των προσφύγων να συμμετάσχουν στο μηχανισμό κατά κατάσταση. Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ σαφέ από την απόφαση ότι δεν είναι προαιρετικός ο μηχανισμός. Και έτσι διαφέρει από το γιουρίμα, αυτό το καθεστώς ε, για τη Μάλτα, το οποίο δεν λειτουργήσε καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η επιφυλακτικότητα των προσφύγων θα πρέπει να υπερκεραστεί. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό και για την επιτυχή υλοποίηση ε, του μηχανισμού μετακατάστασης να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε αποτελεσματικά αυτή την απόφαση. Αυτό τι σημαίνει. Να λαμβάνονται τα την αποτυπώματα για να φτάσω στο ερώτημα της κυρίας Στέιβενς, κάθε παράτιμος μετανάστης ε, περνάει από τα hot spots. Κανένας να μην τα παρακάμπτει αυτά τα hot spots στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Η επιλογή θα πρέπει να γίνεται γρήγορα, όπως είπε η κυρία Κέλλερ, και θα πρέπει να γίνεται και υποχρεωτικά. Σε περίπτωση δευτερογενούς μετακίνησης θα πρέπει να επιστραφούν στο κράτος μέλους μετακατάστασης. Αυτό είναι θέμα συνέπειας και ήδη τώρα και υπό τους έκτακτους μηχανισμούς Υπάρχει αυτή η δυνατότητα με βάση την οδηγία ε, περί επιστροφών. Και ο δισταγμός για τη συμμετοχή ε, θα αντιμετωπιστεί και όταν υπάρχει και ενημέρωση προς τα κράτη-μέλη, προς τους πρόσφυγες μάλλον, από άλλους πρόσφυγες που έχουν μετακατασταθεί. Γιατί δεν... Κάποιοι λένε ότι δεν θέλουν να είμαι ο πρώτο υπήκο Ερυθρέα που θα πάει στην Εστονία. Αλλά αν ξέρει, για παράδειγμα, ότι υπάρχει ομογένεια σε άλλα κρατημέλη, θέλει να πάει προ τα εκεί. Λογικό είναι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτήν την ομογένεια σε όλα τα κρατημέλη. Και τότε θα είναι και ε, πιο δεκτικοί και οι πρόσφυγε. Αναφέρθηκε το ζήτημα τη πρώτη μετακατάσταση στο Λουξεμβούργο, που και εκεί υπήρχε δισταγμό λόγω έλλειψη ενημέρωση. Οι ε, κύριοι Λένερς και Ντεπχέ ε, με ρώτησαν ε, για τα κριτήρια, ότι δεν είναι αρκετά σαφή, πρέπει να είναι πιο λεπτομερή. Ας το θέσω ως εξής. Θεωρούμε ότι ένα περιθώριο ευελιξίας είναι απαραίτητο και είναι πολύ δύσκολο αν εξετάσουμε τις συζητήσεις και εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο, να καταλήξουμε σε έναν συγκεκριμένο κατάλογο πολύ συγκεκριμένων κριτηρίων και έτσι να έχουμε μια ομοιογενή κατάσταση για όλου. Η κατάσταση κρίσεων στα επιμέρου κρατημέλη μπορεί να διαφέρει επικοινοτρόπω, γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε επί όλων των σημείων. Να μην είναι δηλαδή η ίδια λύση για όλου. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ανέφερα τα κριτήρια που έχουμε συμπεριλάβει στην πρόταση. Βασίζονται πολύ στι καταστάσει κατά κεφαλήν και το μέγεθο ε, του κάθε κράτο μέλου όμως σίγουρα θα τα συζητήσουμε περαιτέρω και στους επόμενους τριμμένους διαλόγους. Η κυρία Βίξτρομ ρώτησε τι συμβαίνει με τι μετακαταστάσει από τη Σουηδία. Ο επίτροπο Αβραμόπουλο χθες ήταν στη Στοκχόλμη και συνομίλησε με τη Σουηδική κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε μία πρόταση που θα είναι έτοιμη κατά ψωθενότητα μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω πότε θα υιοθετηθεί από την Κομισιόν, αλλά έχουμε λάβει οδηγίες να εκπονήσουμε την πρόταση για να σημειωθεί η προόδος ε, σύντομα. Προς την κυρία Κέλλερ. «75%-70%» να το συζητήσουμε ποιο είναι το κατάλληλο ποσοστό. Νυχθημερών μπορούμε να το συζητούμε αν θέλετε, όμως ε, ήθελα μόνο να επισημάνω ότι προβλέπεται στην απόφαση στην πρόταση ότι το ποσοστό αναγνώρισης βασίζεται, ε, μάλλον προσδιορίζεται κάθε τρεις μήνες από τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat. Κάθε τρεις μήνες λοιπόν επικαιροποιείται η κατάσταση, μπορούν να συμπεριληφθούν και νέες ε, ηθαγένειες. Εμείς ζητήσαμε το 75% αρχικά για να δώσουμε μεγαλύτερα περιθώρια ασφάλειας και πιθανότητων για το κράτος μέλος ότι ο μετακατεστημένος είναι όντως ε, ετών άσυλο και μπορεί να του χορηγηθεί άσυλο. Μετά μπορούμε να το συζητήσουμε. Για την δευτερογενή μετακίνηση νομίζω και έχω την εντύπωση ότι όλοι συμφωνούμε. Είναι σημαντικό το θέμα πρέπει να το, το λύσουμε. Η Κομισιόν είναι διατεθειμένη να εξετάσει και άλλες προτάσεις εδώ. Απλώς να ξεκαθαρίσω ότι το προφίλ και τώρα λαμβάνεται υπόψη τα κράτη-μέλη μπορούν να δίνουν προφίλ σε αυτό το πλαίσιο. Μόνο ένας λόγος όμως είναι να απορρίψει κανείς το αίτημα είναι η πτυχή της ασφάλειας. Και κάποιος το ανέφερε γιατί αυτό είναι σημαντική ασφάλεια. Κυρία Κέιλερ, για τα οικονομικά ζητήματα δεν έχουμε ακόμα εμπειρία για το κατά πόσο τα κράτη-μέλη ε, αξιοποιούν αυτό το καταποκοπήν ποσό που τους χορηγείται. Είναι πολύ νωρίς, θα πρέπει να επανέλθουμε. Είπατε ότι μόνο 14 κράτη-μέλη συμμετέχουν. Να πω ότι οι έκτακτοι μηχανισμοί προβλέπουν δύο έτη για την υλοποίησή τους. Δεν το είχαμε προτείνει, αλλά προκύπτει από τις διαπραγματεύσεις από τα κράτη-μέλη, γιατί πολλά κράτη-μέλη που δεν έχουν καθόλου πρόσφυγες προς το παρόν είπαν ότι θέλουν και χρειάζονται χρόνο για να προετοιμάσουν τις υποδομές τους, να είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τους πρόσφυγες. Γι' αυτό δώσαμε αυτά τα δύο χρόνια. Και έτσι ε, δεν υπάρχει πρόβλημα που κάποια κράτη-μέλη λένε δεχόμαστε μηδέν προς το παρόν. Αυτό επικαιροποιείται κάθε τρεις μήνες. αλληλεπίδραση μεταξύ του έκτακτου και του μόνιμου μηχανισμού. Οι δύο έκτακτοι μηχανισμοί φτάνουν σε 160.000 όταν υιοθετηθεί ο μόνιμος μηχανισμός και οποιαδήποτε επιπλέον πρόταση θα βασιστεί στο 78.3. Και τελευταίο που ανέφερε ο κ. Ντεπχάη και άλλοι, το ανώτατο όριο του 40%, κατά πόσο είναι λογικό ή όχι. Σας εξήγησα μόλις γιατί προτείναμε αυτό το όριο. Γιατί αν δεν είχαμε όριο, αν κάποια στιγμή από μεγάλο κράτο μέλο κάναμε μετακαταστάσει, τελικά θα είχαμε πολύ υψηλού αριθμούς. Δεν θα μπορούσαν να το δεχθούν οι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα ήταν εφαρμόσιμα τα όρια. Γι' αυτό θέσαμε αυτό το κατόφλι, ούτω ώστε όπω και να έχει να υπάρχει ένα λογικό καθεστώς. Ελπίζω να απάντησα τα περισσότερα ερωτήματα. Ναι, πράγματι καλύψατε πάρα πολλά από τα ερωτήματα. Το εκτιμάμε ιδιαίτερο. Σας ευχαριστούμε. Τώρα στρέφουμε προς την Προεδρία. Ε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κάπως αργοπορημένα ήρθα, αλλά ήμουν σε μια άλλη συνεδρίαση με το Συμβούλιο. Άκουσα όμως να λέγονται πολλά ενδιαφέροντα πράγματα από όσους άκουσα τουλάχιστον για την επαναγκατάσταση γίνονται παράλληλα αυτές οι εργασίες με τον κατεπήγοντα μηχανισμό για την εφαρμογή. Είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή, δηλαδή αυτές τις δύο αποφάσεις από κοινού. Και μετά το μηχανισμό κρίσης, σε αυτό εργαζόμαστε πάνω και είναι οι πρώτες εργασίες. Τώρα ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις και η κατάσταση είναι η ίδια και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για τον κατεπήγοντα μηχανισμό τώρα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί. Χρειάζεται ένα κατάλληλο σχέδιο. Από τη στιγμή υπάρχουν όμως χιλιάδες που μας έρχονται. Μέχρι 20.000 τη μέρα στην Ελλάδα Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δύσκολο, πολύ δύσκολο είναι να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η έννοια του hot spot. Αλλά υπάρχει και το αντίθετο στην Ιταλία. Είναι και μέρες που δεν έρχεται κανείς. Τότε, αν τη στιγμή που δεν έχουμε κόσμο, πώς θα τον ε, μετακινήσουμε. Θα πρέπει να υποφελθούν τα κράτη-μέλη από το χειμώνα για να υπάρξει μια κατάλληλη οργάνωση που να μπορεί να λειτουργήσει στη συνέχεια όταν χρειαστεί. Να σου πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα πολλά που είπαν αρκετοί εδώ, ότι εδώ δοκιμάζεται η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Αυτό συμβαίνει. Το έχουν συντοπίσει τα κράτη-μέλη και ο ήταν σε συζητήσεις μπροστά που δεν ήταν και τόσο εύκολες ε, στο Συμβούλιο. Ορισμένοι όμως που τον λόγο τόνισαν ότι ήταν πρόκληση επίσης οι δευτερεύουσες κινήσεις, δροές κλπ. Νομίζω ότι αλλού είναι η πρόκληση πραγματική, να βρούμε αρκετό κόσμο για τον επανεγκαταστήσουμε και μετά να δούμε ποιες είναι οι δευτερεύουσες δροές μετακινήσεις. Αλλά αν τους υποδέχονται καλά, σωστά, σε ένα κράτος μέλος ας πούμε, τότε δεν υπάρχουν δευτερεύουσες δροές που να γίνουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η κυρία Βίξτρομ ε, είπε το θέμα της Σουηδίας. Εδώ αυτό που λέει αλλάζει τα δεδομένα. Δεν είναι πια μια χώρα άφηξης, είναι μια χώρα αλληλεγγύης σε σχέση με τις χώρες άφηξης, υποδοχής. Αυτό που ζητάει είναι πολύ σημαντικό. Έχετε δίκιο. Θα πρέπει κανείς να απαντήσει άμεσα σε αυτό της Σουηδίας και κάτι ακόμα είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με τις διπραγματεύσεις που εσείς και εμείς ε, διεξάγουμε για το μηχανισμό κρίσης που θα πρέπει να διατηρηθεί μετά, να διαρκέσει και θα πρέπει να τον ερτηθούμε αυτό για το τι γίνεται ε, με την ε, συμφωνία του Δουβλίνου και την μεταρρύθμιση μελλοντική του Δουβλίνου Παράλληλα λοιπόν συνεχίζουμε τις εργασίες μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να σας πω ότι την Παρασκευή οι Υπουργοί Αρμόδιοι για τη Μετανάστευση θα συζητήσουν πολιτικά για το μηχανισμό κρίσης. Χρειάζεται να ληφθούν εκεί υπόψη η πείρα που αποκτήθηκε σχετικά με τις ε, μετακινήσεις επαναγκαταστήσεις της επίγουσες. Είναι καλές, ε, αρνητικές. Αν όχι, τότε να δούμε τι άλλο θα πρέπει να βρεθεί και εμείς σκληρά εργαζόμαστε για να επιδείξουμε περισσότερη ελληνική, Αλλά δεν είναι και τόσο εύκολη αυτή η ελληνική. Δεν υπάρχει συμμετρία. Υπάρχουν οι γραμμέ, οι, τις πρώτες οι χώρες και μετά η, διαμετακόμισης και μετά η ε, τελική γεωγραφικού προορισμού. Καταλαβαίνετε ότι μπορεί να αλλάξει και η ροή, οι αφήξει ανάλογα με το σύστημα που εφαρμόζεται στα εξωτερικά ή στα εσωτερικά σύνορα. Ίσως αλλάξει η ροή αυτή από την μια στιγμή στην άλλη. Σε πολλά μέτωπα δίνουμε τη μάχη μας στο Συμβούλιο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό είχαμε και μια συνάντηση με την Τουρκία εδώ την Κυριακή, τα εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να λειτουργεί το σύστημα και στα εσωτερικά, στα εσωτερικά σύνορα μέσω του μηχανισμού επανεγκατάστασης. Αλλά επίσης οι υπουργοί θα μιλήσουν και για πολλά από τα θέματα που θέξατε εδώ, για τη συνεργασία με τους ίδιους πρόσφυγες. Αν υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης, ε, σίγουρα θα μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα ε, πρόσφυγες αυτοί, είναι κάτι το καινούριο όμως. Προέρχονται από μια ορισμένη κατάσταση και ορισμένες συνθήκες, με σειράξει κλπ. Αυτός ο κόσμος μπαίνει σε αεροπλάνο, καταλαβαίνετε την έλλειψη εμπιστοσύνη που υπάρχει, δυσπιστία. Πρέπει αυτό να το δουλέψουμε και χρειάζεται και μια δυνατότητα ε, υποδοχής ε, και στην άφηξη αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πότε πώς θα τους πείσουμε να παραμείνουν εκεί δύο μήνες μέχρι να λάβει ένα κράτος μία απόφαση. Θα πρέπει ταυτόχρονα και στο τελικό προορισμό μια κατάλληλη οργάνωση δυνατότητα υποδοχής. Ε, υπάρχουν χώρες που μπορούν να το κάνουν αυτό γρήγορα γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν μια συνειδητοποιήσει το θέμα αυτό περί υποδοχής αλλά είναι και κράτη που το κάνουν για πρώτη φορά αυτό για την επαναγκατάσταση και τέλος δίκιο έχετε όλα τα κράτη χωρίς καμία εξαίρεση θα πρέπει να συμμετάσχουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Αυτό κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ. Ένα τελευταίο να πω. Στην Ελλάδα και στην Ιταλία σημειώθηκε μια κάποια πρόοδος. Θέλω να το πω αυτό εδώ πέρα και τώρα να υποφεληθούμε από το χειμώνα, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε καλύτερα την επανεκκίνησή μας τον επόμενο άνοιξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνάδελφοι, για το δεύτερο θέμα, ο κύριος Ντεπρέ συμφώνησε ευγενικά να αναβληθεί το θέμα αυτό σε μια μελλοντική συνάντηση. Έχουμε άλλο ένα θέμα της κυρίας Γκίγιομ μέχρι τις 6.30. Εν συντομία, αν θα θέλετε. Ναι, να αναφέρω κάποια σημεία επιγραμματικά. Καταρχάς, ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε από την ε, βουλευτή Βίκστρομ για την πληροφορία. Πάρα πολύ, για τη συνημέρωση. Πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ. Και προφανώς δεν είναι προς το συμφέρον των διακινητών να ενημερώνουν τους ε, πρόσφυγες για την μετεγκατάσταση, γιατί προφανώς ε, τους τρώει το ψωμί. Άρα είναι δικός μας ρόλος να κάνουμε αυτή την ενημέρωση και ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σκληρά για μια στρατηγική επικοινωνία η οποία αναφέρεται και στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Τζάε. Άρα ναι, οι πληροφορίε και η ενημέρωση είναι σημείο κλειδί. Τι μπορεί να βελτιωθεί τώρα. Το ερώτημα του κυρίου Νταλή. Δεν είναι το θέμα να δακτυλοδείξουμε τον οποιοδήποτε. Κανέναν. Το θέμα είναι να δούμε τι θέματα χρειάζουν βελτίωση ή υποδοχή, πού θα μπουν αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να μεταγκατασταθούν και θα πρέπει να εκπληρώσουν τις υποσχέσεις τους τα κρατημέλα, τα κρατημέλη για τα hot spots και κατά πόσον ε, υπάρχει παράκαμψη των hot spots. Νομίζω ότι διευκρίνησε τα πράγματα η Προεδρία. Αυτά ήταν. Μάλιστα, θα μείνετε και μαζί μας, λέει ο Πρόεδρος, για το επόμενο σημείο. Γι' αυτό, λοιπόν, σας ε, πίεσα στην απάντηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζεράχ, που μπορούμε να αναβάλουμε το 28 και πάμε, λοιπόν, πάρα αυτά στο 29. Και πάλι ζητάω συγγνώμη από την κυρία Κιγιόμ που έχουμε μόνο 30 λεπτά στη διάθεσή μα. Α, Τίμωθη, Τίμωθη. Συγγνώμη. Πρόεδρε, πρόεδρε, κοιτάξτε. Νομίζω ότι είναι επισήμω απαραίτητο να πει κάποια καταληπτικά σχόλια ο εισηγητή. Καταληπτικά σχόλια, λοιπόν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τι παρεμβάσει σα και θα τα λάβω υπόψη όλα αυτά. Ναι, έχετε δίκιο, λέει ο πρόεδρο. Πολύ σα ευχαριστούμε. με στη διασύνη μου ξέχασα τον εισηγητή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τιμωθή. Συνάδελφοι, ας πάμε... Έλεγα συγγνώμη στην ε, κυρία Γεγιόμ που θα αναγκαστούμε να περιοριστούμε σε μισή ώρα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Η πρόταση για την κατάρτιση μιας, ε, ενός καταλόγου ασφαλών χωρών. Δεν θα κάνω εισαγωγικά σχόλια, θα δώσω κατευθείαν το λόγο στην κυρία Γιγιό και μετά στην ΕΑΣΟ και μετά στην πρεδια. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ πολύ σύντομα. Ε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αλλά μας είπε ο συνάδελφος εδώ ότι με αυτά που είπε η Επιτροπή θα τα έκανε όλα μαζί από κοινού. Άρα λοιπόν το ίδιο και εγώ θα ήθελα να τον ευχαριστήσω τον συνάδελφο που θα μας τα δώσει αυτά και μας τα σύντομα. Έτσι. Αυτή η εργασία για αυτόν τον ευρωπαϊκό κατάλογο για την ε, ε, σίγουρη προέλευση είναι λογική, λογικό υπακόλουθο της πολιτικής ασύλου και δείχνει επακριβώς ε, αυτή την έννοια στην οποία θα επανέλθω σε λίγο για να δω ακριβώς να διαπιστώσω ότι όλοι συμμερίζονται το ίδιο. Η σίγουρη προέλευση είναι εκεί που υπάρχει ένα δημοκρατικό σύστημα αξιόπιστο και σε ένα Εκεί δεν υπάρχουν διώξεις, ε, βασανιστήρια, βία, σύραξη κλπ και κάποιος που ζητάει άσυλο από μια σίγουρη χώρα ακριβώς θα πρέπει να είναι και αυτός ασφαλής και να μην χρειάζεται διεθνή προστασία. Εδώ ο στόχος είναι κατά της καταχρηστικής ε, χρήσης ακριβώς διαδικασιών στη διαδικασία αυτή ε, της ασύλου. Εδώ πρόκειται για κάτι το πολύ σημαντικό και για τα κράτη-μέλη, τα οποία αφορά υπόθεση, γιατί μπορούν να το εξετάσουν τάχιστα από τη στιγμή που από μια σίγουρη χώρα, στα σύνορα, είτε σε μια περιοχή τράνζιτ, αλλά είναι σημαντικό και για όποιον το ζητάει αυτό το άσυλο. Και επίσης να πω κάτι ότι ο ασφαλής χαρακτήρας μιας χώρας δεν είναι αυτός καθ' αυτός ε, εμπόδιο. Εξαρτάται από την κάθε αίτηση ξεχωριστά. Ο καθένας μπορεί να ζητήσει άσυλο και από ασφαλή προέλευση και κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά. Σε αυτή τη διαδικασία ακριβώς αναφέρεται μια εθνική, ένας εθνικός κατάλογος. Αυτό αναφέρεται μόνο. Παντός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πει τότε ότι πώς θα υπάρξει μια εναρμόνιση με ένα ευρωπαϊκό κατάλογο μετά από τις διαπραγματεύσεις όμως δεν έχει ληφθεί υπόψη αυτό ενδεχάμενο υπάρχουν εθνικοί κατάλογοι και σύμφωνα με μια κατάλληλη διαδικασία για μια κατάλληλη πλαισίωση σε αυτές τις χώρες η ροή, η προσέγγιση, τα όσα διακυβεύονται διπλωματικά κλπ. Όλα αυτά εξηγούν ε, γιατί τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να επεξεργαστούν αυτόν τον ευρωπαϊκό κατάλογο ασφαλών χωρών. Υπάρχει εθνική κατάλογη σε 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις, χωρίς μια συνοχή ανάμεσά τους πολύ συχνά, ανάλογα με τα κράτη-μέλη, μια αριθμός 1-16, μερικές φορές ακόμα και 26 κάποιες άλλες μια διαφορετική προσέγγιση της έννοιας αυτής γιατί υπάρχουν χώρες σίγουρες όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε, Αυστραλία, Καναδά και η Ιαπωνία και άλλες έχουν άλλο τις ε, χρήσιμες, τους χρήσιμους καταλόγους μόνο από εκεί που προέρχονται αυτοί που ζητούν άσυλο και υπάρχουν και διαφορετικές ε, προσεγγίσεις για αυτές τις χώρες γιατί κάποια κρατημέλη ας πούμε λένε την Κάνα ότι είναι σίγουρη, ασφαλής, ενώ άλλοι λένε είναι μόνο για τους άνδρες και όχι για τις γυναίκες, καταλαβαίνετε. Εδώ λοιπόν και το Βέλγιο που λέει ότι όχι πια η Αλβανία, ενώ το Κωσυφοπέδιο ναι, και από την άλλη μεριά οι Γάλλοι λίγες εβδομάδες πριν είχαν φτάσει σε εντελώς διαφορετική, είχαν διαφορετική προσέγγιση. Ε, δεν περιλαμβάνουν το κοσυφοπέδιο αλλά διατηρούν Αλβανία. Και μετά από νομοθετική πρόταση Επιτροπής υπάρχει ένας καταλόγος με 7 χώρες με την Αλβανία, Βοσνία, Ζεγοβίνη, πρώην ε, Δημοκρατική, Δημοκρατία Μακεδονίας, Τουρκία και μερικές παρατηρήσεις ακόμα σε τέσσερις τομείς που σίγουρα θα πρέπει να προχωρήσουμε, να προοδεύσουμε και στο μέλλον, ε, σε συνοήση με τους συναδέλφους και όλοι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό. Είχα πει ότι υπάρχει μια κάποια σύγχυση που επικρατεί σχετικά με αυτή την έννοια ασφαλής προέλευσης. Το ανακοινωθέν τύπο του Ευρωπαϊκού σήμερα έλεγε τρίτη χώρα, τρίτη χώρα σίγουρη. Αυτό έλεγε ακριβώς ενώ δεν είναι, δεν είναι έτσι. Θα πρέπει να το επεξεργαστούμε κάπως αυτά, ώστε να έχουμε ακριβώς την ίδια έννοια κατά νου. Και κάνουμε τελευταίο σχετικά πώς συνδυάζονται αυτά από εθνικής πλευράς με την ευρωπαϊκή πλευρά. Υπήρχαν διαφορές αποκλήσεις σημαντικές. Τι μπορεί κανείς να περιμένει τώρα ε, από μια εναρμόνιση μετά από πρώτης επιτροπής. Αυτή η επιρροή πώς θα είναι υψηλότερη. Τι ακριβώς θα γίνει από τη στιγμή που ένα κράτος αφαιρεθεί, διαγραφή από αυτόν τον κατάλογο ασφαλών χωρών, σίγουρων χωρών, τι θα γίνει, μπορεί να πάει στις εθνικούς καταλόγους και υπό ποιε συνθήκες, ποιε προποθέσει και ακόμα άλλε προτάσεις, δυσκολίες, δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω. Μέθοδο ε, ε, και μεθοδολογία που χρησιμοποιείται, τι θα περιληφθεί που ο νομοθέτης θα πρέπει να το ελέγχει αυτό ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλούς κράτους και η Επιτροπή θα πρέπει να μας πει με ποιο τρόπο γίνονται αυτές οι εκτιμήσεις, από ποια πηγή, θα δούμε σε λίγο μερικά παραδείγματα όπως επίσης ε, θα πρέπει να δούμε το κατάλληλο τμήμα που θα μας δώσει πληροφορίες και να δούμε και τη μεθοδολογία επαναλαμβάνω που χρησιμοποιείται και είναι κάτι, ένα εργαλείο πολύ σημαντικό να δούμε ακριβώ πώς αυτά συνδυάζονται και με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Κάτι ακόμα τελευταία που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι πώς υιοθετείται και πώς αναθεωρείται αυτός ο κατάλογο, ποιος το κάνει Πώς, με ποιο τρόπο. Ποιος είναι ο αρμόδιος οργανισμός, ο αρμόδιος φορέας για να το κάνει αυτό στην επεξεργασία είτε στην αναθεώρηση του καταλόγου. Η Επιτροπή μόνο μπορεί να το κάνει αυτό. Δηλαδή να επανεξετάζει θα προσθεθεί μια ανακράτωση ή όχι και τα κράτη-μέλη προτείνουν τροποποιήσεις. Τι γίνεται, θα πρέπει να το δούμε αυτό, θα πρέπει να απαντήσουμε για το πόσο γρήγορα θα υπάρχει μια αντίδραση σε αυτό, έτσι. Αυτά είναι από τα στοιχεία που θα ήθελα να σας πω και περιμένω τις παρατηρήσεις σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πολύ Σιλβί. Είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο που είμαστε τόσο πιεσμένοι από χρονική σκοπιά, αλλά έθεσες πολύ σωστά το πλαίσιο της πρότασης. Επομένω, δυστυχώ δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου για μια σύντομη παρέμβαση. Ευχαριστώ. Να σας δώσω και ορισμένα στοιχεία. Αν δείτε τα αριθμητικά στοιχεία για τα Δυτικά Βαλκάνια που περισσότερα μας αφορούν εδώ, ο αριθμός των ετούντων διεθνούς προστασίας αυξάνει συνεχώ από το 2008 και μετά. Και στην περίοδο Ιανουάριο με Οκτώβριο έχουμε ήδη 183.835 ετούντε από τα Δυτικά Βαλκάνια. Αν το συγκρίνετε με πέρυσι, είχαμε 109.000, σχεδόν 110. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, ότι στην περίοδο αυτή 17% όλων των ετούντων άσυλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση προήλθαν από τα Δυτικά Βαλκάνια. Αν δείτε τις κύριες χώρες προέλευσης των ετούντων άσελων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι τον Οκτώβριο τα Δυτικά Βαλκάνια ήταν στην τέταρτη θέση. Αλλά αν δείτε το 2015 συνολικά, αυτοί που έρχονται από τα Δυτικά Βαλκάνια κατατάσσονται στη δεύτερη θέση. κύριος προορισμός η Γερμανία. και στην οδό των Δυτικών Βαλκανίων είχαμε κυρίως Αλβανούς και Κωσοβάρους. Τώρα, ποσοστά αναγνώριση. Εξαιρετικά σημαντικό, γύρω στο 2% αυτή τη στιγμή από του υπηκόου χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. και όλοι τους έχουν ποσοστό αναγνώρισης κάτω από 5% αυτή τη στιγμή. Με υψηλότερο ποσοστό στους Ποσοβάρους, όπως βλέπετε. Η άλλη γραμμή είναι η περίπτωση της Τουρκίας. Γιατί θα πρέπει να εξετάζουμε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων διαφορετικά σε σχέση με τις υπόλοιπες ασφαλείς χώρες. Πρώτον, ε, το μέγεθος ε, είναι πολύ μεγάλη κλίμακα. Ε, συνεχείς επαναλαμβανόμενες αιτήσει και ε, το ποσοστό αναγνώρισης είναι πολύ χαμηλό, όπως είπα. Έχουμε οργανώσει πολλά εργαστήρια, κάνουμε και συγκριτικές μελέτες για τους παράγοντες έλεξης και απόθεσης, για τους αποθετικούς παράγοντες, για παράδειγμα, Εν γέννη δεν υπάρχει δίωξη, δεν υπάρχουν ζητήματα βλάβης, κυρίως έχουμε έλλειψη προοπτικής για το μέλλον και προβλήματα στα εθνικά συστήματα παιδείας, υγείας και το καθεξής. Αυτά τα ζητήματα οθούν από τους ανθρώπους στην Ευρώπη. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα προβληματισμού όπως τα ναρκωτικά, ε, στην Αλβανία και βία κατά των LGBT, το αναγνωρίζουμε. Τώρα για τους ε, παράγοντες έλξης, κυρίως οικονομική, δείχνουν τα στοιχεία μας, και παράγοντες που συνδέονται με το σύστημα ασύλου και τα επιδόματα που δίνονται μέσω αυτού του συστήματος. Υπάρχει η διαθεσιμότητα ιατροφαμιλικευτικής περίθαλψης και τα πακέτα επιστροφών Υπάρχουν επίσης και ταξιδιωτικά παρακτορία, αλλά και ομογένεια και η γεωγραφική εγκύτητα με την Ευρώπη είναι σημαντικοί παράγοντες. Ναι, θα προσπαθήσω να συνοψίσω. Τα κράτη-μέλη έχουν ε, λάβει μια σειρά μέτρων για να εντοπίσουν αυτέ τι ροέ. Προσπάθησαν να μειώσουν το χρόνο επεξεργασίας. έχουν μειώσει και περικόψει τα επιδόματα στο σύστημα ασύλου και έχουν κάνει και εκστρατείε πληροφόρηση ε, στα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν υπάρχει χρόνος. Ναι, όντω, λέει ο Πρόεδρο. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σιλβέστρη, παρακαλώ. the Fundamental Rights Agency, of course. Thank you very much. Πού εστάτ. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και πριν ξεκινήσω θα ήθελα να κάνω ένα γενικό σχόλιο και φυσικά και η Υπηρεσία θεμελιδών Δικαιωμάτων καλωσορίζει τι πρωτοβουλίες που απομακρύνουν τους πόρους από κάποιες ε, τέτοιες ε, σκέψεις οι οποίες ε, ε, ενδεχομένω να μην είναι τόσο αποτελεσματικέ. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σα κάποιε σκέψει σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο τη ε, πρόταση στα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ότι έχουμε κάποια σημεία τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε για να δούμε κατά πόσον ποιος, να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος ε, στα θεμελιώδη δικαιώματα. Καταρχάς να βρούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία θα μετρήσουμε. Να δούμε το περιεχόμενο των δικαιωμάτων, κατά πόσο υπάρχουν περιορισμοί και τις ε, προδιαγραφές των απαιτήσεων στο άρθρο 52.1. Σημαντικό είναι το τεστ αναλογικότητας. Τρία βήματα σε αυτό το τεστ, σε αυτή τη δοκιμή αναλογικότητας, κατά πόσο είναι κατάλληλο το μέτρο, κατά πόσο είναι απαραίτητο και κατά πόσον είναι αναλογικό υπό απόλυτους όρους. Εδώ έχουμε δύο βασικές κατηγορίες. Έχουμε τα απόλυτα δικαιώματα, όπως η μη επαναπροώθηση, η απαγόρευση της συλλογική ε, απομάκρυνσης και ύστερα κάποια δικαιώματα τα οποία περιλαμβάνουν ενδεχόμενους ε, περιορισμούς όπως ε, το δικαίωμα αποτελεσματικών έναμων μέσων, το δικαίωμα της ελευθερίας, το δικαίωμα του παιδιού. Έχω μία διαφάνεια για τα απόλυτα δικαιώματα, για την αρχή της ε, μη επαναπροώθησης, υπάρχει δυνατότητα για θέματα ασφάλειας και θα πρέπει η δικασία αυτή να αποτελεί αποτέλεσμα και προϊόν μεμονωμένης αξιολόγησης και το δικαίωμα ακρόασης του ενδιαφερομένου για, το, για τη συλλογική απομάκρυνση. Αυτό αφορά και τα σύνορα και το ανοιχτό πέλαγος. Κοιτώντας τα μη απόλυτα δικαιώματα, η βασική πρώτη αρχή είναι η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης από δύο πλευρές. Καταρχάς, άμεση διακριτική μεταχείριση βάσει της χώρας προέλευσης και κατά δεύτερον, έμεση διακριτική μεταχείριση σε περίπτωση μειονοτήτων στις χώρες που θεωρούνται ε, ασφαλείς. Αν ο συνάδελφος ε, τους ΛΟΑΔ στα Δυτικά Βαλκάνια, για παράδειγμα. Προφανώς. Ο σκοπός είναι να πετύχουμε τον νόμιμο στόχο. Αλλά τι κάνουμε. Αν θέλουμε να εξετάσουμε κατά πόσον είναι αναλογική και δικαιολογημένη η ανάμειξη με την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης. Καταρχάς, κοιτάμε κατά πόσον είναι κατάλληλο το μέτρο, κατά πόσον θα προωθήσει τις διαδικασίες που χρειάζονται σύμφωνα με τις συνθήκες κατά πόσον επίσης ε, παραμένει ο κατάλογος των ε, ασφαλών χωρών και κατά πόσον θα επιταχύνει τη διαδικασία των ε, αντικαιολόγητων των αιτήσεων. Σε ό,τι αφορά το θέμα της, το κατά πόσον είναι απαραίτητο το μέτρο, θα πρέπει να κοιτάξουμε αν υπάρχουν άλλα μέτρα ανάλογα για παράδειγμα, οι διαδοχικές αιτήσει. Ε, σε ό,τι αφορά τέλος την αρχή και την δοκιμή της αναλογικότητας. Θα ήταν σημαντικό να δείξουμε για κάθε μία από τη χώρα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο ξεχωριστά ότι το ποσοστό δικαιολογεί τη λήψη του μέτρου για να μειωθεί και ο κίνδυνος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες που διακυβεύονται, ιδιαίτερως οι εθνικές, οι εθνοτικές μειονότητες και η ΛΟΑΔΑ. Στις δύο τελευταίες τώρα διαφάνειες, αποτελεσματικά ένωμα μέσα, θα ήθελα να επισημάνω την συμπερίληψη των ετούντων και της αρχής ασφαλούς χώρας. Εδώ ενδεχομένως να δικαιολογείται η διαδικασία αναστολής και ύστερα ένα μέσα κατά του άρθρου 3 για να δούμε κατά πόσο χρειάζονται ή όχι προσαρμογές στην οδηγία για το άσυλο και για τα αποτελεσματικά ενδικά μέσα για να πληρούνται οι όροι των όσων προβλέπει το δικαστήριο. Και τέλος, να επισημάνω άλλα δύο δικαιώματα τα οποία ενδεχομένως να επηρεάζουν το δικαίωμα της ελευθερίας και τα δικαιώματα του παιδιού. Εδώ η οδηγία προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες για άτομα τα οποία ετούνται άσυλο από τρίτες χώρες προέλευσης και είναι σημαντικό να καθορίσουμε τον αντίκτυπο στα παιδιά και ιδιαίτερα στα συνόδευτα παιδιά και τους κανόνες που αφορούν τις εντάσεις και τις τριβές στα σύνορα. Κατά πόσο λοιπόν προαπαιτούνται προσαρμογές. Και στην τελευταία διαφάνεια έχουμε κάποιες συστάσεις και θεωρώ ότι από πλευρά της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αυτό που είναι σημαντικό είναι να γίνεται συνεκτικά η αξιολόγηση και να υπάρχει διαφάνεια σε αυτή την αξιολόγηση και να διατίθεται και σε άλλους στο μέλλον. Τρίτον, να υπάρχει μεμονωμένη αιτιολόγηση για κάθε μία από τις τρίτες χώρες και τέλος να αναλογιστούμε τρόπους με τους οποίους ε, ενδεχομένω να υπάρχει έμεσο αντίκτυπο σε κάποιε εθνοτικέ και σεξουαλικέ μειονότητε χωρών που θεωρούνται ασφαλεί. Και μήπω να εξετάσουμε το ενδεχόμενο λήψη μέτρων για να μειωθεί αυτό ο αντίκτυπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Σα ευχαριστούμε και του δύο για το γεγονό ότι ήσασταν πολύ σύντομοι. Συνάδελφοι, έχουμε τέσσερα λεπτά Ξέρω ότι κάποιοι βουλευτές περίμεναν με υπομονή το τέλος της συζήτησης. Ε, προφανώς ε, θα πρέπει να είσαστε πολύ σύντομοι, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε ερμηνεία. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Ντάτη. Αλλά αν θέλετε σύντομοι. Αν δεν θέλετε να μιλήσετε, σε ένα λεπτό πάντως, σε ένα λεπτό. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας, η κυρία Ντάτη Ντεπρέ Άντερσεν. Έχετε το λόγο, κύριε Ντάτη. Euh, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μετά από αυτό το δράμα στα Παρίσι και την τρομοκρατική επιλή δεν θα πρέπει να κάνουμε να ξεχνάμε και το άλλο με το οποίο ασχολούμαστε εδώ, δηλαδή την προσφυγική ροή. Θα ήθελα να μπορέσουμε να έχουμε μια ήρεμη συζήτηση, γαλήνια συζήτηση, ώστε να μην μπερδεύουμε τα δύο, μια σύγχυση δηλαδή, ώστε να μην έχουμε αυτόν τον κατάλογο των ασφαλών χωρών. Εδώ λοιπόν χρειάζεται ένας κοινό κατάλογος ε, από όλους. Βέβαια θα πρέπει να δούμε αυτές τις προτάσεις που δεν προκαλούν όμως ένα πρόβλημα αυτό που είναι το πρόβλημα τα κριτήρια για αυτή την επιλογή. Και μια χώρα είναι η Τουρκία ας πούμε, εκεί γίνεται πολλές συζητήσεις θα πρέπει να δούμε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για Δικαιώματα Ασύλου, θα δούμε πώς θα μπορέσει να μας βοηθήσει για την επεξεργασία αυτού, τη σύνταξη αυτού του καταλόγου και είναι πολύ σημαντική αυτή η εργασία και θα πρέπει να, να δούμε και το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις εργασίες μας. Ευχαριστώ. Κύριε Διπρέ, έχει το λόγο. Ναι, γρήγορα, γρήγορα, τάχιστα κύριε Πρόεδρε. Για αυτό τον κατάλογο τρία προβλήματα υπάρχουν. Θα πρέπει να υπάρξει λύση. Την όλη διαδικασία πώς μπαίνει κανείς, πώς βγαίνει κανείς δεν είναι και τόσο εύκολο χωρίς πόνο και πώς θα συμπίπτουν ο ευρωπαϊκός κατάλογο με τον εθνικό. Σημαντικά είναι ένα σύστημα μόνο και αυτή η σημερινή πρόταση της Επιτροπής για την Τουρκία να συμπεριληφθεί στον κατάλογο Κάτι όμως που δημιουργεί κάποιες αντιδρασούλες από μας ε, και αμφιβολίες. Ε, τη στιγμή που υπάρχει ε, η χώρα σε αυτόν τον κατάλογο, τι θα γίνει, θα μπορούσε να επιτάξει μια επιτάχυνση διαδικασίας. Αλλά η επιτάχυνση διαδικασίας τι σημαίνει με τη σειρά της. Κάπως αναταραχές στον σημερινό μηχανισμό σχετικά κυρίως, κυρίως, κυρίως με το πόσο θα διαρκέσουν αυτά ε, αυτά είχα να πω. Τέλειωσα, τέλειωσα. Και εντάξει, σίγουρα θα προσέξουμε ιδιαίτερα αυτά που ο Οργανισμός για τα θέματα Δικαιώματα έθεσε τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Άντρασα Μαρτίνα για την ΓΟΕ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Με απασχολεί και με προβληματίζει ιδιαίτερω ε, η μέθοδο και η μέθοδοι, μάλλον ευρύτερα, αξιολόγηση που χρησιμοποιούνται. Ακούσαμε και κάποια σχόλια σε σχέση με την Τουρκία πιο συγκεκριμένα. Αν δείτε τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να δούμε αν κάποια χώρα περιέχεται ε, στον κατάλογο των ασφαλών χωρών μιλούμε για ε, χώρες που δεν υπάρχει ε, ένοπλη σύραξη και σύγκρουση λοιπά μας ακούσαμε τις τελευταίες εβδομάδες ότι η Τουρκία βρίσκεται εν μέσω ειρηνευτικής διαδικασίας. Δεν κατανοώ λοιπόν πώς μια τέτοια χώρα μπορεί να μας παρουσιάζεται ως ασφαλής. Βάσει παρατηρήσεων που έχουν γίνει και τα όσων συμβαίνουν με τους Κούρδους. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Μαρτίνα. Η κυρία Βαλέρο για τους πράσινους, αντικαθιστά τον ε, κύριο Λαμπέρτ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, εμείς θεωρούμε ότι η Τουρκία δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτόν τον κατάλογο ε, επειδή τα είπαμε αυτά τα πράγματα. Είναι μια special κατάσταση όμως ειδική. Έχουμε 25% μας έρχονται μέσω της Τουρκίας. Υπάρχουν και πολιτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται. Τι γίνεται, θα πρέπει να κάνουμε μια εκτίμηση αντικειμενικά στις χώρες. Δεν είναι μόνο τα πολιτικά κριτήρια. Και επίσης για την επικουρικότητα. Εδώ αναφερθήκαμε σε ασφαλείς χώρες που τα λένε, λένε ποια είναι τα κρατημέλη ακριβώς. Εδώ θα πρέπει να δούμε παρόμοια ερμηνεία είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό. Τι γίνεται ακριβώς, ποιες είναι ερμηνείες που θα λυθούν υπόψη, διαφέρουν, ποικίλουν και όταν εξετάζουμε και διάφορες περιοχές μιας χώρας και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σημαντικό το σημερινό θέμα γιατί θα πρέπει να αναχωρήσουν όσοι δεν είναι νόμιμοι. Το σύστημά μας ε, ε, δεν είναι αποτελεσματικό, μόνο το 40% και είναι 300.000 άτομα το χρόνο. Επιβάλλεται να υπάρξει αυτός ο κατάλογος των ασφαλών χωρών και το πρώτο, από την πρώτη σύνταξη έχουμε μόνο 7 υπάρχουν ε, χώρες των Βαλκανίων και η Τουρκία. Είναι δύο πηγές όμως μαζί μας έρχονται ε, πρόσφυγες και τι γίνεται, πώς μπορούν να είναι σε αυτόν τον κατάλογο, γιατί 7 Νομίζω ότι βασιζόμαστε σε εθνικούς καταλόγους, λέει 16 ο γαλλικός κατάλογος ή το με βασίλειο 26. Στο γαλλικό κατάλογο έχουμε την Ινδία, τη Ενεγάλης σίγουρες χώρες που θα μπορούσαν να προσθεθούν. Γιατί εμείς μόνο 7 έχουμε προς το παρόν. Θα πρέπει να το συλλογιστούμε. Και ένα τελευταίο πρόβλημα πώς οι εθνικοί κατάλογοι θα συνεπάρξουν με τον ευρωπαϊκό κατάλογο. Υπάρχουν 12, ευρωπαϊκοί, 12 ε, εθνικοί κατάλογοι. Η κυριαρχία κάθε καθοσμένος νομίζω ε, θα, θα πρέπει να γίνει σεβαστή και να δούμε πώς θα μπορέσουν να συνεπάρξουν αυτοί οι δύο κατάλογοι, ο εθνικός με τον ευρωπαϊκό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος προς ε, του Τερμινής. Ε, τελευταία, η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ, πρόεδρε, εν συντομία. Ακούσαμε πολλά για τα κριτήρια για να εξαπρεθεί ένας ορισμός για το κατά πόσον είναι ασφαλής χώρα προέλευσης ε, η χώρα ή όχι. Για τους πολίτες της δηλαδή ασφαλής. Αλλά κοιτώντας τους εθνικούς καταλόγους, τις εθνικές λίστες, φαίνεται ότι πέρα από τα κριτήρια αυτά υπάρχουν και προφανώς και κάποιες πολιτικές ηλεμένες αποφάσεις για το κατά πόσον θα υπάρξουν ε, Λίστε και ποιε χώρε θα περιλαμβάνουν. Αυτό εξαρτάται λοιπόν και από πολιτικέ αποφάσει, κοιτώντα λοιπόν τις ε, λίστε στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω την εντύπωση ότι και πάλι κρύβεται πίσω από αυτό μία πολιτική απόφαση. Και κάποιο το είπε, είναι δύο χώρε χώρες ε, από τι οποίε προέρχονται πολλοί πρόσφυγε. Ελπίζω να μην είναι αυτός ο λόγος που έχουν μπει στη λίστα. Να προσέξουμε για να μην μπουν σε ένα κουτί σε μια ομάδα διάφορες χώρες και να τις εξισώσουμε. Μιλάμε επίσης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Λες και είναι ίδιοι οι όροι και οι συνθήκες σε όλες τις χώρες στα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν αληθεύει αυτό. Να δούμε τι αποφασίζουμε λοιπόν, να προσέξουμε. Μία πρόταση να πάω προς τον κύριο Γιούγκερ. Είπε ότι όλες αυτές οι χώρες χωρίς καμία αμφιβολία είναι ασφαλείς χώρες προέλευσης γιατί είναι υποψήφιες χώρες για προσχώρηση και ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λυπάμαι, είναι υποψήφιες. Αυτό δεν σημαίνει ότι πληρούν όλα τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Αν τα πληρούσαν τα κριτήρια της Κοπενχάγης, όπως ε, διατείνεται ο κ. Γιούγκερ, θα μπορούσαν ήδη αύριο να ενταχθούν στην Ένωση. Ως εκ τούτου, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί είναι υποψήφιες χώρες επειδή δεν πληρούν τα κριτήρια ακόμα. Πολύ προσεκτικοί να είμαστε με όλες τις χώρες στη λίστα. Και για να λεφτεί μια γρήγορη απόφαση για το κατά πόσο θα μπει κάποιος στη χώρα μας ή όχι. Αυτό μπορεί να γίνει και χωρίς τη λίστα των χωρών ασφαλούς προέλευσης, αν υπάρχουν οι τεχνικές, επαρκείς υπάλληλοι, για να αποφανθούν για το άσυλο, για τις αιτήσει άσυλο. Και ήδη αυτό γίνεται σήμερα. Είναι εφικτό, χωρίς ε, κίνδυνο. Ευχαριστώ η Σιλβή και πάλι για να κάνει κρατικά σχόλια. Ναι. Ναι, πολύ σύντομα γιατί βλέπουμε τις ευρύτερες ε, τάσεις ε, που σχεδιαγραφούνται, αλλά και τα κριτήρια και τον τρόπο που βλέπουμε εξετάζουμε τη συνύπαρξη των δύο καταλόγων. Χρειαζόμαστε λοιπόν επιπλέον πραγματογνωμοσύνη που δεν θα καθυστερήσει τη λήψη αποφάσεων αλλά θα μα βοηθήσει στην διαδικασία αυτή. Ευχαριστούμε πολύ, Σιλβί. Ευχαριστούμε και του συναδέλφου για την υπομονή του. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Θα το βάλουμε πιο ψηλά το θέμα σας την επόμενη φορά στην ημερήσια διάταξη. 7 Δεκεμβρίου η επόμενη συνεδρίαση.